Right, welcome everybody. We've now got, uh, I think... Καλώς ήρθατε όλοι, εκπροσωπούνται λίγο πολύ όλες οι ομάδες. Πολύ καλό αυτό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να ρυθμιστούν τα ταξίδια τη Δευτέρα, παρόλο που είδα ότι οι Βέλγοι τα κατάφεραν να έρθουν εδώ, τα κατάφεραν και τα καλά. Τέσσερι. <laughs> Yes. Ε, εγκρίνεται η μέρη σε διάταξη. Ωραία. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Φοβούμαι ότι έχουμε ανακοινώσει Προέδρου. Πρώτα απ' όλα να σα υπενθυμίσω ότι αύριο δεν είμαστε με την αίθουσα, αλλά στη Μικύκλιο. Οπότε πάρτε μαζί σας τα χαρτιά σας παρακαλώ να μην χαθούν διαφορετικά στη μεταφορά. Να σας ενημερώσω για τους τριμερείς διαλόγους που συνεχίζονται. Παράξενο θέμα αυτό όσον αφορά τα, ευρωπαϊκά επενδυτικά κεφάλαια, κεφάλαια κινδύνου και τα ταμεία τα, για τις επιχειρήσεις. Είχαμε και για τα δύο θέματα ξεχωριστούς τριμερείς διαλόγους στις 12 Ιουνίου και έγινε πρόοδος ε, επί διαφόρων θεμάτων και επόμενος τριμερείς διάλογος έχει σχεδιαστεί για τις 20 Ιουνίου. Για το CRD4 CRR, δύο τριμερείς διάλογοι, 13 και 14 Ιουνίου, έγινε καλή πρόοδος ολοκληρώνοντας τις συμβιβαστικές για τα για τα κεφαλουχικές απαιτήσει με κάποια, κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες θα πρέπει να διευθυνθούν αυτή την εβδομάδα. Υπάρχουν όμως ε, μεγάλα θέματα που εκκρεμούν όπως οι αμοιβέ, σχέδια για την επίλυση προβλημάτων τραπεζών και για συστηματικούς θεσμικά όργανα το κεφάλαιο που θα χρησιμοποιείται σαν απόθεμα, σαν προστατευτικό στρώμα και αυτό το θέμα των προστατευτικών στρωμάτων uh, buffers ε, συμπεριλαμβάνεται και στον κανονισμό οπότε όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε μαζί και την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν και άλλοι τριμερείς ε, διάλογοι για το θέμα των ε, στεγαστικών δανείων και στη οδηγία πέρα από την ψηφοφορία της περασμένης εβδομάδας ο εισηγητής απουσιάζει δεν θα μιλήσουμε για την υπόθηκα δάνεια τώρα αλλά αργότερα όταν εμφανιστεί ο εισηγητής είμαι στη σελίδα 2 υπάρχει κάποια διόρθωση στο ΕΜΕΑ, ΕΜΙΡ, όλες οι γλωσσικές διορθώσεις μετά από αναθεώρηση από τους νομοθήσεις γλωσσικούς διενεμήθησαν στα μέλη της ΕΚΟΝ στις 14 Ιουνίου ε, σύμφωνα με το άρθρο 216 του εσωτερικού κανονισμού εν τη απουσία ιονδήποτε αντιρρήσεων πλευράς Επιτροπής τα διορθωτικά, το διορθωτικό κείμενο θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και θα ανακοινωθεί στην σύνοδο του Ιουλίου στο Στασβούργο και θα θεωρηθούν εγκεκριμένα εκτός αν κάποια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 μέλη ζητήσουν το διορθωτικό να ψηφιστεί. Χρειάζεται να διαβάσω το περιεχόμενο. Εν συντομία, αφε μου, διαβάσω το περιεχόμενο, μου λένε. Άρθρο 14 και 85, στο άρθρο 14, σημείο 5, δεύτερη υποπαράγραφος, προβλέπει ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2014, νομίζω διόρθωση αφορά τον μήνα, θα υπάρξει σχέδιο εκθέσεως για τις συνέπειες της ε, εφαρμογής πρόσθετων απαιτήσεων πλευράς κρατών μελών και στο άρθρο 85.3 προβλέπεται ότι η ΕΣΜΑ θα υποβάλει μέχρι τις 30 του Σεπτεμβρίου έκθεση του 2014. Οπότε το διορθωτικό διαγράφει τη δεύτερη παράγραφο της 14.5 και τροποποιεί τη διατύπωση ούτως ώστε να συμπίπτει, να ταιριάζει και χρησιμοποιεί τη διατύπωση του 14.5. Όλα συμβαίνουν το Δεκέμβριο δηλαδή με άλλα λόγια. Και μετά στο άρθρο 89 υπάρχει μια αλλαγή που εξασφαλίζει την προθεσμία όπου είτε τα κεντρικά τη συμβαλόμενα μέρη και οι διάφοροι εμπορικοί φορεί πρέπει να συμμορφωθούν με τον κανονισμό είναι σαφή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να θετήσει ή τη μορφή τεχνικές υπό τη μορφή κατεξιστότηση πράξεων είναι μόνο η ημερομηνία θέση ισχύ και όχι η ημερομηνία που έθετη τα πρότυπα και δημοσιοποιούνται από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι μια τεχνική φύσεω διευκρίνηση. Στου επόμενου 200 τριμερεί διαλόγου θα διορθώσουμε αυτά. Και τώρα μπορούμε να πάμε στο σημείο 3, αφορά τον οικονομικό διάλογο με το Βέλγιο και ανταλλαγή απόψεων με τον Στίβεν Βανάκερεμ, τον Υφυπουργό και Υπουργό Οικονομικών και Βιώσιμη Ανάπτυξη, τον Αντιπρόεδρο τη Κυβερνήσεω λοιπόν και Υπουργό Οικονομικών και Εφόρου Ανάπτυξη, που είναι φετισμένο με δημόσια διοίκηση, θα αφήσουμε πρώτα τον κύριο Υπουργό να μα μιλήσει και μετά θα ανταλλάξουμε απόψει. Λυπούμε έπρεπε να περιμένετε για τι ανακοινώσει Προέδρου, αλλά βλέπετε ένα κοινοβουλευτικό καθήκον που είμαι σίγουρο, σίγουροι μάλλον ότι γνωρίζετε. Μην ανησυχείτε κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρίε και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με μεγάλη χαρά βεβαίω δέχτην την πρόσκλησή σα. Ω ε, νέο ε, Υπουργό Οικονομικών του Βελγίου, ε, θέλω να δεσμευτώ περισσότερο σε ένα διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ό,τι με αφορά είναι τιμή μου αυτό να μπορώ να το κάνω με την Επιτροπή σας, τη μόνιμη Επιτροπή για Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις. Το 2011 η Βελγική Προεδρία υποστήριξε πλήρως και δέχτηκε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και το ευρωπαϊκό όραμα της χώρας μου είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό και δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι το Βέλγιο και γνωρίζετε είναι πολύ προσιλωμένο στο Κοινοβούλιο το οποίο και θέλω να ε, εξάρω για την προσήλωσή του στις ευρωπαϊκές αξίες και ιδέες. Είμαι στη διάθεσή σας για να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος στον οικονομικό διάλογο. Κυρίες και κύριοι, δεδομένου των συνθήκων, νομίζω είναι σωστό να πούμε ότι η οικονομική κατάσταση στο Βέλγιο ε, υπήρξε καλύτερη από ό,τι στην Ευρωζώνη γενικότερα. Η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου υπολόγισε πρόσφατα ότι από την αρχή της κρίσης το ΑΕΠ του Βελγίου ήταν το πιο κρατεό σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Δυστυχώς Δεν αρκεί αυτό για να δηλώσουμε ικανοποίηση. Αν δείτε όμως την πρώτη διαφάνεια θα καταλάβετε ότι την τελευταία τετραετία η μεγέθυνση της οικονομίας στο Βέλγιο ε, ήταν αρκετά σφριγγυλή και ε, κρατεά. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους. Πρώτον, το Βέλγιο έχει πολύ ισχυρά οικονομικά ε, θεμέλια. Αν δείτε τη δεύτερη διαφάνεια θα δείτε ότι οι Βέλγοι έχουν το μεγαλύτερο ενεργητικό κατακεφαλήν την Ένωση και 200% του ΑΕΠ. Είναι διπλάσιο από το χρέος. Το χρέος, το δημόσιο χρέος είναι πολύ υψηλό, αλλά ε, υπερκαλύπτεται από την ιδιωτική ε, αποταμίευση και περιουσία των Βέλγων πολιτών. Στη συνέχεια, θα ήθελα να σας πω ότι η προσέγγιση του Βελγίου ε, στην κρίση και την καταπολέμησή της ήταν ε, πραγματικά ε, πολύ εύστοχη πιστεύω. Αντιμετωπίστηκαν πολύ γρήγορα τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα ε, και με, έχοντας στο μυαλό του το κράτος της καταθέσης των πολιτών και της περιουσίας του και του ιδίου και πολύ σύντομα συγκρατήθηκε. Αντιμετωπίστηκε επίσης το θέμα της ανεργίας ε, και της παραγωγικότητας. Αν περάσετε στην επόμενη διαφάνεια θα διαπιστώσετε ότι σήμερα η ανεργία είναι χαμηλότερη από την περίοδο πριν ξεσπάσει η κρίση. Οι οικονομικοί σταθεροποιητές και τα ε, μέτρα προσωρινής ανεργίας μας βοήθησαν έτσι ώστε ε, η ανεργία να έχει θετικά αποτελέσματα τουλάχιστον σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Ε, και ένα τελευταίο σχόλιο σε ό,τι αφορά πάντα το βέλιο και τη στρατηγική του για την καταπολέμηση της κρίσης είναι ότι σε τελική ανάλυση είχαμε μια στρατηγική έξυπνη για τα δημόσια οικονομικά. Ε, το πρόγραμμα ανάκαμψης της οικονομίας που προώθησε ε, το ε, κράτος ε, ήταν περιορισμένο και δεν εξεράγησαν ποτέ τα ελλείμματα. Από τον Οκτώβριο του 2009 και μετά το Βέλγιο άρχισε με τη διαδικασία εξυγίανσης του προπολογισμού 2010-2011 και νομίζω ότι αυτή η στρατηγική για τα δημόσια οικονομικά που τη χαρακτηρίζω αρκετά ευφυή μεταφράστηκε σε μια συνεχώς μειούμενη διαφορά του λόγου του βελγικού χρέους σε σχέση με το μέσο όρο στην Ευρώπη. Θα δείτε και πάλι στη διαφάνεια ότι η διαφορά μεταξύ ε, του λόγου του χρέους ε, στην Ευρωζώνη είναι 6,5%. Ε, ξέρω ότι είναι περιορισμένο αυτό το επιχείρημα, είναι λίγο το επιχείρημα του ασθενούς που έχει πυρετό 39 και λέει εντάξει αλλά ο διπλανός μου έχει 40 πυρετό, καλά τα πάω. Είναι ένα επιχείρημα που θα πρέπει να χρησιμοποιείται με φιδό. Αλλά αν κοιτάξετε και τι έγινε στη δεκαετία του 90, που είχαμε διαφορά στο λόγο του χρέους με την Ευρωζώνη περίπου 70% ε, είναι σαφές ότι η στρατηγική της τελευταίας δεκαετίας μας έφερε πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μεσοόρο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ε, θα πρέπει να βαθίζουμε προς τη λογική του 60%. Η πρόσφατη οικονομική κατάσταση στο Βέλγιο μας φέρνει μεταξύ ε, των καλυτέρων για να το χαρακτηρίσω έτσι στις επιδόσεις. Θα πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι το Βέλγιο δεν έχει ε, αποφύγει την προσοχή των χρηματαγορών και τις ε, ανησυχίες ε, που επικράτησαν για τους εξής τρεις λόγους. Το χρέος 98% είναι η πέμπτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να είναι θετικές οι εξελίξεις, αλλά παραμένει πολύ ψηλό το χρέος. Το δεύτερο, έκθεση στον χρηματοοικονομικό τομέα. Τον Οκτώβριο το 2011 το Βέλγιο και η Γαλλία χρειάστηκε να επέμβει ε, στην ε, διάσπαση της τράπεζας Δέξια ε, για να εξηγιαθεί και να σωθεί το υγιές τμήμα. Και βεβαίως υπήρχε και ένα ζήτημα γιατί δεν είχαμε κυβέρνηση. Από τις εκλογές του Ινίου 2010 και μετά η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ήταν υπηρεσιακή και μπορεί να είχε την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και τη δυνατότητα να κάνει ό,τι χρειαζόταν για να διαφυλαχθούν τα οικονομικά συμφέροντα του Βελγίου. Οι αγορές καταλαβαίνετε ότι δεν καθησυχάζονται πλήρως ούτε και μετά από μια επιτυχή ε, Ευρωπαϊκή Προεδρία αφού δείξαμε ότι μια υπηρεσιακή κυβέρνηση μπορούσε να σεβαστεί τι διεθνείς τη υποχρεώσεις υποχρεώσεις. Παρόλα αυτά υπήρχε κάποια αναταραχή στις αγορές. Το Νοέμβριο του 2011 όλα αυτά έφτασαν στο αποκορύφωμά τους και ο Επίτροπος Ρεν μας ε, είπε ότι θα επιβάλλει το six pack από την πρώτη μέρα. Η Standard Poor's ε, μας υποβίβασε κατά ένα βαθμό και ε, έφτασαν τα σπρέτς στο 6%, τα επιτόκια συγγνώμη, στο 6%. Στις 6 ε, Δεκεμβρίου του 2011 απαντήσαμε μια στρατηγική που βασίζεται σε τρεις πυλώνες, ε, μεταρρύθμιση του κράτους, διαστατική μεταρρύθμιση και πολιετές δημοσιονομικό σχέδιο. Μεταρρύθμιση του κράτους. Οι περιφέρειες έχουν τώρα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τα ιδιαίτερα προβλήματά τους με καλύτερο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίσουν οικονομική ανάπτυξη. Είμαι πεπισμένος ότι η μεταρρύθμιση του κράτους θα είναι προς όφελος και της Ομοσπονδίας και των περιφερειών αλλά ε, κυριότερα για τους πολίτες. Τρία είναι τα στοιχεία. Πρώτον, να ξεφορτωθούμε το μήλο της έριδας στη βελγική πολιτική, ε, την περίφημη εκλογική περιφέρεια ε, BHV, ε, Βρυξέλλες, Χάλεβιλ, Βόρτε, που το γνωρίζουν όλοι. Ήταν πολύ σημαντικό να λυθεί αυτό το θέμα, έτσι ώστε στο μέλλον να μην χρειαζόμαστε 500 μέρες για να αποκτήσουμε κανονική κυβέρνηση. Στη συνέχεια, μεταφορά εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ό,τι αφορά τα εργασιακά να προσαρστούν καλύτερα στις περιφέρειες και τις ιδιαιτερότητες τους. Και το τρίτο, ε, ο περιφερειακός ε, νόμος ε, για την οικονομία με περισσότερη φορολογική αυτονομία. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαρθωτική μεταρρυθμίση, στόχος είναι να αυξηθεί η απασχόληση που είναι χαμηλή η ευρωπαϊκή προοπτική, να αυξηθεί να παραταθεί κατά δύο έτη η ηλικία συνταξιοδότησης και να μην είναι ελκυστική η πρόορη συνταξιοδότηση ή η θελουσία έξοδος και επίση οι άνεργοι ε, θα πρέπει να έχουν περισσότερα κίνητρα και περισσότερες ε, ε, αιτίε για να ενταχθούν στην αγορά εργασία με προοδευτικά μειούμενο επίδομα ανεργίας. Το πολιετές επίσης δημοσιονομικό πλαίσιο βασίζεται στη μεταρρύθμιση του κράτους και στόχο έχει να μειωθεί ε, το έλλειμμα σε 2,8%. Το 11 μειώθηκε κατά 3,7 όχι κατά 4,2 όπως αναφέρει το έγγραφο που σας έχει διανεμηθεί. Είμαστε στο 3,7 το 2011, 2,8 ε, φέτος και ο προπολογισμός θα είναι ισοσκελισμένος το 2015. Τα μέτρα ε, είναι ε, εμπροστοβαρή όπως λέγεται ε, και πάνω από 3% του ΑΕΠ αντιστοιχεί σε αυτά τα μέτρα. Το πακέτο επίση βασίζεται στις συστάσεις διεθνών οργανισμών. Το 2014, 53% των προσπαθειών εξυγίαση θα αφορούν τις δαπάνες αυξάνεται η φορολογική βάση και ε, η φορολόγηση του κεφαλαίου και ε, του περιβάλλοντος. Δεν αυξήσαμε λοιπόν ε, το ΦΠΑ ούτε τη φορολόγηση της εργασίας για να μην εμποδίσουμε την αγορά εργασίας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί ότι είναι σημαντικές οι μεταρρυθμίσεις και σημαντικά τα βήματα προς την ορθή κατεύθυνση. Και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Βέλγιο εν μέρει έχει εφαρμόσει πέντε από τις έξι συστάσεις. Βεβαίως, ε, η αντίδραση των αγορών είναι περισσότερο ποσοτική. Τα επιτόκια έπεσαν κατά 2,5% και πλέον τις 100% από 5,8% σε 3,2% την περασμένη εβδομάδα. Το spread με τη Γερμανία μειώθηκε στο μισό και παραπάνω από 366% ε, στα 174%. Ε, δεν χρειάζεται να σας πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ θετικό ως είδηση για τον προπολογισμό μας. Αλλά βεβαίως είναι πολύ νωρίς για να θριαμβολογούμε. Βράχει πρόθεσμα, η προσοχή μας θα δοθεί στην ενίσχυση ε, των προσπαθειών για να φτάσει το έλλειμμα στο 2,8 το 2012. Η κυβέρνηση είναι 100% δεσμευμένη προς το στόχο αυτό. Σε στενή συνεργασία με τον Όλη Ρεν και τις υπηρεσίες του παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο η κυβέρνηση έλαβε επιπλέον ε, δημοσιονομικά μέτρα για να φτάσουμε στους στόχους μας παρά τη μείωση της μεγέθυνσης της οικονομίας. Τον Ιούλιο προβλέπεται νέος δημοσιονομικός έλεγχος και στα πλαίσια αυτά η αρινή πρόβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου ήταν καλή ειδήσει. Η Κεντρική Τράπεζα ε, ύφξησε την πρόβλεψη ανάπτυξης από 1,1% το ΕΠ συν 0,6% το ΕΠ για το 12 και επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση ε, θα καλύψει το στόχο της. Βεβαίως, πιο μακροπρόθεσμα, αυτό μας ενδιαφέρει και είναι σημαντικό. σε ό,τι αφορά τη διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών, το Βέλγιο θα πρέπει να ε, βελτιώσει την εξωτερική του ανταγωνιστικότητα και να μειώσει το δημόσιο χρέος. Δύο προτεραιότητες, δημόσιο χρέος και ε, ε, εξωτερική ανταγωνιστικότητα χρειάζονται μόνιμες προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα πολιτικής. Η εξωτερική ανταγωνιστικότητα και η μείωση του δημοσίου χρέους είναι και ευρωπαϊκά προβλήματα και η ε, ευρωπαϊκή θεσμοί και τα θεσμικά όργανα είναι μέρος της λύσης. Σε βελγικό επίπεδο η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη να επενδύσει περαιτέρω στρατηγική 2020 για να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις αυτές. Ποια είναι τα διδάγματα τώρα για να συμπεράνουμε από την περίπτωση του Βελγίου σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Πρώτον, η δέσμη έξι νομοθετημάτων, το six-pack, οδήγησε στη χώρα μου σε πιο στενή παρακολούθηση των στόχων του προπολογισμού και είναι ε, σωστό αυτό και θετικό. Σε μια ε, νομισματική ένωση η εξέλιξη κάθε κράτους συνδέεται στενά με μια άλλη χώρα. Αν είναι σε ανισορροπία τα οικονομικά μιας χώρας ε, πλήττεται όλη η νομισματική ένωση. Το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Ε, ίσως καλύτερα από κάποιους άλλους. Γι' αυτό υποστήριξαμε και το ΣΥΚΣΠΑΚ και όλη την ιδέα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτούς τους νέους κανόνες δεν τους θεωρώ υποχρέωση, μάλλον κίνητρο και ενθάρρυνση. Το δεύτερο δίδαγμα, πιο ειδικό, λειτουργεί πλήρως ε, η αντίστροφη διπλή ε, ενισχυμένη πλειοψηφία. Τώρα βλέπουμε ότι είναι βελτίωση ε, σε σχέση με περιόδους που το Συμβούλιο μπορούσε να αλλάξει τους κανόνες κατά τη διάρκεια της πορείας. Είναι καλό αυτό και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης ε, λειτουργεί προληπτικά για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης γιατί τα κράτη-μέλη ακόμα περισσότερο έχουν κάθε συμφέρον να ε, προλάβουν τις εξελίξεις γιατί οι κυρώσεις είναι όλο και πιο αναπόφευκτες. Τρίτο δίδαγμα από τη βελγική εμπειρία είναι το εξής. Πιστεύω ότι οι γερές οικονομικές βάσεις, ε, ε, η μείωση του χρέους και ε, τα υγιή δημόσια οικονομικά όπως και στρατηγική που βοήθησαν το Βέλγιο να βγει σχετικά αλόβητο από την κρίση δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να έχει κανείς μακροπρόθεσμο όραμα και κανόνες σε ό,τι αφορά το υπερβολικό έλλειμμα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω εδώ λέγοντας ότι η Ευρώπη δεν έχει βγει ακόμα από την κρίση που την έχει συγκλονίσει η θέμελα από το 2008, αλλά η άλλη ε, όψη του νομίσματος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουδέποτε προχώρησε τόσο πολύ. Είναι ε, εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Six pack, ε, ε αντιπυρική προστασία, το δημοσιονομικό σύμφωνο. Και όπως λέει ο Φαν η Ευρώπη προχωράει μέσα από κρίσεις. Την περασμένη Πέμπτη, ενέκρινε το Κοινοβούλιο μας την αλλαγή της συνθήκης για τον ε, μηχανισμό σταθερότητας. Ε, στην Ολομέλεια... Εγώ παρέθεσα το Ζαν Μονέ που είπε ότι οι άνθρωποι δέχονται ε, την αλλαγή μόνο σε περίπτωση ανάγκης και την ανάγκη τη βλέπουν μόνο σε περίοδους κρίσης. Αυτό είναι γεγονός και έτσι προχωρεί η Ευρώπη μέσα από κρίσεις και η χώρα μας καλωσορίζει όλες τις ιδέες που είναι τώρα επιτάπητος και ε, θα συζητηθούν στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ενίσχυση της ε, Οικονομικής ε, και Νομισματικής Ένωσης, δημιουργία Τραπεζικής Ένωσης και πρόοδο προς μια πιο πολιτική ένωση. Είμαι πεπισμένος ότι η μόνη απάντηση είναι περισσότερη Ευρώπη γιατί οι μοίρε μας είναι δεμένες ελέγχετες πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. με την πεποίθηση αυτή ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις ερωτήσεις, να απαντήσω και να έχουμε ανταλλαγή απόψε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ναι, φρόντιζα το σημαντικό θέμα του καφέ. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Σας υπενθυμίζω ότι η ανταλλαγή αυτή απόψεων είναι τμήμα του οικονομικού διαλόγου που καθόρισε η Επιτροπή μας ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου επιμέναμε πολύ κατά τις διαπραγματεύσεις της εξαμέτρου γιατί είναι σημαντικό το θέμα της διαφάνειας και του εκδημοκρατισμού για να το πω έτσι της οικονομικής διακυβέρνησης governance και τώρα οι ομιλητές και ομιλήτριες από τις ομάδες όπως δήλωσαν. Αρχίζω με τους σοσιαλιστές και σοσιαλίστριες. Σαΐντ Χατράου, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης για την εισαγωγή του και σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι ήρθατε και θέλετε να συζητήσετε μαζί μας. Είναι πολύ χρήσιμο και διδακτικό για μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι και παίρνω ως προσανατολισμό τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξεδόθησαν πρόσφατα. Μια διαπίστωση πρώτα. Διαβάζω τις συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προς το Βέλγιο και επανέρχονται ξανά και ξανά μερικά πράγματα, αλλά φαίνεται ότι έχουν χαμηλώσει λίγο τους τόνους, είναι λίγο πιο πολλές οι αποχρώσεις. Συμφωνείτε εσείς με αυτό, ότι έχει μαλακώσει λίγο το είδος των συστάσεων. Και είναι σε καλύτερη μοίρα το Βέλγιο. Το είπατε κι εσείς βέβαια. Αναγνωρίζω αυτό που λέτε για την κριτική που έχει ακουστεί, για τις συστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίω εμένει στην τήρηση των στόχων, αλλά και προσπαθεί επιγόντω να εξηγήσει πώ θα φτάσουμε στου στόχου που έχουμε συμφωνήσει από κοινού. Και σα παραπέμπω λίγο ε, στη συζήτηση για την αυτόματη τη προσαρμογή ε, του Βελγίου, το ίντεξ όπως λέγεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το τονίζει αυτό για μας, όμως και για άλλους η αγοραστική δύναμη είναι πάρα πολύ σημαντική και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μιας χώρας με την καταπολέμηση του πληθωρισμού από τη συγκράτηση των τιμών, έτσι δεν είναι. Ε, δηλαδή, ιδιαίτερα σκέφτομαι εδώ τις τιμές της ενέργειας ή αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα και με άλλο τρόπο, όπως ε, με την καινοτομία, με τη διαβίου μάθηση και τέτοια πράγματα. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής τώρα, κατά την άποψή σας, πόση ευελιξία θα μπορεί να διατηρεί μια χώρα μέλος Δηλαδή πόσο δεσμευτικά εσείς ως κυβέρνηση και προσωπικά ως Υπουργός ερμηνεύετε τις συστάσεις της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα τώρα μερικά ζητήματα. Στις συστάσεις ε, της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει στην ε, παράταση και την αύξηση της ηλικίας επίσημης συνταξιοδότησης. Στο Βέλγιο αυτό δεν είναι σήμερα ζήτημα. Έχω την αίσθηση ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες αυτή τη στιγμή για να αυξηθεί η ουσιαστική ε, και όχι η νόμιμη ας πούμε ηλικία συνταξιοδότηση, η πραγματική ηλικία στην οποία βγαίνει ο κόσμος στη σύνταξη. Εσείς πώς το αξιολογείτε αυτό και πώς εξελίσσετε με βάση τις εξελίξεις και τις περιστάσεις. Ίσως είναι πολύ νωρίς από τώρα. Κάποια μηνύματα έχετε ε, λάβει, πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση. Επόμενο θέμα. Θετικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκκληση ε, να φύγει αυτή η τρομερή επιβάρηση από την εργασία και να επιβαρυνθεί το περιβάλλον, φορολογικά εννοώ, ε, εκτός ETS, δηλαδή ε, αυτοί που εξαιρούνται από το σύστημα ανταλλαγής δικαιωμάτων ρήπων, μεταφορές κλπ τον επόμενο μήνα ή το μεθεπόμενο έχετε ένα σχέδιο, σχέδιο για την ανάκαμψη που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση. Πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση, μετατοπίζεται δηλαδή η επιβάρηση της εργασίας, φεύγει από την εργασία και πηγαίνει στο περιβάλλον. Και θα το δούμε και στο σχέδιο προπολογισμού για το 2013, το οποίο έχετε εξαγγείλει για τον Ιούλιο. Υπάρχουν τέτοια μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Και ένα τελευταίο, ε, τελευταία ερώτηση. Διαβάζω στα κείμενα κάτι που με ανησυχεί για τα κεφάλαια τα τραπεζικά των βελγικών τραπεζών που λέει ότι χρειάζονται ενίσχυση. Βέβαια δεν είναι αυτό το θέμα, θέμα της κυβέρνησης, συμφωνώ, αλλά ξέρετε ότι στο Βέλγιο, και το είπατε και στην αρχή στην ομιλία σας, ε, ε, υπάρχει και δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, οι τεράστιες εγγυήσεις για την τέξια που σε περίπτωση που πάει στραβά η κρίση του ευρώ θα έρθει η κυβέρνηση να κληθεί να εξυπηρετήσει αυτές τις εγγύησεις. Μπορεί το κράτος να ταποκριθεί σε αυτό το θέμα, σε μια τέτοια δύσκολη κρίση και κατά αναλογία με τα όσα συνέβησαν ε, με τις ισπανικές τράπεζες. Δεν θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός εγγυήσεων και για άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Ένας μηχανισμός αλληλεγγύης ενδεχομένως και μεταξύ των τραπεζών των ιδίων. Γιατί καλό θα ήταν να αναλαμβάνει και τον κίνδυνο και το ρίσκο ο ίδιος ο κλάδος. Μέχρι εδώ ορισμένε παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης. Uh, Ίσως. Να τα πω αγγλικά ή ολλανδικά. Είναι πολύ ωραία να μπορώ να απαντήσω ε, στα ολλανδικά site. Ναι, βεβαίω έχουμε αλακώσει τον είναι πιο ήπιοι, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλά. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει κάποιε έντονε συστάσει, τι ακολουθεί, στη συνέχεια ε, λίγο τα μαζεύει και χαμηλώνει του τόνου. Ε, θα πρέπει, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συνεχίσουμε τις προσπάθειες στον δρόμο που ήδη έχουμε ε, αρχίσει. Ε, Βεβαίω είναι πιο ήπια σε σχέση με κάποιου άλλου που δεν κάνουν τίποτα, που βγαίνουν και του λένε δεν έχετε κάνει τίποτα. Έχει χαμηλώσει του τόνου, αλλά ε, ακόμα και η ήπια επιμένει. Είναι νέε επιλογέ πολιτικών θα πρέπει να επιβληθούν και δεν θα πρέπει ε, να επαναπαυθεί μια κυβέρνηση που μια κυβέρνηση έξι μηνών έχει λάβει κάποιε αποφάσει και είναι όλα ωραία και καλά. λοιπόν, δεν είναι ήπιος τόσο και μαλακός ο τόνος, είναι μεν ενθαρρυντικός, αλλά επίμονος ότι συνεχίστε τις προσπάθειες. Δεν σου λέει ότι μετά από λίγους μήνες θα έχει λήξει η υπόθεση και θα τα έχει όλα ρυθμίσει. Και πιστεύω ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να τονίσουμε τους στόχους και δέχεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είμαστε στο σωστό δρόμο Και βέβαια αυτά παραμένουν θέματα εθνική κυριαρχία, αλλά θέλω να πω και σε όλου του πολιτικού πρωταγωνιστέ που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την γνώμη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή δίνει συμβουλέ. Ε, σου χαράζει μια πορεία. Και δεν μπορούμε να ε, τα αγνοήσουμε και να θεωρήσουμε ότι είναι φιλολογίες. Καλό είναι να μιλάς για εθνική κυριαρχία και πολιτικές αποφάσεις, αλλά έχεις κάποιους στόχους που πρέπει να ε, καλύψεις. Και ο σημερινός Πρωθυπουργό και ο προηγούμενος ε, ανέκαθεν επέμεινε στην εθνική κυριαρχία του Βελγίου ότι εμείς θα ορίσουμε το δρόμο προς τους στόχους, αλλά ταυτόχρονα από πλευράς ε, συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι δεσμευτικές, διότι τα κράτη, οι μέλη έρχονται αντιμέτωπα με ελλείψεις, με προβλήματα και, που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν για την ηλικία συνταξιοδότησης και παράτηση. Έχετε δίκιο. Δεν είμαστε στο μοντέλο της Νορβηγίας που τα προσαρμόζει ε, ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής, δηλαδή όσο αυξάνει η ηλικία του πληθυσμού, αυξάνεται και η ηλικία συνταξιοδότησης, αυτόματα και δημογραφικά. Εμείς κοιτούμε την πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης και όχι αυτή που ορίζει ο νόμος. Και εκεί θα μπούμε σε ένα διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω να δείξει κατανόηση. Τώρα, να φύγει η επιβάρυνση φορολογική της εργασίας και να πάει στο περιβάλλον. 13 εκατομμύρια ήταν αυτό το εγχείρημα τον περασμένο Δεκέμβριο. Μαζί με τον έλεγχο του προπολογισμού που έγινε το Μάρτιο, Και είναι απάντηση αυτό στην σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα διαπιστώσατε ήδη ότι δεν αυξήθηκε η φορολόγηση εργασίας και το 3% του ΕΠ πρέπει να βρούμε από κάπου. Και αν το συγκρίνουμε με άλλους συναδέλφους είναι τεράστιο αυτό το εγχείρημα. Και θα πρέπει να διαπιστώσουμε και να ομολογήσουμε ότι στη φορολογία ε, είδαμε ε, το εισόδημα από κεφάλαιο, ε, κάποια υπηρεσιακά αυτοκίνητα που παρέχουν οι εταιρείε στους εργαζομένους και εκεί κοιτάξαμε να επιβαρύνουμε τη φορολογία ε, δυστυχώς μέχρι στιγμής ε, δεν είμαστε αποκλειστικά σε ε, κλάδους άσχετους με την εργασία, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλάς για ένα σχέδιο ανάκαμψη. Εγώ μιλώ πάντα για ένα σχέδιο ανταγωνιστικότητα και μεγέθυνση τη οικονομία. Το είπε είναι από τα στρατηγικά ατού αυτά του Βελγίου για την καταπολέμηση τη κρίση του 2008. Ακριβώ το γεγονό ότι δεν είχαμε μεγάλη επίβολα σχέδια ανάκαμψης γενικά του προπολογισμού. Αυτό μας βοήθησε να περάσουμε καλύτερα την κρίση ε, από ότι ε, αν είχαμε αυξήσει πολύ το έλλειμμα είναι πραγματικά κάτι που αποδίδει και τώρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο στο σχέδιο του Ιουλίου για την ε, μεγέθηση της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα να έχουμε στο μυαλό μας τη δημοσιονομική ε, ορθοδοξία. Όταν έχεις ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, ε, ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο για τις επιχειρήσεις, ότι ο δανεισμό, τα επιτόκια δεκαετία έχουν πέσει από το 5,8 στο 3,2. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο για τις εταιρείε. Για τις τράπεζες και τα κεφάλαιά του μπορώ να πω πολλά, αλλά ε, να μην μιλάμε για ευρωπαϊκή ε, αλληλεγγύη. Σήμερα ε, έχουμε και το σχέδιο της μόχλευσης και άλλους τομείς και, και πρέπει να κάνουν πολλά σε αυτό το τομέα όλα τα ευρωπαϊκά κράτη με ενίσχυση κεφαλαίκη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η ώρα τώρα να κάνουμε συγκρίσεις με άλλες χώρες. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και με τον Επίτροπο Αλμούνια και ε, θα προσπαθήσουμε το συντομότερο να εξασφαλίσουμε ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας στο Βέλγιο που ανέκαθεν ήταν πηγή ευημερία να μπορέσει να βοηθήσει την πραγματική οικονομία με πιο γερή κεφαλαϊκή βάση και με κανόνες που και εδώ ορίζονται και ε, επιβάλλονται πανευρωπαϊκά. Uh, uh, Ευχαριστούμε, η Σιλβή τώρα. Ευχαριστώ Σαρών, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την προσέλευσή σας. Ναι, εμείς με τη συζήτησή μας της εξαμέτρους σας φέραμε εδώ. Εγώ βέβαια δεν είμαι Βελγίδα, αλλά νομίζω ότι είναι καλό που δεν παραμένει εθνικό το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για τα μακροοικονομικά, που είναι επίσης από τις καινοτομίες της εξαμέτρου. Ένα διπλό ερώτημα. Πώς θα ανταποκριθείτε στο αίτημα της Κομισιόν σχετικώς, διότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες είναι ακόμη σοβαρότερες από τις δημοσιονομικές τι αυτές. Δηλαδή όλο και περισσότερο θα διαφέρει η πολιτική των χωρών μελών και δεν θα είναι πια ενιαία η νομισματική πολιτική έπειτα. Όπως είπατε πράγματι το Βέλγιο έχει παίξει πάντα επικοδομητικό ενωσιακό ρόλο αλλά στο Συμβούλιο Υπουργών, στο ΕΚΟΦΗΝ, πώς διασφαλίζεται κάποιον αμοιβαίο έλεγχο και σεβασμό έτσι ώστε αυτά που δεν καταφέραμε να κάνουμε τα πρώτα χρόνια του ευρώ να τα καταφέρουμε στα ύστερα δηλαδή να μπορέσουν όλες οι χώρες μαζί να προοδεύσουν. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Και θα αρχίσω από κάτι που ίσως να μην σας φαίνεται το σημαντικότερο από όλα, αλλά θέλω να επιμείνω επί του ότι ο διάλογος και στο ΕΚΟΦΗΝ και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με όλους τους παράγοντες εξαρτάται από τη δυνατότητά μας να συμφωνήσουμε επί του ποια είναι η πραγματικότητα. Σε πρώτη μορφή της έκθεσης της Κομισιόν ταυτιζόταν ως πρόβλημα για το Βέλγιο τα ιδιωτικά χρέη, το ιδιωτικό χρέος private indebtedness που λέμε και εμείς και αναρωτήθηκα πώς μπορεί να ταυτίζουν για μια χώρα ποιο είναι το ιδιωτικό χρέος. Το δημόσιο εντάξει, αλλά εμείς με τόσα πολλά κέντρα συντονισμού που έχουμε, μου απάντησαν δεν έχουμε τους ίδιους αριθμούς και στατιστικά στοιχεία για, όπως για τις άλλες χώρες, γι' αυτό βάλαμε τους ανεπεξέργαστους αριθμούς, αλλά έχουμε κάνει λέει μια υποσημείωση, έτσι μου είπανε. Εγώ νομίζω ότι αν θέλουμε πραγματικό διάλογο πρέπει να έχουμε ένα πολύ αξιόπιστο στατιστικό σύστημα που να μην επιτρέπει σε οποιονδήποτε να κρύβεται πίσω από τους αριθμούς αυτούς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό που είπα. Έπειτα, όταν ρωτάτε για ποιο θέμα να επιμείνουμε ιδιαίτερα, θα έλεγα ως πρώην υπουργό Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου ότι το Βέλγιο τα τελευταία πέντε χρόνια έχει χάσει 5% του μεριδίου αγορών της στην διεθνή αγορά. Αλλά και άλλες χώρες, και άλλες. Άλλοι 15, 16, 17, 14. Όλοι το πάθαμε αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται μια πολύ πιο φιλόδοξη στρατηγική που να μην βασίζεται μόνο στο πώς θα δαπανίσουμε τι, αλλά και στο πώς θα βάλουμε τις επιχειρήσεις μας σε μια θέση όπου θα είναι ικανές να δημιουργήσουν ανάπτυξη, όπου βρίσκεται αυτή. Υπάρχει μένει η ενιαία αγορά, αλλά χρειάζεται ισχυρή θέση και ως προς τη διεθνή αγορά. Κατ' εμέ, οι μακροοικονομικές αυτές ανισότητες, macroeconomic imbalances, είναι για το Βέλγιο ειδικά κάτι αρκετά θετικό. Δηλαδή, όπως είπε και ο κύριος Χαντράουι, υπάρχει το θέμα που έθιξε, αλλά η μυθολογική ανταγωνιστικότητα της χώρας μας σε σύγκριση με τρεις γειτονικέ χώρες, Ολλανδία, Γαλλία, δεν είναι σε άσκημη θέση ως προς την τιμαριθμική αναπροσαρμογή τουλάχιστον. Άρα δεν χάσαμε ανταγωνιστικότητα. Χάσαμε μόνο σε σχέση με τη Γερμανία, αλλά όλοι χάσαμε σε σχέση με οικονομίες εκτός της Ένωσης επίσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να το λύσουμε και ως προς το κόστος αλλά και ως προς την παραγωγικότητα. Να δούμε δηλαδή τι μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Φίλιππος Λαμπέρ. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε στις Βρυξέλλες κύριε Υπουργέ, αλλά μετά στα γαλλικά γιατί είναι η μητρική μου. Και θα συνεχίσω πάνω στη γραμμή που ξεκίνησε η Σίλβια. το Βέλγιο είναι μια χώρα που ίσως περισσότερο από το μερτικό τόσο αφορά συστημικά χρηματιστικά ιδρύματα. Είμαστε μικρή χώρα που συναθρίζει πολλού μεγάλους χρηματιστικού φορείς που ε, ε, βρέθηκαν σε δύσκολη θέση στην αρχή της χρηματοστικής κρίσης. Ανήκατε ε, σε μια κυβέρνηση που έδωσε του ύψους 15% ΑΕΠ του Βελγίου σε ένα μόνο τέτοιο χρηματιστικό ίδρυμα. Δεν ξέρω αν ήταν υπεύθυνη στάση αυτή είτε όχι αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το Βέλγιο κινδύνευσε τα δημοσιονομικά του κινδύνευσαν από την κακή δημοσιονομική προσέγγιση και επιχειρησιακή λειτουργία των πεζικών ομίλων. Το ερώτημα μου το εξή. Είναι μέλος του Συμβουλίου. Διαπραγματευόμαστε την οδηγία που θα θέσει πολύ περιοριστικούς όρους στις τράπεζες, διαπιστώνω ότι το Κοινοβούλιο πήρε μια σημαντική, πιο, σημαντικά πιο φιλόδοξη θέση σε σχέση με το Συμβούλιο όσον αφορά τους ίδιους πόρους, αμοιβέ, ρευστότητα, επίλυση τραπεζικών κρίσεων κλπ. κλπ. Εμείς εδώ και αρκετές εβδομάδες που διαπραγματευόμεθα χτυπάμε σε ένα Συμβούλιο που δεν μετακινεί τη θέση του ε, και δεν είναι πιο ευέλικτο. Και δεν ξέρω ποια θέση του Βελγίου στο Συμβούλιο. Ανήκεται σε εκείνου όπω και εκείνοι, όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, που ζητούν να υπάρχουν πιο μεγάλε απαιτήσει από αυτέ τη Βασιλεία 3 και από αυτέ που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ή αντιθέτω, ε, έχετε μια στάση που λέτε ότι θέλετε να δημιουργείτε αναταραχέ, ε, να μην ε, κινδυνεύσει το σκάφο και θέλουμε μια ρύθμιση στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Απάντηση να σα πω ότι αποφεύγω πάντα να χρησιμοποιώ τη λέξη μικρή και χώρα μου σε μία φράση. Θεωρώ ότι είμαστε μία μετρίου μεγέθους χώρα ε, απλευράς οικονομικής, ε, σε μέγεθος εννοώ, αλλά οικονομικά δεν είμαστε μικρή χώρα. Τώρα όσον αφορά τη συζήτηση ε, για τις, αν θα είναι πιο φιλόδοξη η στάση του Κοινοβουλίου από ό,τι αλλού για τα μέτρα που συζητάμε. Θεωρώ ότι αυτός είναι και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι φιλόδοξο. Τούτου λεχθέντος δεν είμαι απόλυτα βέβαιο ότι η βούληση να καταλήξουμε σε κάτι που θα επιτρέψει πραγματικά όχι μόνο σε επίπεδο λόγων αλλά και έργων να πετύχουμε κάποια συνένεση που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε αυτό μπορεί να θεωρηθεί και φιλοδοξία. Είναι... Θέλουμε την ομοφωνία διακόπτη ο μιλητής. Ναι, στο κοινοβούλιο σας συγχαίρω, αλλά στο συμβούλιο υπάρχουν άλλοι κανόνες του παιχνιδιού και κυρίως όσον αφορά μεταρρυθμίσεις στο χρηματοστικό τομέα. Πρέπει να έχει κανείς υπόψη του πάντα τους μικρούς κινδύνους ε, μεταγκατάστασης, ε, εάν κάποιοι φύγουν, κάποιοι δεν συμφωνήσουν ε, κλπ. Θέλουμε να έχουμε τη μέγιστη υποστήριξη. Να καταλήξουμε σε κάτι θα ατύχει τη μεγαλύτερη υποστήριξη. Ξανά διακοπή. Είμαστε φιλόδοξοι, αλλά όχι τόσο υπεύθυνοι πολιτικώ. Είστε λιγότεροι φιλόδοξοι γιατί είστε πιο υπεύθυνοι πολιτικά. Διακόπτω Δεν τολμώ να το πω αυτό, λέω. Ο κ. Δημόσιο τη Βελική Κυβερνήσεω. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι σε επίπεδο Συμβουλίου. Αυτή ε, η επιμονή με την οποία πρέπει να επιδιώξουμε common ground, το κοινό έδαφος, Μα μονίμως μας λένε ότι δεν είμαστε τόσο σοβαροί όσο εκείνοι. Είναι ο εισηγητής, λέει, πρόεδρος που διακόπτει, ο κύριος Κάρας. Ή δεν εκφράστηκα καλά. Ε, μου δεν καταλαβαίνει γιατί αντιδράτε έτσι. Ε, να απαντήσω σε αυτό, στα αγγλικά, λέει ο κύριος Αντιπρός Κυβέρνησης. Τι προσπαθώ να εξηγήσω δεν προσπαθώ να, να, θεωρήσω, να χαρακτηρίσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να θεωρήσω πιο φιλόδοξο, λιγότερο φιλόδοξο, ότι ανησυχεί περισσότερο, λιγότερο, σε σχέση με τις φιλοδοξίες που συζητάμε. Καθόλου. Λέω, η λογική της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων διαφέρει στο Συμβούλιο εν συγκρίση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι εντροπή, απλώς είναι να γνωρίζουμε ποιος είναι ο ρόλος του καθενός, ότι είναι διαφορετική ρόλη. Όσον αφορά την ε, μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού τομέα, Θέλουμε να βρούμε κοινό έδαφος μεταξύ κρατών μελών που έχουν διαφορετικά οράματα σχετικά με το ε, δέον να γίνει. Κυρίως όσον αφορά τη χρηματοδοτική μεταρρύθμιση, για μας τους Βέλγους ε, είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση ή δυνατόν ομοφωνία. Να συμφωνήσουν οι περισσότερε χώρε. Ο φόρο χρηματοστικών ε, συναλλαγών, Φερρυπίν. Για να δώσω ένα παρόμοιο παράδειγμα. Για εμά του Βέλγου Όσον αφορά τη δήλωση τη νέα κυβερνήσεω, ο φόρο χρηματοστικών ε, συναλλαγών είναι κάτι που υποστηρίζουμε απόλυτα. Για να το πετύχουμε όμω, για να το εφαρμόσουμε, πρέπει να κινηθούμε ούτω ώστε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τι περισσότερε χώρε για να είμαστε ρεαλιστέ. Ακόμα και όταν συμφωνούμε με τη φιλοδοξία, γι' αυτό ακολουθούνται διαφορετικέ προσεγγίσεις. Δεν ξέρω αν σα απάντησα απόλυτα σε αυτό που με ρωτήσατε. Α, έχω την εντύπωση να κάνει προτάσει. Λέτε ότι δεν θέλετε να κινούμαστε μόνοι, αλλά εδώ και 10, 20, 30 χρόνια το Βέλγιο ε, ήταν πιο τολμηρό προτάσει από ότι είναι σήμερα. Να πω κάτι άλλο, λέω και Αντιπρό Κυβερνήσεω, για τη λέξη χαλαρή προσέγγιση. Χαλαρό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή. Εγώ είχα προτείνει στο Συμβούλιο να υιοθετηθεί μια τροπολογία που προερχόταν νομίζω και αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε πει όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις θα πρέπει να φροντίσουμε ούτω ώστε η στάθμιση αυτών των πιστώσεων να μην βαρύνει 100% τα liquidity rules, τους κανόνες περιευστότητας. Από τη στιγμή που ο Βέλγος υπουργό σα μίλησε και το πρότεινε, δεν έγινε αποδεκτό το σημείο. Μπορούμε να πούμε ότι μειώντα το 100% εξαγωγικών πιστώσεων προς 50 και 25% ότι ήμουν πιο χαλαρός, πιο υποχωρητικός, αυτό θεωρείτε όχι. Νομίζω ότι τροποποιώντας τους κανόνες μπορούμε καλύτερα εκ των προτέρων να εγγυηθούμε ότι οι κανόνες λειτουργούν υπέρ της πραγματικής οικονομίας. Και γνωρίζοντας ποια είναι η σημασία των εξαγωγικών μας δυνατοτήτων, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τις επιχειρήσεις, είμαι περήφανος που το υπερασπίστηκα αυτό σαν θέση. Εξάλλου, υπησέρχεται αυτό στην λογική που υπερασπίστηκε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είναι ένα παράδειγμα που όπω φαίνεται το Συμβούλιο δεν ήθελε να προχωρήσει τόσο μακριά. Το Συμβούλιο, ζητώ συγγνώμη μιλητή, δεν ήθελε να προχωρήσει τόσο μακριά στο το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό είναι κανείς πιο υποχωρητικό, ε, δεν νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλοσύνη σας που μπήκατε στις ε, λεπτομέρειες του θέματος αυτού, του CRD που δεν έχετε και την Προεδρία του Συμβουλίου, δεν είστε Προεδρεύων. Εντάξει, καλά τα καταφέρατε και ελπίζουμε να μας βοηθήσετε περισσότερο και στις άλλες φιλοδοξίες ε, που έχει το Κοινοβούλιο. Ο Ντέρκ Ιαν Έπινγκ είναι ο επόμενος που λόγο. Κύριε Βανάκερε, καταρχάς θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμότατα εξ ονόματος της βελγικής αντιπροσωπείας των Ευρωπαίων μεταρρυθμιστών και συντηρητικών. Ποιο είναι το σημαντικότερο για τη βελγική ε, ε, ανταγωνιστικότητα. Το μεγαλύτερο ατού του Βελγίου είναι η γεωγραφική του θέση για να μπορεί ε, να παίζει ένα ρόλο κλειδί ε, στην ευρωπαϊκή οικονομία. Όταν σας άκουγα Μα ακουστήκατε λίγο θριαμβευτής ότι δεν έχουμε προβλήματα ενώ πριν από μερικά χρόνια είχαμε και όλα αυτά ε, λύθηκαν και έλειωσαν οι φόβοι. Η Ντέξια υπό την εποπτεία του συναδέλφου κυρίου ε, Ντεχάνε γνώρισε μεγάλες δυσκολίες και χρειαζόταν οπωσδήποτε βοήθεια από ε, το βελγικό κράτος εγγύτη και ε, πραγματικά αυτό είναι πολύ μεγάλη επιβάρηση για το κράτος. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής και έχει να κάνει με μια ιδιαιτερότητα, ε, μάλλον με τις ειδικές συστάσεις για τη χώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαβάζουμε διάφορα πράγματα και βλέπουμε συχνά να επανέρχεται η τιμαριθμική αναπροσαρμογή του μισθού που ανέφερε και ο συνάδελφος από τη Σοσιαλιστική Ομάδα η διάρκεια της ανεργίας ε, με εκθέσεις διεθνών οργανώσεων και η πολύ χαμηλή ε, συμμετοχή της αγοράς εργασίας στην πραγματική οικονομία. Αυτά είναι προβλήματα που συνδέονται όλα με ένα πράγμα που είναι η ισχυρή θέση των συνδικάτων στην κοινωνία. Ρώτησα και τον κύριο Ρεν που δυστυχώς δεν απάντησε, παρέλειψε να απαντήσει σε αυτό το θέμα και το, το υπέδειξα ξανά. Βέβαια, όταν έχει κάποιο ε, προθέσεις να κάνει οικονομικές μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να φανταστεί τη Γερμανία πριν από μια δεκαετία. Θυμάστε ποια ήταν η θέση και ο καγκελάριο Σρέντερ κατάφερε να επιβάλλει μεταρρυθμίσεις με την υποστήριξη των συνδικάτων και έχω καμιά φορά την εντύπωση ότι τα συνδικάτα στο Βέλγιο και μάλιστα τα βαλονικά συνδικάτα που είναι πολύ πιο ακραία από τα φλαμανδικά, και ε, εσάς σας εντάσσουν ε, στο γενετικό υλικό και στην ομάδα αίματος του ΑΣΕΒΕ, του Καθολικού Φλαμανδικού Συνδικάτου. Ε, γίνονται λοιπόν μεγάλες δράσεις και αντιδράσεις, απεργίες, καταλήψεις εργοστασίων, κρατούν όμοιρους τους μάνατζερ και τους διευθυντές, δεν είναι αυτά τα πράγματα ευχάριστα. Λοιπόν, στις συστάσεις που είναι ειδικέ για τη χώρα, ε, γίνεται λόγος και για τα συνδικάτα, αλλά αυτό ε, κάπως το παρακάμπτουμε, το αποφεύγουμε συνεχώς, είναι ταμπού, δεν το συζητάμε. Ε, είναι αυτό που λένε στα αγγλικά ένας ελέφαντας ο οποίος θεωρείται στο χώρο και κάνουν όλοι όπως δεν το βλέπουν. Λοιπόν, γιατί το αποφεύγετε αυτό το θέμα, τι θα γίνει, πώς μπορείτε λίγο να περιορίσετε την εξουσία των συνδικάτων. Κύριε Έπινγκ. Έχω την αίσθηση ότι η εικόνα που περιγράφεται δεν είναι πια ε, ακριβή η εικόνα. Ο ελέφαντας αυτός δεν είναι ούτε στο σαλόνι ούτε στην αίθουσα, είναι στον κήπο και οδεύει προς το ζωολογικό κήπο. Δεν λαμβάνεται υπόψη με αυτό το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου ας πούμε ε, ε, ε, τα επιδόματα ανεργίας θα βαίνουν μειούμενα. Έχουμε κάνει κινήσεις. Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι όταν υπάρχει κατάλληλη προσφορά εργασίας για έναν άνεργο σήμερα, ε, μέχρι 60 χιλιόμετρα θα είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει και να δέχεται αυτή τη θέση εργασίας. Στο παρελθόν ε, συνέβαινε πάρα πολύ λιγότερο. Όλα αυτά τα μέσα που αφορούν λοιπόν την αύξηση της απασχόλησης ή την αύξηση ε, της ηλικίας συνταξιοδότησης, να μην είναι πια ελκυστική η αποχώρηση από την εργασία σε χαμηλότερη ηλικία. Να παραμένει ο κόσμος στη δουλειά και να φροντίζουμε και τα επιδόματα ανεργίας να μειώνονται προοδευτικά. Όλα αυτά είναι απαντήσεις λοιπόν σε αυτό που πραγματικά αναφέρεται και περιγράφεται στην ανάλυση. Με αλφαγιώτα. Και αυτό που ανέφερε και ο κύριος Αλχαντράουι. Σήμερα το ύφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στο Βέλγιο είναι πιο ήπιο Δεν είπα εγώ ότι είναι όλα εντάξει. Μήπως δεν με ακούσατε προσεκτικά ε, στην εισαγωγική μου τοποθέτηση. Γιατί το τόνισα ότι αυτή η άσκηση δεν είναι κάτι που μπορείς να πεις ε, μετά από έξι μήνες ότι εντάξει τα καταφέραμε και σταυρώνουμε τα χέρια μας και είναι εντάξει. Το είπα τρεις-τέσσερις φορές ε, κόντεψα ο ίδιος να βαρεθώ από αυτά που έλεγα. Καθόλου δεν θεαβολογώ ότι είναι όλα τα προβλήματα λιμένα και όλα καλά και όλα ωραία. Απλώς αναγνωρίστε ότι αυτό που είπατε με τον ελέφαντα δεν είναι πια στο σπίτι μας, είναι έξω και το στέλνουμε και στο ζωολογικό κήπο, προσεχώς. Και επίση όλα αυτά που κάνουμε δεν τα κάνουμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά για τους Βέλγους. Και είναι ο καλύτερο τρόπο να βγούμε από την κρίση, είμαι πεπισμένο. Για θριαβολογία δεν νομίζω, μάλλον λάθο κάνετε. Αλλά μην λέμε ότι δεν έγινε και τίποτα το τελευταίο εξάμεινο, γιατί και αυτό είναι λάθος. Thank you. Θέλεις να πεις κάτι. Έχω ένα κατάλογο, εντάξει. Ήθελα να ξέρω μήπως θέλει και κανείς να μιλήσει από την ΚΟΕ. Ναι, ο Γιούργεν, ο Γιούργεν, να τον γράψω. Φίλιπ Ντεμπάκερ Περβάνς, Ποιος άλλος είναι. Ναι και σένα σε είδα Λεόντα. Ο Γιούργεν. Γιούργεν Κλούτα. Ευχαριστώ Σάρα. Θα ήθελα να επανέλθω στην ΆΤΑ, την αυτόματη τη μαριθμική αναπροσαρμογή. Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη για το ίντεξ. Από πλευράς των εργαζομένων, βεβαίως, είναι κάτι το θετικό και το καλωσορίζουν οι εργαζόμενοι, αλλά από εκεί και πέρα έχει και πολιτική σημασία. Το είπε και ο Σαΐτ προηγουμένως. Είναι ένα μέσο αποτελεσματικό για να αποφευθεί η φτώχεια. Η καταπολέμηση και η πρόληψη της φτώχειας είναι και στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν σας καλέσουν αυτό το μέσο να το μεταρρυθμίσετε, να το ξανασκεφτείτε, θα με ενδιαφέρει πώς θέλετε να το κάνετε χωρίς να θίξετε ή να απεμπολίσετε αυτά τα θετικά, γιατί τονίζεται και η αγοραστική δύναμη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε σύσταση στη Γερμανία που είναι η χώρα μου να προσαρμόσουν λέει τους μισθούς στην εξέλιξη της παραγωγικότητας για να αυξηθεί η εσωτερική ζήτηση και η αγοριστική δύναμη και να έρθουν κάποιες ανισορροπίες στο εσωτερικό της χώρας. Με εκπλήσει λίγο λοιπόν αυτή η σύσταση και θέλω να μου πείτε πώς θα το κάνετε. Και το δεύτερο φορά τη φορολόγηση. Να περάσει λοιπόν η φορολόγηση από τους άμεσους φόρους περισσότερα στους έμεσους. Κατά την άποψή μου όμως εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος άνθρωποι χαμηλού εισοδήματος να πληγούν ε, ιδιαίτερα και να επιβαρυνθούν ε, από ότι οι πιο εύποροι. Γιατί είναι λογικό γενικότερα να συμμετέχουν οι πιο πλούσιοι περισσότερο στα δημόσια οικονομικά από ότι οι φτωχότεροι και όχι με έμεσους φόρους που επιβαρύνουν τους πάντες. Και επίση μας δώσετε κάτι στατιστικές και τις κοίταξα και εκεί το Βέλγιο στο χρέος βρίσκεται λίγο ε, πάνω από τον ευρωπαϊκό όρο λίγο, όχι πολύ δραματικά. Από την άλλη όμως το Βέλγιο είναι πολύ μεγάλη ιδιωτική περιουσία και στη στατιστική εδώ έχουμε το μεγαλύτερο εισόδημα ή περιουσία ανα στο Βέλγιο. Έχετε σκεφτεί κανένα φόρο περιουσίας να επιβάλλετε ε, για να μειωθούν αυτές ε, οι ανισότητες και τα έλλειμματα. Ευχαριστώ. ich möchte versuchen... Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα γερμανικά. Όχι, στα αγγλικά. Κατανοώ, καταλαβαίνω γερμανικά, αλλά δεν τα μιλώ τόσο καλά. Äh, Πρώτον, ας αφορά το σύστημα τιμαριθμικής ε, προσαρμογή Πράγματι, αν ρίξει κανεί μια ματιά και δει τους φτωχού εργαζόμενους στη χώρα μα, είναι πολύ μικρό ποσοστό σε σύγκριση με άλλες οικονομίες που έχουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα ο αριθμός των εργαζομένων φτωχών είναι σχετικά περιορισμένος και μπορεί να πει κανείς ότι η αριθμική αναρρύθμιση είναι ένα σύστημα που εξασφαλίζει επάρκεια εσόδων των οικοκυριών. Όταν μιλάμε για αυτόματους σταθεροποιητές, κάτι που είδατε στο γράφημα, είδαμε ότι όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, το Βέλγιο τα πήγε αρκετά καλά, πιθανότατα ανάμεσα στους ε, οικονομικούς σταθεροποιητές και αυτόματη μαριθμική αναρρύθμιση ε, ε, προσαρμογή μπορεί να θεωρηθεί ένας από τους παράγοντες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα πρέπει η λογική που ακολουθείται είναι σωστή. Δηλαδή οι αμοιβέ θα πρέπει να μετακινούνται ανάλογα με την ανάπτυξη παραγωγικότητας. Η ίδια συμβουλή που δόθηκε και στη Γερμανία δόθηκε σε εμά. Είναι κρίσιμος παράγοντα. Όσον αφορά τη σύγκριση με τη Γαλλία και την Ολλανδία, όπω έλεγε ο φιλελεύθερο συνάδελφο, δεν έχουν σύστημα τιμαριθμική προσαρμογή και δεν απολέσθη ανταγωνιστικότητα την τελευταία διετία. Και η πειθαρχία στις κοινωνικές, στον κοινωνικό διάλογο είναι κάτι πιο σημαντικό από το σύστημα τιμαριθμικής προσαρμογής. Τι πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από κάθε χώρα, σαν συμβουλή δηλαδή ότι η εξέλιξη των αμοιβών και η εξέλιξη των, της παραγωγικότητας ε, θυγραμμίζονται. Έχουν αντιστοιχεία. Και συμφωνώ με αυτούς που είπαν ότι είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας. Να δουν ποια λογική ακολουθείται στον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Ο κ. Σέπινγκ λέει ότι δεν υπάρχει Απάντηση όσον αφορά το βαθμό εξουσία δύναμη που έχουν τα συνδικάτα στι διαπραγματεύσει. Εγώ λέω α δούμε μια ματιά και να δούμε κατά πόσο θα επιτεθεί κοινωνική συνένεση. Με ένα πρόγραμμα πάνω από 3% του ΑΕΠ που είναι τεράστιο ποσό. 3% του ΑΕΠ σε ένα έτο ε, οικονομικό. Δεν το έκαναν πολλά κάτι μέλη αυτό. Αν δείτε και την κοινωνική συνένεση που επεκράτησε στη χώρα μου, νομίζω ότι είναι ένα σύστημα που έχει κάποια αξία αυτό που εφαρμόστηκε. Όσον αφορά το άλλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά λέει ότι το κόστος εργασίας και η φορολόγηση αυτού του κόστους πιθανότατα είναι ε, πολύ υψηλή και χρειάζεται επανεξισορρόπηση ίσως εξετάζοντας τι άλλο μπορεί να φορολογηθεί πέρα από την εργασία. Βλέποντας όμως τη οικονομική κατάσταση της χώρας μου και την οικονομική εξυγίανση που ακολουθείται, είμαι πεπισμένος προσωπικά ότι σε πρώτο βαθμό πρέπει να φτάσουμε στο 2015 με ε, ισολογισμένο προπολογισμό. Και αυτό ζητά ήδη τεράστιες προσπάθειες. Όχι μόνο πλευράς δαπανών, αλλά εν μέρη και στα έσοδα τι ούτω τρόπος και ταυτοχρόνως προσθέτοντας και άλλες προσπάθειες, ούτως ώστε να δημιουργηθεί χώρος για μείωση του εργατικού κόστους μέσω χαμηλότερης φορολόγησης θα είναι ένα έργο δυσκολότατο. Γιατί? Διότι ζω σε μια χώρα όπου περίπου 40-50% του λαού ζει σε ακτίνα 15 χιλιόμετρων από σύνορα μπορείτε να μου ζητήσετε να είμαι πολύ προσεκτικός και έξυπνος όσον αφορά τις αλλαγές της φορολόγησης, τις επιλογές φορολόγησης διαφόρων κατηγοριών, όμως η μετεγκατάσταση είναι και αυτός ένας παράγοντας στη ζωή. Όσον αφορά το ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη, η φορολόγηση εισοδήματος από κεφάλαιο. Ξέρω ότι αυτό το κοινοβούλιο, και το εκτιμώ αυτό, είναι πολύ άσχολο θέλει να επικρατούν δίκαιες συνθήκες στον τομέα αυτό. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν φτάσαμε ακόμα εκεί. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι κάποιες επιλογές που κάνουμε έχουν αντίκτυπο στη φορολογική βάση. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά αυτό το θέμα. Καλώ, ευχαριστώ. λέει ναι, κυρία Μπόλτ, έχω άλλου τρει ομιλητέ φίλε, Ντεμπάκε, Προβάν Σουμπερέ και Λίαμ Βανκόκ. Εκεί κλείνει ο κατάλογος. Ο Φιλίπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Υπουργό που ήρθε. Έχουν υποθεί πολλά και δεν θέλω να κάνω κανένα βέλγο-βελγικό παιχνίδι σήμερα, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που αν δει κανείς από το ευρωπαϊκό πρίσμα στο Βέλγιο, υπάρχουν και μερικά πράγματα που δεν ακούστηκαν. Είπατε ότι έχετε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, μήνες, ε, χρόνια για μεταρρυθμίσεις και ε, για τη δημοσιονομική εξυγένση και να είναι ισοσκελισμένος ο περιοπολογισμός το 2015. Βλέπουμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι τα ε, σενάρια που προβλέπεται για το 2014 και το 2015 είναι υπεραισιόδοξα και οι μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να οδηγήσουν σε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς δεν έχουν ακόμα εκπονηθεί και σε σχέση με τη συζήτηση που γίνεται τώρα για την ανάκαμψη της οικονομίας, όπως είπατε για το σχέδιο ε, ανταγωνιστικότητας και μεγέθυνσης της οικονομίας που για μένα είναι καλύτερος όρος, αλλά πώς θα γίνουν ε, οι προσαρμογές, τι ε, προσπάθειες απαιτούνται από το Βέλγιο και ποιες μεταρρυθμίσεις θα γίνουν τα επόμενα χρόνια σε αυτό το σχέδιο για την ανταγωνιστικότητα. Πώς να το φανταστούμε, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές σας, ποια είναι τα πρώτα μηνύματα που διαβάζω και λαμβάνω είναι αντιφατικά και σε σχέση ε, με αυτά που σύστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας. Μια δεύτερη ερώτηση, ίσως τεχνική, αλλά δεν είναι ασήμαντη. Το είπατε κι εσείς. Γίνεται συζήτηση για την περιπλοκότητα της κρατικής μεταρρύθμισης του κράτους στη χώρα μας. Ε, είναι διάφορα τα επίπεδα, τοπική αυτοδιοίκηση, επαρχίες, περιφέρειες και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Όλοι έχουν ξεχωριστούς προπολογισμού που θα πρέπει να συντονίζονται μεταξύ τους. Είδαμε και τους περασμένους μήνες τι σημαίνει αυτό και στην περίπτωση της Ισπανίας με τις περιφέρειές της. Εσείς τι κάνετε έτσι ώστε και στο εσωτερικό να έχετε καλύτερη εποπτεία και καλύτερο συντονισμό και πρώτερη συνεννόηση σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο για να γίνονται καλύτερα οι προπολογισμοί και πιο συνδυασμένοι. Ξέρω ότι με το νέο σύμφωνο για τη χρηματοδότηση, έγινε μια συμφωνία ε, με τις περιφέρειες, αλλά είναι σημαντικό επίσης να μην χάνουμε ε, και τις ε, τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις και τι προσπάθειες κάνουν και αυτές. Και ένα τελευταίο ερώτημα, πολύ συγκεκριμένο, για κάποιες μεταρρυθμίσεις. Μιλήσατε για την ανταγωνιστικότητα και τους μισθούς. Ταυτόχρονα όμως βλέπω ότι αυτό συνδέεται με πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα. Συχνά έχω την αίσθηση ότι το Βέλγιο προσπαθεί πολύ λίγο να προσαρμόσει τα επενδυτικά του προγράμματα, τις μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με ε, τον κοινοτικό προπολογισμό. Σε λίγο θα έρθει η νέα προγραμματική περίοδος των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών γιατί το Βέλγιο δεν επιζητεί περισσότερα κονδύλια ε, στις μεταφορές, στην εφοδιαστική, ε, στην έρευνα, στην καινοτομία; Υπάρχουν κονδύλια ευρωπαϊκά τα οποία πολύ λίγο εμείς επιζητούμε ε, για να συμμετέχουμε ως Βέλγιο. Ευχαριστώ. Κύριε Ντεμπάκερ, σας ευχαριστώ που δεν θελετε βελγοβελγική βέλγο-βελγική συζήτηση, αλλά αυτά που με ρωτήσατε είναι τελείως εσωτερικά και στο Βελγικό Κοινοβούλιο. Ε, η βελγική στρατηγική, και δεν θέλω να την αποκαλύψω τελείως εδώ, είναι πολύ ε, σημαντική και βασίζεται, και θέλω να το πω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, σε μια πάρα πολύ καλή πρόβλεψη και εκτίμηση το τι μπορεί να σημαίνει για μας το σχέδιο Ευρώπη 2020. Όταν κάνουμε μια στρατηγική, αυτό δεν είναι μια διανοητική συζήτηση φιλολογική. Πρέπει να το συνδέσουμε με τη στρατηγική το 2020, αλλιώς κάνουμε λάθος. Δεν λέω ότι δεν μπορούμε να έχουμε ή δεν πρέπει ξεχωριστή στρατηγική κράτος μέλος, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα ο καθένας να έχει εθνικές στρατηγικές που να μην λαμβάνουν ε, τουλάχιστον υπόψη τη στρατηγική της Λισαβόνας και το 2020. Αυτό θα πρέπει να γίνει κτήμα ιδιοκτησία όχι μόνο της Ένωσης αλλά και των 27 κρατών μελών. Ξέρετε τα συστατικά αυτής της στρατηγικής και εμείς ε, τα λαμβάνουμε υπόψη και τα συνυπολογίζουμε. Και το τελευταίο εξάμεινο σε αυτή τη σύντομη θητεία που θα είναι 30 μήνες μόνο γιατί είδαμε και πάθαμε να φτιάξουμε κυβέρνηση Αυτούς τους 30 μήνες που μας απομένουν θα τους αξιοποιήσουμε για να επιμείνουμε εκεί. Για τη μεταρρύθμιση του κράτους. Ξέρετε ότι το σχέδιο σταθερότητας που υποβάλλουμε το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ με τις περιφέρειες και τις ε, ε, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για μεγαλύτερη ε, οικονομική ε, ανεξαρτησία, προσαρμογή του νόμου χρηματοδότησης για να έχουν και εκείνη ευθύνη στη στρατηγική εξυγίανση των οικονομικών μας. Συμβαίνει αυτό σήμερα και είμαι πεπισμένος ότι οι ευαισθησίες όσο και η συνειδητοποίηση της ευθύνης από τις περιφέρειες και μετά από την τόση πίεση που έχει γίνει στη δημόσια συζήτηση έχει αυξηθεί. Και το βλέπω και με τους ε, πρωθυπουργούς των περιφερειών του Βελγίου και ε, τους ε, ομολόγους μου υπουργούς οικονομικών των περιφερειών. Σε μια ομοσπονδιακή χώρα ο καθένας θα πρέπει να κάνει τα καθήκοντά του, να βάλει το λιθαράκι του και τελικά θα υπάρξει και μεγάλη πολιτική κύρωση και σοβαρή σε εκείνον που δεν το κάνει. Τώρα κατά πόσο συμμετέχουμε αρκετά στα κοινοτικά προγράμματα. Όταν ήμουν υπουργό εξωτερικών, το άκουγα σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο καθένας νόμιζε ότι δεν αξιοποιεί σωστά τα ευρωπαϊκά προγράμματα και, τα, ε, και επαρκώς. Και με εκπλήσει που το ακούω και στο Βέλγιο. Σίγουρα οι περιφέρειες και ε, η τοπική αυτοδιοίκηση απευθύνεται και στα ευρωπαϊκά προγράμματα και τη χρηματοδότηση, αλλά γιατί η χώρα μας νομίζω σε γενικές γραμμές καλά τα πάμε. Κυρίως σε τέτοιους καιρούς. Όπου γίνεται μεγάλος λόγος για το τι κάνει η Ένωση και τι μπορεί να κάνει ο προπολογισμό της. Και με εκπλήσει που πολλοί ε, δεν έχουν την ίδια άποψη για τον κοινοτικό προπολογισμό με το Βέλγιο. Εμεί θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ένα σοβαρό, ένα αξιοπρεπή προπολογισμό. Δεν το θεωρούν όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών αυτό. Αυξάνεται πάντα η φιλοδοξία μα και όλα αυτά που θέλουμε να κάνει ο κοινοτικό προπολογισμό και παραμένει στο πενιχρό 1% του ΑΕΠ. Είναι απορία άξιο αυτό. Πάντως προσωπικά πιστεύω ότι αν εφαρμόσουμε όλα αυτά που πρέπει να κάνει μια χώρα σαν το Βέλγιο, συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα, ε, δεν χρειάζεται να θεωρούμε ε, ότι θα Δεν έχω αυτή την αντίληψη. Μπορεί να διαφέρουμε, δεν λέω. Euh, Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα σας ρωτήσω κάτι όχι για το Βέλγιο, αλλά για τις συστάσεις που γίνονται αναχώρα για το σύνολο της Ευρωζώνης. Ζητούμε περισσότερο συντονισμό και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτές οι συγκεκριμένες στάσεις χώρα πρέπει να συμβάλλουν και αυτές στο συντονισμό. Αλλά από το Μάστριχτ ο συντονισμός των οικονομικών προγραμμάτων δεν έχει και πολύ πετύχει. Ο συνδυασμός δηλαδή κεντρικής διακυβέρνησης και επικουρικότητας και οι εθνικοί βουλευτές και οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν με τον τρόπο τους αυτά που αποφασίζουν οι Τι θεωρείτε λοιπόν ότι πέτυχε η Κομισιόν εφέτος ή μάλλον για τη χώρα μου θέλω να πω ότι δημοσίευσε συστάσεις με ένα ενημερωμένο λέει έγγραφο της προηγούμενης κυβέρνησης στις 4 Μαΐου. Το έγγραφο δημοσιεύτηκε αγγλικά και ποτέ, καμία στιγμή, κανένα του κομμάτι δεν λέει, δεν κάνει λόγο για τον προγραμματισμό μιας κυβέρνησης που τότε είχε μόνο δύο ημερών ακόμη ζωή. Τι είδου συντονισμό είναι αυτός. Εμείς χρειαζόμαστε θέλουμε να εμπνευστούμε από μια τόσο πρωτοποριακή ενωσιακός χώρα όπως η δική σας. Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνησή σας για τη φορολόγηση των δοσοληψιών εφόσον γίνεται. Υπάρχει βέβαια το πρόβλημα των εσόδων μέσα στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας που θέλουν να μας επιβάλλουν. Εγώ εντυπωσιάζομαι γιατί από τότε που ιδρύθηκε η ομάδα εργασίας του Βαν Ρόμπουι τον Μάιο του 2010 δεν έγινε λόγος για, έσοδα, Ενώ εσείς είπατε αν κάνουμε φορολογική μεταρρύθμιση ε, στο Βέλγιο οι γείτονέ μας εδώ 30 χιλιόμετρα παρακάτω μπορεί να κάνουν με την καταστάσει. Στη δική μου χώρα οι μετεγκαταστάσεις γίνονται προς εσάς μάλλον βέβαια. Τι θα γίνει λοιπόν για τα έσοδα. Έγινε λόγος για την Ελλάδα, Αλλά Δεν είμαι βέβαιο ότι είναι η μόνη χώρα όπου αν θέλουμε να υπάρξει διόρθωση των δημοσιονομικών πρέπει να ενδιαφερθούμε και για τη φοροδιαφυγή. Άρα να μιλήσουμε για κάποιο είδους φορολογική εναρμόνιση για να μην υπάρχει φορολογικό dumping. Τι φρονείτε. Για το πρώτο σας ερώτημα Ερωτώ και εγώ. Θεωρούμε ότι η δουλειά της Κομισιόν είναι να δίνει συμβουλές στις κυβερνήσεις ή μάλλον να περιγράφει αντικειμενικά την κατάσταση κάνοντας συστάσεις ανά χώρα ακριβώς. Είναι πολλές οι κυβερνήσεις που λένε στην Κομισιόν, εσείς λέτε αυτά που λέτε αλλά οι άλλοι φταίνε γιατί εμείς είμαστε καινούργια κυβέρνηση και φταίνε οι προηγούμενοι. Το καταλαβαίνω αυτό πολιτικά, αλλά και καταλαβαίνω ότι για την κοινή γνώμη πρέπει να μιλήσουμε και για τις επιλογές που έκαναν οι προηγούμενοι, για τις καλύτερες επιλογές που θα κάνουν οι επόμενοι, αλλά πώς να, πώς να κάνει μια αξιολόγηση η Κομισιόν ηθική λέγοντας έκαναν λάθος οι προηγούμενοι και γι' αυτό θα σας δώσουμε περισσότερο χρόνο και λοιπά. Όχι, μια κομισιόν δεν μπορεί να είναι αντικειμενική παρά μόνο εάν κάνει συστάσεις country specific. Country specific το ξαναλέω. Όταν ήμουν υπουργό εξωτερικών πήγα στο Πεκίνο και εξήγησα ότι μετά από δύο χρόνια ενασχόλησης με τα εξωτερικά ήμουν μεταξύ των 27 Ευρωπαίων Υπουργών δέκατος από αρχαιότητα μετά από δύο χρόνια. Ζούμε άρα σε ένα κόσμο όπου γίνονται πολλές εκλογές και εναλλάσσονται οι Υπουργοί. Συχνά. Δεν μπορεί μια πολιτική να καθορίζεται με βάση την κάθε κυβέρνηση. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος παρά να θεωρήσουμε ότι οι συστάσεις και οι συμβουλές είναι country specific. Όχι για κάθε κυβέρνηση, αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Ακόμη και αν φταίει κάποιο παρελθόν. Δεύτερο ερώτημα. Η θέση μας για τους ίδιους πόρους. Ξέρετε τη βολονταριστική θέση της κυβέρνησής μου. Ας πούμε τη φορολόγηση των δοσοληψιών Πρέπει να τη συνδυάσουμε όμως και με τη μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων ως προς το γιατί η Κομισιόν πρότεινε τα 2 τρίτα, 1 τρίτο, αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα μεν διανοητικά, αλλά καταρχήν πρέπει να δούμε τι επιτρέπει Uberhaupt, για να το πω γερμανικά, να εφαρμοστεί αυτός ο φόρος και σχεδόν ομόφωνα πρέπει, σχεδόν όλες οι χώρες πρέπει να ε, τον εφαρμόσουν. Άλλο αυτό από το πώς θα κατανεμηθούν τα έσοδα από το φόρο αυτόν όταν θα εφαρμοστεί. Η Λέα. Λοιπόν. Όχι, ο Ερωτώ για τους αριθμούς που βάλατε στη σελίδα 2 του εγγράφου που μας δώσατε. Α, δεν είναι δικό σας, α, καλά, τέλος πάντων, γνωρίζετε τους αριθμούς αυτούς. Είναι οι προβλέψεις ανάπτυξης για το 13. Εκεί λέει ότι οι προβλέψεις για το Βέλγιο της Κομισιόν είναι 1,2% και οι δικές σας 1,3%. Όταν όμως βλέπουμε τα ελλείμματα που προβλέπονται διαπιστώνουμε ότι μείον 2,3 λέει η Κομισιόν, άρα δεν είστε εντάξει ούτε εσείς, ενώ εσείς λέτε μείον 1,1. Ερωτώ λοιπόν πώς εξηγείτε τις διαφορές αυτές. Πάνω από ένα, μία ποσοστιαία μονάδα για το ίδιο μέγεθος είναι κάτι που θέτει το πρόβλημα της μεθόδου υπολογισμού θεωρείτε ότι η Κομισιόν έχει αξιόπιστα στοιχεία από ό,τι είπατε, ε, τότε τους αριθμούς της Κομισιόν θα πιστέψουμε και εμείς. Και άρα, αν υπάρχει έλλειμμα μείον 1,3, που μάλλον θα είναι και υψηλότερο, γιατί ολόκληρη η Ευρωζώνη βρίσκεται σε ύφεση και όλες οι προβλέψεις μειώνονται, θα υπάρξει μεγαλύτερο έλλειμμα και ερωτώ το εξής πολιτικά. θα ακολουθήσετε τους Ιταλούς μας φίλους που προτείνουν επαναδιαπραγμάτευση τουλάχιστον για το χρονοδιάγραμμα εκτός αν ληφθούν νέα μέτρα λιτότητας που όμως θα μειώσουν την ανάπτυξη ή μήπως θα παραμείνετε σε μια θέση που θα επιμένει στο 3% το 13% και επομένως τότε τι μέτρα λιτότητα θα λάβετε, λιτότητας θα λάβετε, θα κόψετε δαπάνες και ποιες, μειώνοντας πάλι την ανάπτυξη ή θα αυξήσετε τα έσοδα και άρα τους άμεσους φόρους επομένως το ΦΠΑ. Μήπως τότε όμως πάλι μειωθεί η ανάπτυξη γιατί ο ΦΠΑ αφορά άμεσα την κατανάλωση. Ευχαριστώ. Καταρχήν αυτό το έγγραφο δεν είναι δικό μας. Είναι των υπηρεσιών σας εδώ. Ήδη σας είπα ότι για το 11 υπάρχει κάποιο λάθος στο έγγραφο αυτό. Το έλλειμμά μας ήταν 3,7% και όχι 4,2% όπως λέει εδώ. Αυτό εξηγεί ήδη εν μέρη τη λογική μας, γιατί αν συγκρίνετε τους λεγόμενους βελγικούς αριθμούς και τους αριθμούς της Κομισιόν, Ξε, θα δείτε ότι οι αριθμοί και του Δουνουτού είναι σαν του Βελγίου και του ΩΣΑ. Σήμερα οι υπηρεσίες της Κομισιόν, που τις σέβομαι ιδιαίτερως και το λέω αυτό χωρίς καμιά ηρωνία, αντιμετωπίζουν μια κατάσταση όπου αν πούν στο Βέλγιο θα ξεπεράσετε το 3% διστάζουν να το κάνουν και άρα επί των συνολικών ποσών που υποβάλλουμε ως ρεαλιστικά ποσά θέτουν κάποια αμφιβολία αλλά βλέπουμε σιγά σιγά ότι είμαστε όντως σε θέση να εφαρμόσουμε αυτά που λέμε και σας το λέω ειλικρινά και σαφώς. Το 2013 θα έχουμε έλλειμμα 2,15%. Τελεία. Να το πείτε όπου θέλετε αν ξαναειδωθούμε μέσα στο 14 θα δείτε ότι θα το έχουμε εφαρμόσει. Και οι αριθμοί της Κομισιόν βασίζονται σε μια λογική μάλλον διαπραγματευτική μεταξύ υπηρεσιών. Η καταπολέμηση παραδείγματος χάρη της φοροδιαφυγής και των απατών αναφέρει αρκετά ψηλά ποσά, 700 εκατομμύρια ας πούμε. Και είναι φυσικό μια κομισιόν που έχει διαπιστώσει επανειλημμένως ότι οι κυβερνήσεις ζητούσαν όλο και περισσότερα και τα έγραφαν αυτά ως καταπολέμηση της απάτης, αυτό θα έκανε. Αλλά σας εγγυώμαι ότι στη χώρα μου πέρασαν πολλά νομοσχέδια που έχουν πραγματική επίπτωση και διορθώνουν τα πράγματα. The proof will be in the pudding. Αλλά μπορείτε να ρωτήσετε και το ανάλογο. Γιατί λέει τους αριθμούς αυτούς το δουνού του. Το ίδιο ερώτημα τίθεται. Θα δείτε όμως σιγά σιγά ότι τα κάνουμε όσα λέμε. Αξάλλου και για το 11 μέχρι το τέλος είχαμε αριθμούς που προέβλεπαν 4,2% έλλειμμα και στην πραγματικότητα ήταν 3,7 μισό της εκατό λιγότερο. Και αυτό είναι σίγουρο, δεν ήταν πρόβλεψη. Είναι αποτέλεσμα. Η Κομισιόν βάζει τους αριθμούς αυτούς για να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να αντιδράσουν. Φαίνεται ότι θέλει να διευκρινίσει τις θέσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα στοιχεία. Πολύ σύντομα όμως, ε, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ που με αφήνετε να μιλήσω. Θα είμαι πολύ σύντομος και ακριβής επί τεχνικών σημείων. Όταν δείτε τις προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλάμε για το μέχρι το 2013, Υπάρχει μεγάλη τεχνική απόκληση μεταξύ των προβλέψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των δικών μας. Εμείς εφαρμόζουμε το σενάριο μη αλληλεγγύη πολιτικών. Δηλαδή, ένα κομμάτι της απόκλησης οφείλεται, όπως είπε και την πρώτη κυβερνήσεως, στη διαφορετική αντίληψη των σύλληψη των μέτρων. Μεγάλη διαφορά οφείλεται στο ότι λαμβάνουμε υπόψη ότι θα υπάρξει προπολογισμό. Δεν προδικάζουμε. Προβλέπουμε το έλλειμμα σαν να συνεχίζεται προβάλλοντας το μέλλον την οικονομία. Όλοι ξέρουν βέβαια ότι καταρτίζεται ένα προπολογισμό, θα υπάρχουν εξελίξει κλπ. Διαβάζοντα τι προβλέψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επόμενα χρόνια, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θεωρούμε ότι θα, θα είναι 3,3 το έλλειμμα. Λέμε ότι με τα σχέδια μέτρα θα είναι 3,3, αλλά περιμένουμε και προπολογισμό. Και η απόκληση θα είναι πολύ μικρότερη. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο προβλέπει κανονιστικά σενάρια. Φαντάζονται ποιο θα είναι ο προπολογισμό και γι' αυτό τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ πιο κοντινά. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσάς είναι μια προβολή, μια πορεία που αγνοεί βήματα τα οποία ήδη να έχουν δρομολογηθεί. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να καταστεί σαφέστερο. Εν πάση περιπτώσει σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας. Νομίζω ότι είστε η δεύτερη χώρα που επέλεξε να έρθει και να μιλήσει στην Επιτροπή μας. Πέρα βέβαια από την υποχρέωση της ε, Προεδρίας να παρίσταται. Ε, βρίσκεται να εξελίξει η διαδικασία, αλλά είναι χρησιμότατη και θα ε, αυξάνεται σε σημαντικότητα, σε σημασία και έτσι θα σταθούν όλοι οι πίεση ούτω ώστε να λειτουργήσει η οικονομική διακυβέρνηση και το ευρωπαϊκό εξάμεινο για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα πριν συμβούν και να μην πρέπει να καταφεύγουμε σε κάποια πιο δρακόντια μέτρα που είναι διαθέσιμα όταν τα πράγματα πήγαινουν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. We Θα κάνουμε σύντομο διάλειμμα για να αποχωρήσει καταρχήν ο κύριος Υπουργός. Okay, thank you everybody. I think we can... Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Just like to now go back to the... Ας επιστρέψουμε στις ανακοινώσεις της Προέδρου και το ανυπόθηκα δάνεια, τα στεστικά δάνεια, το ΚΑΡΠ και τη σχετική οδηγία. Right, so, so Έγινε ψηφορία την περασμένη εβδομάδα. Αντολίν Σάντσε Πρεζέιδο, ο εισηγητή, είπε ότι θέλει να ξεκινήσει τριμερεί διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Σύμφωνα με τη συνηθισμένη διαδικασία, η διαπραγματευτική εντολή θα είναι η ψηφιστήσα έκθεση και η διαπραγματευτική ομάδα θα αποτελείται από, τους, από τον πρόεδρο εισηγητή και σκιώδης εισηγητές. Και ο εισηγητής της ΣΥΜΚΟ θα παρίσταται στον τριμερή διάλογο. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, τότε οι διαπραγματεύσεις θα ακολουθήσουν αυτή την πορεία από αυτής της βάσης. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, ο εισηγητής παρίσταται. Συμφωνούν όλοι. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Ούτως θα γίνει. Ευχαριστώ, Αντολή. Μπορούμε να πάμε στο 2-4. Σκοπιμότητα της εισαγωγής ομολόγου σταθερότητας. Η συγγήτρια είναι η Γκουλά, η οποία θα παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης. Σιλβή, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους. Είμαι ικανοποιημένη που μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα σήμερα, παρόλο που είναι ένα θέμα το οποίο ήδη μας απασχόλησε στο Six Pack και αποτέλεσε αντικείμενο ψηφίσματος που ψηφίστηκε στην Ολομέρεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου στις 15 περασμένου Φεβρουαρίου. Σε αυτή την έκθεση αισθάνομαι υποχρεωμένη να ακολουθήσω μια πορεία πάρα πολύ ακριβή μεταξύ των δύο, που των δύο υπερβολέων που χαρακτηρίζουν τη συζήτηση. Από τη μία πλευρά υπάρχει και επικίνδυνη θέση εκείνων παρουσιάζουν τα ευρωομόλογα σαν πανάκια, ένα είδος πανάκιας και ένα μέσο να απελευθερωθούμε από τις μεταρρυθμίσεις και τους περιορισμούς που φαίνονται επαχθείς. Δεν είναι ο καλός τρόπος να παρουσιαστούν αυτά τα μέσα. Δεν υπάρχει ένα φάρμακο θαυματουργό που θα αποφύγει την εξέταση των δημοσιονομικών ή να εξετάσουμε την κατάσταση των οικονομιών. Αντιστρόφως, θα ήταν υπερβολικό να αποκλείσουμε σαΐ e, κάθε μορφή κοινή αντιμετώπιση του χρέους στο βαθμό που κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αντιστοιχεί ε, σε κάποιους καλούς λόγους για να ακολουθεί σαν προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα, κατά την άποψή μου, Είμαστε υπέρ και η μεγάλη πλειοψηφία του ψήφου στο Κοινοβούλιο στο να παραμείνει η δημοσιονομική πειθαρχία. Και αυτή εδράζεται επί της ύπαρξης αγορών ρευστών. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το επίπεδο κάθε χώρα, αλλά αντικατοπτρίζεται η επίδοση κάθε χώρα. Όμω, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι αγορέ δεν εξασφαλίζουν τέλεια λειτουργία και μεταξύ κρατών της Ευρωζώνης υπάρχει διαφορά που δικαιολογείται εν μέρη από τις επιδόσεις που είναι διαφορετικές και θα πρέπει να παραμείνουν για να υπάρχει και μια, ένα κίνητρο για να παραμείνει η πειθαρχία. Υπάρχει όμως και μια υπερβολική πτυτικότητα που ίσως οδηγήσει χώρες που κάνουν δύσκολες μεταρρυθμίσεις να βρεθούν σταδιακά σε θέση να μην μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τις αγορές. Οι επενδυτές απ' την άλλη το βλέπουμε όταν συζητάμε με του ασφαλιστέ και αυτού που χειρίζονται τα συνταξιωτικά ταμεία και διαχειρίζονται τι αποταμιεύσει μα, χρειάζονται όλοι αυτοί ένα ρευστό, ευέλικτο εργαλείο που είναι ασφαλέ. Να μην είναι πολύ επικίνδυνο, αλλά να του δίνει επαρκέ κέρδο για να ε, εξυπηρετούνται τα κέρδη που πρέπει να έχουν και να πληρούνται και τα ασφάλιστρα. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που τις έχουν ανατεθεί και να μην μπει σε χώρους ξένους. Διότι μπορεί να χρειαστεί να καλύψει τα κενά και τις ελλείψεις ε, του πολιτικού τομέα. Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε. Κυρίως όταν βλέπουμε μείωση των επενδύσεων και εξυπηρέτηση των εθνικών των κρατικών χρεών. Βλέπουμε μία αποδόμηση εσωτερικής αγοράς που δεν είναι κάτι ευκταίο και δεν ταιριάζει με αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Εγώ επιμένω και το έγραψα στην έκθεση ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού το χρέο, αλλά δεν μπορούμε να το εξετάσουμε ελαφρά την καρδία αυτό. Δεν είναι εύκολη απόφαση. Θα βαρύνει κάποιε χώρε. Θα δημιουργηθούν ιδιαίτεροι περιορισμοί και υποχρεώσει. Όπω στη Γερμανία, Φιλανδοί, Ολλανδοί, Αυστριακοί, Γάλλοι ε, έχουν δισταγμούς για αυτό το λόγο. Αντιστρόφως, στο βαθμό που θα μπορούσαμε να περιορίσουμε τα ιδεολογικά προβλήματα, θα πρέπει να στερηθούμε αυτό το εργαλείο. Γι' αυτό προσπάθησα να ετοιμάσω ένα είδος φιλοπορίας, οδικό χάρτη, που καθησυχάζει εκείνους που λένε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια. Πράγματι, το άρθρο 125 συνθήκη μπορεί να υπάρχουν νομικά εμπόδια σε κάποιε σε κάποιες χώρε μέλη. Πήγα και σε ένα σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Humboldt με συνδυματολόγου Γερμανού, με τον καθηγήρα Μπαμάς και άλλους ε, να δούμε ποια είναι τα εμπόδια τα οποία προβάλλονται στη συζήτηση στη Γερμανία. Αντιστρόφως δεν νομίζω ότι οι Γερμανοί φίλοι μας θα πρέπει να αγνοούν ότι αν δεν βρούμε λύσεις μικρότερου εύρους θα έλεγα αλλά πιο άμεσα μέτρα ότι μπορούν να υπάρξουν δυσκολίες που θα συνεπέφεραν ε, συνέπειες για όλη την Ευρωζώνη. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν δύο είδη λύσεων που έχουν τεθεί επιτάπητος, υπάρχουν και άλλε λύσει, αλλά έχω διαλέξει δύο. Πρώτη λύση είναι του Ταμείου διάσωση Redemption Fund, ένα ταμείο απόσβεση του χρέους, που επιτρέπει κοινή αντιμετώπιση του χρέους, αλλά χρονικά περιορισμένα και στο χώρο περιορισμένα, διότι ο στόχος αυτού του Ταμείου Σωτηρίας είναι να εξαφανιστεί το χρέος. Εξορισμού λοιπόν Στόχος είναι η εξαφάνιση, η εξάλληψη του χρέους. Δίνουμε εχέγγυα για να εξαφανιστεί το, ε, το υπερβάλλον χρέος πάνω το 60% του ΕΠ. Η Οικονομική Επιτροπή ψήφισε δημιουργία του ταμείου αυτού, ψηφίστηκε στην Ολομέλεια, το ΤΟΥΠΑΚ. Είναι μία από τις λύσεις που ακολουθεί μία λύση με πάρα πολύ μεγάλους περιορισμούς για τις χώρες που θα συμμετάσχουν όσον αφορά τις εγγυήσεις όσον αφορά την διάθεση κάποιων εθνικών φορολογικών εσόδων και μια άλλη ριζικά διαφορετική λύση είναι τα ευρωμόλογα ε, πολύ βραχυπρόθεσμα το χρέος, το βάζουμε σε ένα σύστημα που μπορεί να ανακληθεί και αντίθετα την πρώτη λύση που έχει σαν στόχο να βρούμε μια λύση με ορίζοντα 20-25 χρόνια, εδώ έχουμε πιο κοντινό χρονικό περιθώριο, πολύ κοντά και θέλουμε ρευστότητα στις αγορές να πετύχουμε μέσω του Eurobills. Ε, εγώ δεν αποφάσισα, θεώρησα ότι πρέπει να το συζητήσουμε μαζί, διότι αυτές είναι λογικές που δεν αποκλείουν η μία την άλλη και οι δύο λύσεις, και το λέω ειλικρινά, έχουν και τα συν και τα πλήν. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει το θετικό ότι δίνουμε στην αγορά το μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μαζί κάποια πράγματα με ένα χρονικό όριο 20-25 χρόνια που δείχνει ότι διαρκεί η Ευρωζώνη και, και αυτό έχει κάποια ωφέλη και δεσμεύονται κάποιες χώρες να ρυθμίσουν πραγματικά το πρόβλημα του χρέους. Από την άλλη πλευρά, με την άλλη λύση, έχουμε τα αντίθετα ωφέλη. Κινούμε θα βραχυπρόθεσμα με ό,τι συνεπάγεται αυτόν την δυνατότητα αντιστροφής της πορείας ε, μπορούμε να καθισκάσουμε αυτού που θέλουν να δεσμευτούν υπερβολικά, αλλά δίνουμε στην αγορά μόνο την εγγύηση ότι υπάρχει κοινή αντιμετώπιση σε πολύ βραχυπρόθεσμη ε, πορεία. Αυτά είναι τα υπέρ και τα κατά των δύο λύσεων. Αυτό που θεωρώ σημαντικότατο και επιμένω από αυτού είναι να καταλάβετε ότι δεν μπορούμε να μην δώσουμε σήμερα λύσεις σε χώρες που για μία ακόμη φορά δεσμεύονται σοβαρά να κάνουν μεταρρυθμίσεις για κάποιες αυτέ τι χώρες ε, κάνουν θεσμικέ καινοτομίε όπως η Ιταλία όπου έχει μια τεχνοκρατική κυβέρνηση αλλά και αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία οι σχέσεις μεταξύ περιφερειών και κεντρικού κράτους και κυβέρνηση. κυβέρνησης κάποιες χώρες Ευρωζώνης με σοβαρότητα αλλάζουν συμπεριφορά και είναι σημαντικό να συνοδευτούν αυτέ οι διαδικασίε και να δούμε ε, κατά, εάν δεν μπορούν να είναι να μην δημιουργηθεί αστάθεια αν αποτύχουν αυτές τις που θα κάνει να υποφέρουν και οι χώρε του Βορρά και του Νότου. Βραχυπρόθεσμα υπάρχουν εμεί λύσεις που τι ανέφερα ακροαθυγώς στην έκθεσή μου προ υπόμνηση, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί το FSF ή το SM που θα πρέπει να τεθεί ισχύ σύντομα. Βέβαια αυτές οι δομές μπορούν να χρησιμεύσουν ε, για κοινή αντιμετώπιση. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο ούτε για αυτά τα ομόλογα σταθερότητα ούτε για το Ταμείο Σωτηρίας από πληρωμή του χρέους. Χρειάζεται μια ευθύνη ε, υπεύθυνη αντιμετώπιση που επεδείχθη από το Κοινοβούλιο και να το δείξουμε. Δεύτερη δυνατότητα ε, είναι η πρόταση από την οποία ξεκινήσαμε. Blue Bond τον, του Μαΐου του 2010. Το Ταμείο Διάσωσης είναι παιδί του Blue Bond που αντέστρεψε τη λογική. Στην πρόταση Blue Bond, υπενθυμίζω, επρόκειτο περί κοινής αντιμετώπισης του χρέους κάτω από το 60%. Δύσκολο να συνδυάσουμε το πάνω από το 60% και κάτω από το 60% και να πούμε ότι αντιμετωπίσαμε από κοινό το χρέο. Υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν μου ξέφυγε. Όμω, ήθελα να πω για εκείνου που το ανέφεραν, ο κ. Βαντσέικερ και ο Ζαν Πλάτ, ε, που επεξεργάστηκαν κάποιε ιδέε και νομίζω ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια καινοτόμα λύση στον οδικό χάρτη. Αν θέλουμε να φτάσουμε πραγματικά σε κοινή αντιμετώπιση του χρέου. χρειάζεται να κάνουμε ένα βήμα. Τροποποίηση των συνθήκων, πιθανότατα. Δεν θα έπρεπε να το απαγορεύσω σε αυτού μου. Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται να προετοιμαστεί προσεκτικά και γι' αυτό έθεσα αυτή την ιδέα που σα υποβάλλω. Ο κ. Λάγκεν ησυχάζει το γεγονό ότι ότι επιμένω ότι είναι ένα βήμα που δεν μπορούμε να το κάνουμε εύκολα και το λέω αυτό. Και κάποια εποχή δεν θεωρήσαμε ότι ήταν δυνατόν και το νέο νόμισμα και αυτό μπορούμε να το εξεργαστούμε παρόμοιως. Γιατί έφτασα λοιπόν σε αυτό το θέμα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να μελετήσουμε ε, που μπα καταλήξουμε. Η Επιτροπή Ντελόρ είχε επιτρέψει τότε να εργαστούν εκπρόσωποι των κρατών μελών με ένα είδος γραμματείας που εκαλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τότε, και το επενθυμίζω για εκείνους που το έχουν λησμονήσει, ήταν οι εθνικέ κεντρικέ τράπεζε που έπαιξαν το ρόλο του. Βεβαίω, θα έπρεπε αυτή τη φορά να εργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έχει δημιουργηθεί πλέον και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που ήθελα να πω ότι πρόκειται για περισσοβαρού βήματος, άρα χρειάζεται τεχνική ανάλυση βάθο χωρίς να χάνουμε όμως και την πολιτική διάσταση και αυτό ταιριάζει βέβαια και με τη δημιουργία ενός ταμείου ευρωπαϊκού και θα πρέπει αυτό το κέντρο αποφάσεων σε εμβριονική μορφή κάπως να πλαισιωθεί σωστά. Δεν μπορούμε αύριο να κάνουμε το βήμα, γιατί είναι πολύ δύσκολο βήμα. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις. Ο Μάριο Ντράγκη το ζήτησε σε αυτό το βήμα. Στα πλαίσια μεσοπρόθεσμου οράματος, η ομάδα εργασίας είπε όπου ο κ. Μπαρός, ο κ. Γιούνκερ, ο κ. Ντράκη, ο κ. Βαν Ροπόη συζητούν. Μήπως θα μπορούσε να επιληφθεί και τη πολιτική ενώσεω, τη δημοσιονομική ενώσεω. Είναι αόριστοι όροι που δεν σημαίνουν πολλά οι πολίτες αυτοί και είμαι επιφυλακτική σε αυτή τη χρήση. Θα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση και ξεκινάει κατά πρωτοβουλία τη Γερμανία τη Καγκελαρία και ίσω η όλη προσέγγιση χρειάζεται πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Και κλείνω εδώ Ήθελα να δείξω κυρία Πρόεδρε ότι μέχρι τώρα στην Ευρώπη υπάρχει μια τάση να γίνεται λόγος για κοινή αντιμετώπιση του εθνικού χρέους αντίθετο με αυτό που έγινε σε ένα σύνολο που έκανε βήματα πριν από φτάσει οι Αμερικής. Αν δούμε τι έκανε οι Πολιτείες τέλος του 18ου αιώνα, βλέπουμε ότι οι Πολιτείες έκαναν επιλογή εντελώς διαφορετική και θεώρησε ότι είναι χρήσιμο να υπενθυμίσω. Να μην παρέμβουν οι πολιτείες, η, πολιτική στις άλλες. Δεν ασχολείται η, Καλιφόρνια, η Φλόριδα με αυτά που κάνει η Καλιφόρνια. Η, δεν γίνεται έλεγχο τη Νεμπράσκα όσον αφορά τη διαχείριση. Δεν, ανα, δεν ανακατεύεται η Νεμπράσκα σε αυτά που κάνει το Κάνσα. Στη, ΣΥΠΑ έχουμε πολιτείε που ε, είναι υπεύθυνε για τον προπολογισμό του. Έχουμε χώρες που ε, έχουμε πολιτείες που δεν έχουν βοηθηθεί, ε, υπάρχει φεντεραλισμός προχωρημένος εκεί, αλλά σέβεται και την ελευθερία κάθε πολιτείας, κάθε φορέα που δημιουργεί την ε, Ομοσπονδία, που αποτελεί την Ομοσπονδία. Στην Ευρώπη φοβούμε ότι ενώματι ονόματι της αρνήσεως του φεντεραλισμού πάμε σε ένα πάρα πολύ πιο παρεμβατικό σύστημα από αυτά που έχουν τα ομοσπονδιακά κράτη. Οι Αμερικανοί λοιπόν αυτό που έκαναν μετά το 18ο αιώνα έκαναν ομοσπονδιακό προπολογισμό επιβάλλοντα ε, ομοσπονδιακού φόρου. Δεν ξέρω αν αύριο το πρωί πρέπει να κάνουμε το βήμα. Αυτό που είμαι υποχρεωμένη να κάνω στην έκθεσή μου είναι να εντοπίσω διανοητικά, θεωρητικά, τα διάφορα είδη λύσεων που προσφέρονται, μας προσφέρονται και να δείξω τα υπέρ και τα κατά κάθε λύσης. Ευχαριστώ τους σκιώδες συζητητές με τους οποίους είχα επικοδομητικές επαφές Έγινε υπευθύνη μου η έκθεση, αλλά υπήρξαν άκρως ενδιαφέρουσες συνομιλίες και επαφές μεταξύ μας. Υπάρχει αυτή η κοινή μέρημνα όλων. Να λάβουμε υπόψη τους δισταγμούς δικαιολογημένου κάποιων χωρών που καλούνται περισσότερο από άλλε από ό,τι φαίνεται, αν υπάρχουν κοινέ εγγυήσει να συμμετάσχουν, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Ευρωζώνη περνά μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και αν θέλουμε να συνεχίσουμε να κινούμεθα μεσοπρόθεσμα, να κινούμεθα μαζί, θα πρέπει ραχυπρόθεσμα να βρούμε λύσεις για χώρες ε, που έχουν σοβαρά προβλήματα. Είμαι ανοιχτή για συζήτηση και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε στην έγκριση ενός κειμένου που θα μπορούσε να δώσει κίνητο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο να κάνουν κάτι. Ευχαριστώ. Now... Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης τώρα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο Διέγκο. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω ε, για ε, την παρουσίαση και για το έργο της συνολικά. Και το επικοδομητικό πνεύμα με το οποίο προσεγγίζει όλα αυτά τα θέματα είναι διαφορετικές οι λύσεις που προσφέρονται εδώ, βραχή, μέσο και μακροπρόθεσμες. Και βέβαια το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει την πρόθεση να τα συζητήσει όλα αυτά εντατικά, αλλά έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα. Πρώτον, δημοσιονομική πειθαρχία. Δεύτερον, τα δημόσια οικονομικά θα πρέπει να είναι υγιή, ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί. Και τρίτον, να υπερασπιστούμε την έννοια της Δημοσιονομικής Ένωσης. Διότι μόνο εφόσον έχουμε εξυγίανση και υγιή οικονομικά παντού, με μεταρρυθμίσεις, τότε και μόνο τότε θα έχουμε ανάπτυξη βιώσιμη και αηφόρο και σταθερότητα σε τελική ανάλυση στην Ευρωζώνη. Για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με σοβαρότητα, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολιτικές προϋποθέσεις και οικονομικές σίγουρα. Δεν είναι μόνο τα δημόσια οικονομικά, αλλά είναι και ορισμένα νομικά ζητήματα σε σχέση με τις συνθήκες. Τώρα που θα συζητήσουμε αυτή την έκθεση, πρέπει να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο και την ίδια πορεία που είχαμε και στη δέσμη των έξι οδηγιών, το λεγόμενο six-pack, όπως και το two-pack πιο πρόσφατα. Θα θυμάστε ότι συμφωνήσαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει μελέτη και είχα ήδη την ευκαιρία να το συζητήσω αυτό με την εισηγήτρια. Δεν θέλω να επεκταθώ αυτή τη στιγμή γιατί πρέπει να μιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Θυμίζω ότι η κρίση είναι ευρωπαϊκή και το πρόβλημα. Δεν μπορεί να λυθεί σε επίπεδο ενός κράτους μέλους το πρόβλημα. Αυτά εισαγωγικά και πρέπει να πω ότι χαίρομαι και προσβλέπω στη συνεργασία με την εισηγήτρια. Και περιμένω να ακούσω και τη συζήτηση. Ε, ε, Ευχαριστώ. Εξ ονόματος του Σικλούνα Υπερβάνς να με βάλετε όμως στον κατάλογο και εξ ονόματός μου. Γιατί εγώ απλώς θα διαβάσω το έγγραφο του Σικλούνα. Μόνο θα το διαβάσω. Μάλιστα. Αγαπητοί Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να συγχαρώ την κυρία Κουλάρ για τη σκληρή εργασία της για την έκθεσή της. Ως κοιόδης σοσιαλιστής επί του θέματος Βρίσκομαι σε συμφωνία με πολλά από όσα έχει πει. Παρόλα αυτά υπάρχει και μια ανησυχία για μας που αφορά την παράγραφο 8 που φαίνεται να δηλώνει ότι χρειάζονται περισσότερα και ταχύτερα μέτρα λιτότητας. Αυτό θέλουμε να το διαγράψουμε. Όσο για την προσθήκη, έχουμε και εκεί ορισμένες αμφιβολίες για την χρονική πραγματοποίηση όλων αυτών, διότι αν κινηθούμε προς ένα σύστημα ευρωομολόγων, δεν πρέπει να ακολουθήσουμε το ίδιο χρονοδιάγραμμα με το υπάρχον. Όσο για το πώς θα λειτουργήσουν τα διασωστικά ταμεία, υπάρχουν ερωτήματα. Πώς θα μπορούσαμε να καταφέρουμε να συλλειτουργήσουν τα ευρωμόλογα με το Ταμείο Διάσωσης και τι σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να χρειαστεί αλλαγή των συνθήκων. Τα ευρωμόλογα δεν είναι τρόπος λύσης της τρέχουσας κρίσης, αλλά είναι ζωτικά αν θέλουμε να αποφύγουμε μια μελλοντική κρίση. Ένα από τα δομικά προβλήματα της Ευρωζώνης είναι ότι είναι τόσο δυνατή όσο πιο αδύνατος κρίκος της. Τα τελευταία δύο χρόνια το είδαμε ότι αυξήθηκε, υπερχρεώθηκαν οι πιο αδύνατες χώρες πέρα από το όριο που μπορούν να αντέξουν και υπέστησαν ύφεση που έπληξε και τις ε, στεναρότερες τράπεζες. Τα ευρωμόλογα μπορούν να λειτουργήσουν μόνο αν πρώτα λυθεί το πρόβλημα των ηθικών κινδύνων. Πρέπει να υπάρχουν κριτήρια και εισόδου και εξόδου. Η κρίση σε υπερβολικά πολύ και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι ηγέτες της Ένωσης δεν επέδειξαν τιμιότητα ως προς τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται. Εμείς πρέπει να δείξουμε το δρόμο. Τα ευρωμόλογα δεν είναι πανάκια αλλά θα είναι τμήμα του μέλλοντος της Ευρωζώνης. Μάλιστα. Άσλι. Στο πρόεδρε. Να πω δύο λόγια εξ ονόματος πρώτα του κυρίου Έπιγκ που είναι ο σκιώδης μας και μετά να πω και δύο δικά μου. Η ομάδα μου δεν είναι ευχαριστημένη με την έκθεση αυτή και την όλη ιδέα των ευρωομολόγων και ή των ομολόγων σταθερότητας. Και πριν προχωρήσω θα έλεγα ότι η ιδέα του Ταμείου Διάσωσης πρέπει πρώτα να αναλυθεί καλύτερα. Υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος, οι χώρες, οι λίγες χώρες που αυτή τη στιγμή έχουν ακόμα τριπλό αλφα να υποβαθμιστούν αν αναλάβουν περισσότερο χρέος και περισσότερο κίνδυνο. Και υπάρχει και το θέμα του ηθικού κινδύνου που έθιξε ο κύριος Κυκλούνα προηγουμένως. Τι κίνητρα υπάρχουν για να μειώσουν οι χώρες που βρίσκονται σε δυσκολία τις δαπάνες τους αν ξέρουν ότι θα δανειστούν πάλι από τη Γερμανία με την πιστοτική της κάρτα. Ο λόγος που υπάρχει κρίση είναι ότι πολλές χώρες δαπανούν υπερβολικά πολλά για πολύ χρόνο. Και βρίσκω εκπληκτικό ακόμη και τώρα ότι υπάρχουν πολιτικοί που λένε ότι ο τρόπος που θα, για να βγούμε από την κρίση είναι να δαπανίσουμε ακόμη περισσότερα. Αν υπάρξουν τα ευρωομόλογα ή ομόλογα σταθερότητα που θα τα εγγυηθούν η Ολλανδία και η Γερμανία, τότε λένε λύνονται όλα, θα δαπανίσουμε κι άλλα. Και δεν καταλαβαίνουν ότι ο λόγος που βρίσκονται σε αυτό το χάλι ο λόγος που η Ελλάδα έχει φαλυρίσει είναι γιατί για πολύ χρόνο δαπανούσε υπερβολικά πολλά. Και το μόνο πράγμα που δεν έθιξε η κυρία Γκουλάρ στην έκθεσή της είναι το θέμα του ενιαίου νομίσματος και του πώς δημιουργήθηκε. Έκανε ένα σχόλιο που σημείωσα, είπε δεν σκεφτόμασταν, παλιά δεν νομίζαμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει το ενιαίο νόμισμα Θεωρεί όμως ότι λειτουργεί. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ενιαίο νόμισμα αν δεν υπάρχει ένας και μόνο υπουργό Οικονομικών που να ελέγχει τις δαπάνες. Τώρα βλέπουμε ότι η κρίση στην Ελλάδα που επεκτάθηκε και στην Ισπανία και αλλού was badly put together. οφείλεται στο ότι κακώς έγινε η διοργάνωση του ευρώ. Αυτά είναι οι επιπτώσεις της κακής αυτής της οργάνωσης. Αν δεν το πούμε αυτό δεν βρίσκουμε λύση. Μου φαίνεται ότι αν θέλουμε να επιβιώσει το ενιαίο νόμισμα τότε είτε χρειάζονται πολύ μεγάλες φορολογικές μεταφορές από τις χώρες που έχουν πλεονάσματα όπως η Ολλανδία και η Γερμανία σε άλλες χώρες, πράγμα το οποίο θα γίνει μόνιμη κατάσταση, είτε Μερικές χώρες πρέπει να φύγουν από το Ευουρό. Και φαίνεται ότι αυτό το θέμα δεν έχει ακόμα συζητηθεί. Η γερμανική κυβέρνηση είπε ότι θέλει η Ελλάδα και οι άλλοι να μείνουν στο ευρώ. Αλλά δεν είναι διατεθειμένη να δώσει χρήματα που χρειάζονται για να παραμείνουν. Και υπάρχουν και οι πολιτικοί στην Ελλάδα και αλλού που λένε θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε τις απαραίτητες θυσίες. Αυτό είναι και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χαρτάτο. Στην έκθεσή σας λοιπόν γενικότερα η ομάδα μας είναι αντίθετη. Πρόκειται όντως για συμβιβασμό, αλλά δεν λύνει το βασικό πρόβλημα που είναι η δομή της ενιαία, του ενιαίου νομίσματος. Και ακόμα πολλοί πολιτικοί δεν είναι διατεθειμένοι να επιδείξουν το απαραίτητο θάρρος για να μιλήσουν είτε για τη διάλυση του ενιαίου νομίσματος είτε για μια κανονική δημοσιονομική ένωση. Οι χώρες της Ευρωζώνης έχουν αυτή την επιλογή και επειδή δεν επιλέγουν τίποτα δημιουργείται τέτοια αστάθεια. Ευχαριστώ, Ο Φίλιππος. Συμφωνώ με τον Άσλη αυτά που είπε στο τέλος τουλάχιστον. Πράγματι πρέπει να διαλέξουμε κάποιο δρόμο και επειδή δεν επιλέγουμε χειροτερεύει η κρίση. Εδώ συμφωνώ απόλυτα. Εκεί που διαφωνούμε είναι ποιο είναι ο δρόμο, ποιοι είναι οι δρόμοι. Εγώ νομίζω ότι η έκθεση δείχνει ένα δρόμο. Μία φράση του Τρισέ είναι ότι το μέλλον μας είναι αναφυσβήτητα κοινό. Δηλαδή κανείς από εμά δεν μπορεί να διασωθεί μόνος του και να αντιμετωπίσει όχι μόνο την κρίση αλλά και όλα τα προβλήματα του 21ου αιώνα. Είτε θα πετύχουμε όλοι μαζί είτε θα αποτύχουμε ένας ένας. Δεν υπάρχει λοιπόν λύση χωρίς δημοσιονομική ένωση. Και με αυτό εννοώ κοινού κανόνες, κοινού στόχους για τις δαπάνες. Αλλά ο προϋπολογισμός σημαίνει και δαπάνες και έσοδα. Άρα κανόνες κοινού και για τα έσοδα. Δεν μπορούμε να έχουμε συνεργασία για τις δαπάνες αλλά όχι για τα έσοδα. Και για το ένα και για το άλλο. Και αυτό συμπεριλαμβάνει τα ευρωμόλογα. Και κάποιον κοινό τρόπο να δούμε τι θα κάνουμε με, το, με τη λεγόμενη τραπεζική ένωση. Δηλαδή κοινή ανάληψη των δεσμεύσεων και των ρίσκων. Αυτά δεν γίνονται χωρίς πολιτική ένωση. Οι Αμερικανοί επαναστάτες έλεγαν ε, να μην υπάρχει φορολόγηση χωρίς εκπροσώπηση. Κάτι ήδη ανάλογο ισχύει και εδώ. Δεν μπορούμε να λάβουμε κοινούς δημοσιονομικούς στόχους χωρίς να έχουμε κοινέ πολιτικές αποφάσεις. Και για μένα οι εξτρεμιστές είναι αυτοί που λένε θέλουμε ένα από αυτά τα στοιχεία και όχι τα υπόλοιπα. Ας πούμε, θέλουμε να αναλάβουμε από κοινού το χρέος και όχι τα άλλα. Ή θέλουμε δημοσιονομική πειθαρχία κοινή, αλλά όχι τα υπόλοιπα. Αυτά νομίζω ότι είναι απάτη και λάθος διανοητικό καθώς και οικονομική ανοησία και άρνηση επιλογής. Γι' αυτό νομίζω ότι η έκθεσή σου δείχνει το σωστό δρόμο. Εκεί όπου έχω μια διαφορά είναι ο βαθμός κατά πόσον όλα αυτά είναι πήγοντα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα μέτρα, το σύνολο, όχι μερικά, ένα-ένα, είναι κάτι που μπορούμε να το αναβάλουμε παόριστον. Γιατί είναι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σύντομα. Ήδη τέσσερα χρόνια διαρκεί η κρίση. Πάντοτε αναβάλαμε την απόφαση και φοβάμαι ότι αν δεν έχουμε το θάρρος να την λάβουμε αυτή τη τολμηρή απόφαση τώρα και ελπίζω ότι η διάσκεψη της 28ης-29ου θα καταστήσει την εκθεσή σου αχρίαστη. Αν δεν το κάνουμε τώρα τότε ο αγώνας δρόμου για την καταστροφή της Ένωσης μπορεί να χαθεί. Συμφωνούμε με τα περισσότερα σημεία της έκθεσης. Υπάρχουν μερικές όπου θα προτιμούσαμε να γίνεται αναφορά σε κοινοτική νομοθεσία μάλλον παρά στο καινούριο δημοσιονομικό σύμφωνο δηλαδή σε ενωσιακή μάλλον παρά διακυβερνητική λογική. Και τελειώνω με δύο τελευταία σημεία για την ΑΣΛΕΙ και τη Σιλβή. Για σένα Σιλβή θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα να πάψουμε πλέον να λέμε ότι η ΕΚΤ πάντοτε βοηθούσε τα κράτη-μέλη που δεν είχαν το πολιτικό θάρρος να, αναλάβουν, να λάβουν τα μέτρα που έπρεπε. Καμιά φορά είναι σωστό, αλλά γενικά έχει τεράστια ευθύνη η ΕΚΤ για το ότι αναβλήθηκε και για δύο χρόνια η αναγνώριση ενός απλού γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να πληρώσει ήδη από το 2009. Και είναι το λάθος της ΕΚΤ που έλεγε ότι ένα κράτος της Ένωσης δεν μπορεί να απτοχεύσει. Διότι αυτό κατέστησε την επίλυση του ελληνικού προβλήματος βαρύτερη και για τους Έλληνες και για τους υπόλοιπους φορολογούμενους στην Ευρώπη. Η ΕΚΤ δεν έχει πάντα δίκιο λοιπόν, κάνει λάθη. Άσλι Φόξ. Βλέπω ότι φεύγει. Έχω βαρεθεί πλέον να ακούω να μιλάτε για ηθικολογίες για κυβερνήσεις ενώ δεν το λέτε για τράπεζες. Ωραίο είναι να λέτε «Α, ένα κράτος δεν επέδειξε την απαραίτητη πειθαρχία και χρησιμοποιεί τα λεφτά των άλλων», αλλά το ίδιο είναι κύριε Άσλεϊ, το να λέμε ότι δεν είναι πρόβλημα να συνεχίζουν οι τράπεζες να υπερδανίζουν και αυτοί αυτό κάνουν. Αν θέλετε να είστε σοβαρός λοιπόν για τους λεγόμενους ηθικούς κινδύνους πρέπει να το λέτε και για τα κράτη και για τις τράπεζες. Όχι να λέμε ναι ναι να προσέχουμε και τα λοιπά. Το ειδικό χρέος δεν είναι πρόβλημα μόνο το δημόσιο. Ω και τα δύο είναι. Και Επομένως δεν είναι όλα αυτά που είπατε και τόσο αδιαμφισβήτητα. Φαντάζομαι ότι εύκολα θα συμφωνήσουμε με τη Σιλβή και ελπίζω ότι τα γεγονότα τελικά θα μας ξεπεράσουν. Ελπίζω να βρεθεί δηλαδή λύση πριν τελειώσει η συζήτηση του θέματος. Εντάξει, ευχαριστώ. Η Αρίσα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να πω κάτι για την έκθεση, αλλά και να σχολιάσω τα λεγόμενα του συναδελφού Φόξ. Τα ίδια ακούμε ξανά και ξανά στις χώρες που έχουν ελλείμματα. Και δεν είναι θετικά. Δεν βοηθούν ε, αυτές οι κατηγορίες. Η έκθεση είναι καλή και για τα ευρωομόλογα, τα είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη συνεδρίαση. Είναι ένα έγγραφο που μπορεί να αποτελέσει βάση εργασίας για να συζητούμε τέτοια σημαντικά θέματα. Υπάρχουν ορισμένα ανοιχτά ακόμα κρεμή ζητήματα, όπου πραγματικά πρέπει να γίνει πολιτική συζήτηση και να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Αυτά τα τρία πρέπει να τα απαντήσουμε αλλιώς θα εωρείται ένα κενό και δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε. Για τα λεγόμενα ομόλογα σταθερότητας. Δεν θα πρέπει να συζητούμε μηχανισμούς στήριξης χωρίς ε, να συζητούμε και αυτό το πρόβλημα, ε, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες. Γιατί το λέω αυτό. Αναφέρθηκαν κάποια προγράμματα προσαρμογής που δεν ήταν ουσιαστικά προσαρμογής και στη συνέχεια δόθηκε χρηματοδότηση που συνδέεται με προϋποθέσεις και όρους τρομερά κατασταλτικούς και ασφικτικούς και ήταν μοιραίο ότι ε, θα αποτύχαναν. Δηλαδή και αυτά τα χρήματα που πήραμε δεν μπορέσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε προς το σκοπό που έπρεπε. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Προφανώς πολλές χώρες έχουν πολλά οικονομικά προβλήματα, αλλά όταν μιλάμε για προσαρμογές πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις ιδιαιτερότητες αυτές για χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία. Αν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα δεν βοηθάει μόνο η αποταμίευση και οι περικοπές και οι οικονομίες. Χρειάζεται ανάπτυξη οπωσδήποτε πέρα από τις ε, προσαρμογές. Δεύτερον, Καλή πρόταση, επαναλαμβάνω, ως έγγραφο και βάση εργασίας, αλλά τα ευρωομόλογα πρέπει να ε, εκδοθούν, λένε κάποιοι, αφού ξεπεραστεί η κρίση και έχουν λυθεί τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα δηλαδή. Ωραία. Έτσι κάπως ορίζεται και το Ταμείο Αποπληρωμής ή Απόσβησης. Ε, το χρησιμοποιούν χώρες που βρίσκονται σε προγράμματα προσαρμογής. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Είναι περιορισμός που σημαίνει στην πράξη ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν μπορούν να βοηθήσουν αυτές τις χώρες. πρέπει να δούμε τι ε, ρόλο θα δώσουμε εμείς στα ευρωομόλογα. Δεν είναι ανταμοιβή, δεν είναι επιβράβευση των χωρών που έκαναν ε, ωραία τα προγράμματα. Έχουμε πολλά αντίθετα και αρνητικά παραδείγματα και αποδείξεις για αυτά. Λοιπόν, αν δεν τα καταλάβουμε όλα αυτά, δεν θα βγάλουμε και τη σωστή διάγνωση για τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Και αυτή τη διάγνωση τη χρειαζόμαστε για να βρούμε και το σωστό φάρμακο. Έχει γίνει καλή δουλειά, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε συγκεκριμένα, αλλιώς δεν θα γίνει διάγνωση, θα είναι νεκροψία. Okay, thank you very much. the name. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Θα διαβάσω αυτούς που έχω στον κατάλογο. Astrid Lulling. Sanchez Prezedo, Provence Beres, Werner Langen, Peter Simon, and Sophie Intveld, and myself. Um, yes, well, he should go first, shouldn't he? Are you the shadow for your... Είστε ο σκιώδης για την ομάδα σας εσείς. What? Mr. Terre. Κύριε Τέρε. EFT, no. Ο κύριε Τόιρε. Θα σας βάλουμε και σας τον κατάλογο. Άλλος ουδή άλλου. Και η Άστριντ, έχει πρώτη το λόγο. Εκτό μικροφώνου. Μετά, μετά το Werner θέλεις πρώτο Werner Langen και μετά. Burg Weiß schon, was es an deutschem Geld hat. Ξέρει το Λουξεμβούργο τι σημαίνουν τα γερμανικά λεφτά. Έχουν γνώση φύλακε και η κυρία Λούλινγκ. Ναι, ναι, ναι. Οι Λουξεμβούργοι εδώ και χρόνια έπαιρναν ε, και υπέθαλπταν τα γερμανικά λεφτά που φοροδιέφευγαν. Αλλά τώρα υπάρχει και φορολόγηση της έδρας και στο Λουξεμβούργο. Οπότε το πρόβλημα άλλαξε και μειώθηκε κατά πολύ. Παρ' όλα αυτά το Λουξεμβούργο παραμένει ενδιαφέρον τραπεζικός τόπος, όχι μόνο από αυτά που μας λέει ε, ο Πρωθυπουργό, αλλά και η Άστρικ Λούλινγκ ε, επανειλημμένα. Λοιπόν, ανεξάρτητα από όλα αυτά, θέλω να πω εγώ κάτι τώρα πρώτα για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή τη λεγόμενη πράσινη βίβλο του Νοεμβρίου. Αρκεί να κοιτάξει κανείς τη σελίδα 24 για να διαπιστώσει ότι στις νομικές σκέψεις λέει ότι και οι τρεις ε, Προτάσει ενδεχομένω, στην πρώτη χρειάζονται αλλαγέ των συνθηκών, στη δεύτερη ενδεχομένω, επίση και στην τρίτη περί αυτού πρόκειται δεν χρειάζεται αλλαγή των συνθηκών, δεύτερογενέ ρυθμίσει νομοθετικέ. χρειάζονται. Αυτά είναι τελείω απαράδεκτα. Στο άρθρο 125 τη συνθήκη τι ορίζεται ρητά, ότι απαγορεύεται η συλλογική ανάληψη του χρέους. Μπορεί κανείς να φανταστεί εδώ μέσα ότι χωρίς αλλαγή των συνθήκων Μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα σε σημαντικό κράτη-μέλη. Να αναφέρω Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, ε, κάτω χώρες, Φινλανδία, Σουηδία, οι τρεις χώρες της Βαλτικής, Πολωνία, Τσεχία και πάει λέγοντας, εκεί ε, μπορούν να συμφωνήσουν σε ομόλογα τέτοια ε, κοινή ανάληψη του χρέους χωρίς μεταρρύθμιση των συνθήκων. Αυτό είναι σκέτη χήμερα. Ήδη η Επιτροπή το λέει. Γιατί δεν έλαμψε τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όταν έπρεπε να κάνει λογικές προτάσεις ε, για τη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης. Ο κύριος ο Ρόζος το πρώτο πακέτο για την Ελλάδα 10 Μαΐου του 10 ε, δεσμεύτηκε να δοθούν 60 δισεκατομμύρια από τον κοινοτικό προπολογισμό χωρίς να υπάρχει κονδύλι. Σύμφωνα με το άρθρο 122 της συνθήκης, αντιμετώπιση θεομηνιών τη βάφτισε. Άνευ προηγουμένου σκάνδαλο είναι αυτό. Το έχω πει πριν από δύο χρόνια αυτό. Και για το μηχανισμό σταθερότητας στον ευρωπαϊκό που δεν έχει ακόμα ψηφιστεί χρησιμοποιούμε το άρθρο και αλλάξαμε το άρθρο 136. Αυτό ήταν το ελάχιστο που χρειαζόταν. Και στο άρθρο 125 τώρα με μια πράσινη βίβλο να το καταργούμε και να μην συμπεριλαμβάνονται τα σημαντικότερα θέματα, αυτό είναι τελείως απαράδεκτο. Και έτσι προστίθεται τώρα το ένα στο άλλο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, σήμερα ε, αντιτάχθηκε σε αυτό, αλλά ο κύριος Λάμπρες, ε, μεγάλος ρήτορ, λέει ότι πράττει κατά το δοκούν. Είναι αξιοσημείωτη αυτή η δράση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ανεξάρτητη και μας μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να παραμένει ανεξάρτητη και σήμερα ε, απεφάνθη κατά του Ταμείου Απόσβεσης του Χρέους και τέτοιων ε, μορφών. Δεν ξέρω μήπως δεν τα έχουν καταλάβει αρκετά. Δεύτερον, δεν πρέπει να κάνουμε το δεύτερο βήμα πριν από το πρώτο. Κοινώς να μην προτρέχουμε. Το πρώτο είναι το δημοσιονομικό σύμφωνο, η εξυγίανση του προπολογισμού. Και επειδή τώρα η ελληνική πολιτική απέτυχε εκτρά, εγκάρσια. Όλα τα κόμματα έχουν ευθύνε τι τελευταίε δεκαετίε. Επειδή έγιναν όλα αυτά, θα πρέπει εμεί τώρα να παραβιάσουμε και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τι είναι οι συμπεράσματα αυτά άνευ προηγουμένου, ανήκουστα. Και ότι υπάρχουν ε, ε, δάνεια ε, ομοσπονδιακά στην Αμερική, ναι, εντάξει, αλλά κάθε πολιτεία ε, ευθύνεται για το ίδιο σου χρέος. Παραλίγο να χρεοκοπήσει η Νέα Υόρκη, παραλίγο να χρεοκοπήσει η Καλιφόρνια. Δεν αναλαμβάνει κανεί το χρέος, κάθε πολιτεία το δικό της. Και μετά μπορεί να έχουν ομόλογα. Το τρίτο, ομόλογα σταθερότητα. Πολύ ωραία έκφραση. Όπως στη Γερμανία όταν η οικονομία είχε ύφεση εφήβραν τον όρο μηδενική ανάπτυξη. Και τι είναι αυτά τώρα τα ομόλογα σταθερότητα προϋποθέτουν ότι τα κράτη-μέλη θα τηρήσουν τις συνθήκες. Δεν είναι νέες οι συνθήκες. Το 97 κυρώθηκαν και πολλοί τις κατήργησαν γιατί δεν τις τηρούσαν και μεταξύ αυτών και η Γερμανία και η Γαλλία. Οπότε δεν πιστεύω ότι πρέπει να πάμε τώρα στα ομόλογα έργων. Επενδύσεις υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτό μπορεί να είναι ένα βήμα ε, καλό, θετικό, πρώτο και δεν ε, παραβιάζει το έρθρο 125 περί μη ανάληψη χρέους. Λοιπόν, όλα αυτά μπορούμε να τα αεροποιούμε όπως θέλετε, αλλά γι' αυτό και εγώ και κάποιοι άλλοι κατά τη διάρκεια τη συζήτηση, θα ακούσετε ότι απορρίπτουμε το σχέδιο έκθεση Γκουλάρ, την οποία εκτιμώ και σέβομαι προσωπικά, αλλά εδώ νομίζω ε, έχει πάρει λάθος τον δρόμο και που οδηγεί αυτό το έδειξαν χτες ε, τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών. Ευχαριστώ. Ε, okay, now, Antolin. Sanchez Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια για την έκθεσή της μου φαίνεται πάρα πολύ απαραίτητη και αναγκαία. Τα τελευταία 50 χρόνια έχουμε δύο οράματα για την Ευρώπη. Μια Ευρώπη η ζώνη ελευθέρων συναλλαγών και μια Ευρώπη που είναι όλο και πιο τέλεια ένωση. Και αυτή τη στιγμή ισχύει μόνο η πρώτη, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ε, και για τα ευρωομόλογα προφανώς δεν είναι θέσφατο ούτε πανάκια ούτε τίποτα. Αλλά και επίσης δεν υπάρχει μια ενιαία αντίληψη για τα ευρωομόλογα μοναδική. Είναι πολύ σήμαντο. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ευρωομολόγων. Εμείς καλούμαστε να επιλέξουμε ανάμεσα σε ένα ρεπερτόριο που μπορεί να μας ε, λύσει προβλήματα και να έχει τις λιγότερες δυσκολίες. Εγώ νομίζω ότι το ενιαίο νόμισμα είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι εξωτερικό ε, νόμισμα για κάποιες χώρες κρίσης που δεν έχουν ίδιο νόμισμα, αλλά δεν θα πρέπει να είναι εξωτερικό συνάλλαγμα. Υπήρχαν προβλήματα στη διακυβέρνηση στην Ευρώπη, γιατί όταν έχουμε σύγκληση ε, σε 200 ε, μονάδες βάσης με τη χώρα που έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό και να είναι αυτή η σύγκληση, θα πρέπει να είναι και η σύγκληση και το μονοπάτι της σταθερότητας. Δεν είναι μόνο θέμα διακυβέρνηση όμω ορισμένων κρατών μελών. Γιατί αν τα προβλήματα ήταν δημοσιονομικού χαρακτήρα, των δημοσίων οικονομικών δηλαδή, θα βάρινε η απόφαση των κρατών μελών. Υπάρχουν και άλλα θέματα όμως για το πώς λειτουργεί η νομισματική πολιτική και οι αγορές και αυτό είναι συν ευθύνη. Οπότε αν η Ευρώπη είναι μέρος του προβλήματος θα πρέπει να είναι και μέρος της λύσης. Και αυτή η συζήτηση για τον ηθικό κίνδυνο, εντάξει υπάρχουν χώρες που έχουν σπαταλήσει πολλά, και αν ήταν δικά τους λεφτά είναι ηθικό κίνδυνο, αλλά και άλλες χώρες που έχουν δώσει πολλά χρήματα σε άλλες χώρες φέρουν ευθύνη επίση. Γιατί πρέπει κάθε φορά να αξιολογείται. Υπάρχουν οι οργανισμοί. Και τι γίνεται με το ιδιωτικό εξωτερικό χρέος, αν μπορεί να γίνει δημόσιο εσωτερικό χρέος. Είναι μια συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη θεμητή και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε κι εμείς. Έρχομαι στα ευρωομόλογα. Αυτό που έχει σημασία είναι ο σχεδιασμός. Πώς θα τα φτιάξουμε αυτά. Με ρεαλισμό που να λύνει προβλήματα χωρίς να δημιουργεί επιπλέον ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να σχεδιαστούν ακριβώς ε, γνωρίζοντας για ποιο στόχο θα χρησιμοποιηθούν. Όχι για την επόμενη κρίση. Ήδη από τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια υποφελή και θα φέρουν μεγαλύτερη ισορροπία, χρειαζόμαστε περισσότερο οικονομικό συντονισμό και ο οικονομικός συντονισμός δεν χρειάζεται μόνο κυρώσεις αλλά και ε, κίνητρα και ενθάρρυνση. Μπορεί να χρειάζεται να διορθώσουμε κάποιες λειτουργίες της αγοράς. Ορισμένες χώρες λαμβάνουν μέτρα και κάνουν μεταρρυθμίσεις διορθωτικές για να έχουν μακροπρόθεσμα ε, αποτέλεσμα, αλλά αυτό που χρειάζονται τώρα είναι ενίσχυση βράχη πρόθεσμα και θα πρέπει να επιβραβεύεται αυτή η προσπάθεια. Και τα ευρωομόλογα είναι σημαντικά για να υπάρχουν ομόλογα σε ευρώ και το ευρώ να είναι ένα νόμισμα που θα βαρύνει διεθνώ. Η έκθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ αναγκαία, πάρα πολύ επίκαιρη και εύστοχη και θα πρέπει όλοι να αγωνιστούμε για να επιτύχει. Thank you. Ευχαριστώ, υπερβάμωση έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα κατανομάσω κάποιους, αλλά να υπενθυμίσω στο Βέρνερ Λάγκεν ένα κείμενο που διαπραγματευτήκαμε σκληρά και συζητήσαμε και συντάξαμε μαζί μια έκθεση για την οποία ήμασταν και δύο υπεύθυνοι και όπου κανένα σημείο δεν εισήχθη κρυφά, όλα τα σημεία συζητήθηκαν από εμά, του πολιτικού ε, υπαλλήλου, του βοηθού, κινητοποιήθηκαν οι πάντε. Και στην παράγραφο 38 του ψηφίσματο, που υιοθετήσαμε τον Οκτώβριο του 2008, υιοθετήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέγαμε, ζητούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν ευρωπαϊκά ομόλογα και να επεξεργαστεί μια βραχυπρόθεσμη στρατηγική που θα επιτρέπει αυτά τα ομόλογα να, διατεθούν στο, να τεθούν στο επίκεντρο της Ευρωζώνης και επιπλέον των εθνικών ομολόγων αναφερόμενοι στην ανάγκη να αξιολογηθούν οι συνέπειες αυτού του μέτρου στις χρηματοστητικές αγορές και το... Όχι, όχι, όχι αγαπητέ συνάδελφε. Θυμάμαι πολύ καλά τη συζήτηση και αν διαβάσετε το σύντομο κείμενο της εκθέσεως που δεν αφορούσε την ανάπτυξη αλλά τη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση. Δεν προχώρησαν τα γρήγορα τα πράγματα και εγώ δεν θέλω να επαναλάβω την όλη φιλοσοφική προσέγγιση για να φτάσουμε στα ευρωμόλογα και ποιο θα πρέπει να είναι το πλαίσιο και ποιο θα είναι το γενικό, η γενική συμφωνία που θα μας επέτρεπε να προχωρήσουμε προς τα εκεί. Αλλά διαπιστώνω ότι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 28-29 Ιουνίου, αυτό το θέμα, παράλληλα με εκείνο για την Τραπεζική Ένωση, θα είναι στο επίκεντρο, στην καρδιά του μηνύματος που έχει κρατών και κυβερνήσεων θα θέλουν να στείλουν. Και για αυτό το λόγο ε, λυπούμε που δεν προχωρήσαμε πιο πέρα όταν ε, ψηφίσαμε την περασμένη εβδομάδα το 2 Διότι στο 2 Αναφερόμασταν στα ευρωμόλογα, το Ταμείο Διάσωσης, δυνατότητα οδικού χάρτη προς τα ευρωμόλογα κλπ. Και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσον αφορά την κατεύθυνση στην οποία θα θέλαμε να κινηθούμε. Εν γέννη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προηγείται του Συμβουλίου. Και η ιδέα μιας Επιτροπής Δελόρ, όταν όλα πηγαίνουν άσχημα, είναι μια ιδέα την οποία αρπάζονται όλοι. Και πρέπει να πω ότι οι παρούσε ομάδε εξάντλησαν ήδη αυτό το τύπο, αυτή την προσέγγιση. Όταν το Μάιο του 2010 ανέθεσαν στον πρόεδρο τον κύριο Βαν Ρομπόη να δημιουργήσει μια ομάδα εργασία όσον αφορά τη λειτουργία τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Λαμβάνοντα υπόψη τη ένθεση τη ομάδα, ε, δεν ήταν επιτροπή εντελώ αποκλειστικά και θα πρέπει να ξαναρχίσουμε, αλλά ε, Κάποιοι, αρχηγών, κάποιοι από του αρχηγού κρατών κυβερνήσεων αυτό έχουν υπόψη του το επόμενο συμβούλιο. Εάν ακολουθήσουν αυτή την πορεία τα πράγματα, καλό θα ήταν να συμμετάσχουμε κι εμείς όσον αφορά την ουσία. Είναι σημαντικό να ξεκολλήσουμε σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν και κάποια ανταλλάγματα και αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη πέρα των τεχνικών ρυθμίσεων. Διότι όσο προχωράμε στο θέμα βλέπουμε ότι περιπλέκονται τα πράγματα. Και όταν πούμε ευρωομόλογα δεν σημαίνει τίποτα αυτό, δεν λέμε τίποτα. Και κάθε θεωρητικός μπορεί να μας δείξει έναν νέο τρόπο προσέγγισης. Blue Bond, Euro Bills κλπ. Τι κρύβεται πίσω από αυτά αυτό που Βέρνα Λάγκεν ανέφερε, το δίκαιο, το νόμο. Πώς ερμηνεύεται η συνθήκη. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλες ερμηνείες στις συνθήκε. από την ερμηνεία του Βέρνα Λάγκεν. Πέραν αυτού, τίθεται και θέμα πολιτικού πλαισίου. Αντιστάθμιση χρειάζονται ευρωομόλογα. Και τα ανταλλάγματα δεν είναι αποδεκτά στις περισσότερες, ε, στην κοινή γνώμη των περισσότερων χωρών της Ευρώπης και χωρίς τα ευρωμόλογα, αν δεν ενισχύσουμε το πλαίσιο, αν δεν δώσουμε ευρωπαϊκό χαρακτήρα στην δημοσιονομική πολιτική, ε, πρέπει να ακολουθήσουμε σωστή προσέγγιση και να μην καταλήγουμε σε μέτρα λιτότητας. Άρα πρέπει να καθοριστούν προτεραιότητες Μιλάμε για δημιουργία νέων θέσεων εργασία και ανάκαμψη οικονομία, που είναι προπετούμενο για τελική συμφωνία όσον αφορά τα ευρωομόλογα. Τα λέμε αυτά όταν χρειάζονται κατεπήγοντα μέτρα. Αν μιλάμε για τα Ευρωπήλ, δεν είναι απλώ για θεωρία, γιατί κάποια κράτη-μέλη χρειάζονται κατεπηγόντω ε, χρηματοδοτήσεω των αγορών. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αν θέλουμε να βγούμε από τη θηλιά στην οποία παγιδευτήκαμε σήμερα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε απλώς επί ενός τομέα, επί ενός θέματος. Δεν είναι η τραπεζική ένωση ή ανάπτυξη, τα ευρώ ομόλογα ή η ολοκλήρωση, είναι ένα συνολικό πακέτο. Και είναι θεμητό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιληθεί του θέματος αντί να αφήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ασχοληθεί μόνη της. και να ασχολούνται με μονομένα κάτι μελη κάτι που βγάζει την πίεση από την ανάγκη ολοκλήρωσης. Αυτά ήθελα να πω σε αυτό το στάδιο των συζητήσεων, που είναι γενικού χαρακτήρα για την ώρα. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και αυτά που είπε ο Βέρναρ Λάγκεν, είπαμε ότι έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας και δεν την πειράξουμε παραπέρα. Πολύ λίγες αλλαγές θέλουμε να κάνουμε, ούτε στο δάχτυλο ενός χεριού. Αλλά δεν πρέπει να αυτό να το θεωρούμε. Αλλάξαν Αλλάξαμε συνθήκε τουλάχιστον δύο φορέ. Μπορούμε να το θεωρήσουμε σε ενδεχόμενο αυτό. Και να μην βάζουμε τις χώρες που είναι οι καλές και τα κάνουν όλα σωστά και άλλες. Αυτές τα πάνε καλά ευνοούνται από ένα ισχυρό νόμισμα, ένα νέο νόμισμα και θα πρέπει να επικρατήσει γενικά σε όλο το χώρο ένα πνεύμα αλληλεγγύης. Λυπάμαι που μακρηγόρησα όσον αφορά τις Ηνωμένες Δεν να συγκρίνουμε την Αμερική, τις Ηνωμένε Πολιτείε με την Ευρώπη και το είπε και η συγγήτρια. Ο Ομοσπονδιακός Υπολογισμός Αμερικανικός είναι ανάμεσα στο 20 και 30% του ΑΕΠ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί που είναι αντίθετοι στην προσέγγιση θέλουν τέτοιο επίπεδο ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αλλά σε αμερικανικό ομοσπονδιακό επίπεδο υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αντικυκλικού προπολογισμού. Οπότε δίθεται πρόβλημα χρέου με τον ίδιο τρόπο στι πολιτείε Αμερική όπω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε κοινή αντιμετώπιση των χρεών εδώ, ούτε δυνατότητα να έχουμε πραγματικά έναν προπολογισμό σε τέτοιο επίπεδο που να κινείται αντικυκλικά από την κρίση. Ευχαριστώ. Thank you. Um, now it's Astrid. Ευχαριστώ. Η Άστριντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα τα πω γερμανικά. Ε, μια σύντομη παρατήρηση για τον Βέρνερ Λάγκερ, αυτό που είπε για το Λουξεμβούργο ορίστε του έδωσα και τη σειρά μου και τι βρήκε να πει, είχα την καλοσύνη. Το πρώτο πράγμα που του ήρθε ήταν να επιτεθεί στη μικρή μου χώρα. Ε, πρέπει να πω ότι αν τόσοι Γερμανοί αφήνουν τα κεφάλαιά τους να τα διαχειρίζεται το Λουξεμβούργο, αυτό ονομάζεται, ξέρετε, ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου. Το έχουμε αυτό στην Ευρώπη. Εσωτερική αγορά, τέσσερις ελευθερίες. Των ανθρώπων, των εργαζομένων, του κεφαλαίου, των υπηρεσιών και των εμπορευμάτων. Οπότε Λοιπόν, να αναρωτηθούν οι Γερμανοί γιατί τόσες γερμανικές τράπεζες υπάρχουν στο Λουξεμβούργο. Για ρωτήστε τους ποια φορολογική πολιτική και τραπεζική πολιτική έκαναν στη Γερμανία για να οδηγήσει όλες αυτές τις γερμανικές τράπεζες στο Λουξεμβούργο. Αυτή είναι η ελευθερία του κεφαλαίου. Αυτά τα είπα λοιπόν στα γερμανικά και πάω στα γαλλικά τώρα. Θέλω να σας πω κυρία Πρόεδρε ότι στην έκθεση της συναδέλφου μου Σίλβιας Γκουλάρ έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία αλλά και μερικές ασάφειες που πρέπει να τις διορθώσουμε. Η ιδέα της κοινή ανάληψης των χρεών υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία είναι τα γαλάζια ομόλογα κοινά κάτω από τα όρια που θέτει η συνθήκη της Μαστρίχτης και για το χρέος άνω του 60% αυτό θα παραμείνει εθνικό. Κίνητρο λοιπόν για τα κράτη-μέλη να επανέλθουν στα όρια της συνθήκης. Γιατί το εθνικό χρέος θα ήταν έτσι πολύ πιο ακριβό από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αυτό λογικό. Το δεύτερο, η δεύτερη εκδοχή όμως ένα ευρωπαϊκό ταμείο απόσβεσης του χρέους που παρουσίασαν πρόσφατα γερμανοί οικονομολόγοι και που είναι και η πρόταση που συνήθως αναφέρεται ένα μέρος της μόνο καταλαβαίνω αλλά όχι το σύνολο γιατί μου φαίνεται ότι το κίνητρο για περισσότερη δημοσιονομική πειθαρχία είναι πιο ισχυρό από ό,τι στην προηγούμενη εκδοχή. Η να μου το λύσει αυτό. Ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά των δύο συστημάτων, των δύο εκδοχών. Η κοινή ανάληψη του χρέους άνω του 60% του ΑΕΠ μου φαίνεται κάτι πιο λογικό και λιγότερο επικίνδυνο αλλά θα έπρεπε να διαλέξουμε τη μία από τις δύο εκδοχές. Δεύτερον, η έκθεση της κυρίας Γκουλάρ θέλει να ευχαριστήσει όλους και γι' αυτό κάνει ένα σοβαρό λάθος. Αυτοί που γνωρίζουν τα πράγματα ξέρουν ότι η κοινή ανάληψη του χρέους δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνον εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει και δημοσιονομική ένωση αυστηρότατη. Δηλαδή τα κράτη ακολουθούν σιδηρούς κανόνες δημοσιονομικούς και να λέμε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία είναι κάτι καλό αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και πρόσθετα κριτήρια μου φαίνεται κάπως ελαφρότης. Τα ευρωομόλογα είναι νομίζω θα ήταν ό,τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Η συνθήκη δημοσιονομικής σταθερότητας δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου. Βέβαια οι αριστεροί δεν χαίρονται ιδιαίτερα, αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει εδώ επιβολή πάνω στα κράτη-μέλη των ευρωομολόγων, όποιο όνομα και να θέλουμε να τους δώσουμε. Όπως είπα και πριν, δεν γίνεται να υπάρξουν όλα αυτά χωρίς κάποια επιβολή. Και όλα αυτά θα παραμείνουν λοιπόν θεωρητικά. Αν η έκθεση θέλει να προχωρήσουμε τότε πρέπει να ενδυναμωθεί σημαντικά σε αυτό το επίπεδο έστω και αν ορισμένοι παρεξηγηθούν. Αλλιώς κινδυνεύει να καταλήξει ένα σιρτάρι και να μην χρησιμεύσει σε τίποτα. Αυτά ήθελα να σας πω. Αυτά. Θα αποφασίσουν άλλοι βέβαια και οι άλλοι για να δουν αν συμφωνούν όλα αυτά με το 125 της συνθήκης ή αν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε δηλαδή έτσι όπως λέει η έκθεση ή αν απαιτείται για να γίνουν όλα αυτά και μεταρρύθμιση των συνθήκων. Εγώ δεν πιστεύω πια σε μεταρρυθμίσεις των συνθήκων γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ δύσκολο μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα ενώ πρέπει ταχύτατα να βρούμε μια λύση για τα τωρινά μας προβλήματα στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό νομίζω ότι αν μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στα πλαίσια της υπάρχουσας συνθήκης, πολύ καλύτερα θα ήταν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αναθεώρηση της συνθήκης σύντομα. Ε, Ευχαριστώ. Λυπάμαι πάρα πολύ που ο κύριος Φόξ τα είπε και έφυγε. Μιλάει από μόνο του. πατάς το πόδι του άλλου, το κλωτσάς και μετά σηκώνεσαι και φεύγεις. Δεν θα πρέπει να αφήσω αναπάντητο κάτι που είπε, ότι που οφείλεται η κρίση του χρέους ότι πολλές χώρες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν υπερβολικές δαπάνες. Επιλέξει τα είπε αυτά. Μα τι είναι αυτές οι αναλήθειες. Η Ισπανία ε, βλέπε πριν ε, τη βρει η κρίση των τραπεζών, βλέπε η Ιρλανδία. Δεν μπορούμε να τα λέμε αυτά αβίαστα, αλλά μήπως δεν πρόλαβε να μάθει την απάντηση γιατί σηκώθηκε και έφυγε. Ε, ζήτησα το λόγο για να ευχαριστήσω και να συγχαρώ ε, την εισηγήτρια για αυτή την έκθεση, ε, ιδιαίτερα τα όσα είπε για το κρατικό χρέος και το Ταμείο Απόσβεσης. Προσωπικά με ενδιαφέρει αυτό και αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δώσουμε μια προοπτική για το μέλλον. Ότι κάποια στιγμή ε, θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και την κατάσταση που βρεθήκαν με χωρίς να θέλω. Θέλω να ρωτήσω κάτι για το σημείο 11. Καλό θα ήταν λίγο να επιμείνουμε εκεί και να αναφερθούμε και με άλλα πεδία που είναι λίγο γύρω-γύρω, δεξιά και αριστερά από το πραγματικό αντικείμενο της έκθεσης, αλλά δεν ξέρω αν το Ταμείο και Κεφαλαιοποίησης και ένας μηχανισμός ε, σταθεροποίησης ε, πρέπει να ε, αναφερθεί εδώ. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ε, σύστημα ασφάλειας των καταθέσεων ε, πανευρωπαϊκό ήταν κάτι που μας ε, απασχόλησε και την περασμένη εβδομάδα για οξύς κινδύνους και απειλές. Γιατί δεν είχαμε έναν τρόπο άμεσης αντίδρασης σε απειλές, παρά μόνο μεσοπρόθεσμες. Γνωρίζει η Πρόεδρος ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να έχει ενιαία άποψη, αλλά οι εξελίξεις προχωρούν με βραδείς ρυθμούς γιατί δεν ε, τα βρίσκει το Συμβούλιο. Για το σύστημα εγγύησεων και ε, εξασφάλισης ε, είναι πολύ διαφορετική και η παράδοση από χώρα σε χώρα γιατί είναι και τελείως διαφορετικό το τραπεζικό σύστημα κάθε χώρας. Και μπορεί κάπου να υπάρχουν κάπου καλές και πολύ παλιές εγκατεστημένες και δρομένες τράπεζες και συστήματα εθνικά, ισπανικά βλέπω τον Ισπανό συνάδελφο δίπλα. Ε, σε αυτή λοιπόν τη συζήτηση δεν θα πρέπει να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Ε, μπορεί να είναι ε, παραπλήσιο, αλλά δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει σε τούτη εδώ την έκθεση. Θέλουμε να αποφύγουμε ε, στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, αλλά να αφήσουμε όσο γίνεται ελεύθερη την επικουρικότητα προς τα κάτω, γιατί ακριβώς έχουμε διαφορετικές τραπεζικές παραδόσεις. Ε, παρακαλώ λοιπόν να το αλλάξουμε αυτό ή να μην το συζητήσουμε στην παρούσα έκθεση. Η Σοφή, είναι τβέλτς. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποια γενικά σχόλια. Αφού άκουσα την όλη συζήτηση αναφερθήκαμε σε διάφορα μοντέλα. Συζητήσαμε την ε, σωστή μελλοντική πορεία. Δύσκολο να αποφασίσουμε. Υπάρχουν πολύ καλά επιχειρήματα για τις διάφορες ε, λύσεις. Νομίζω ότι είναι σημαντικότερο να διαλέξουμε, να πάρουμε μια απόφαση να μην κάνουμε αυτό που κάναμε πριν από 10-12 χρόνια με, που καταλήξαμε σε ημίμετρα ατελείς λύσεις μια ευρωζώνη ατελή λόγω του φόβου να πάρουμε αποφάσεις λόγω του φόβου μας απέναντι στο εκλογικό σώμα ό,τι και αν κάνουμε θα πρέπει να το κάνουμε μέχρι τέλους δεν θέλουμε ημίμετρα δεν θέλουμε μισές λύσεις δεν θέλουμε αποδυναμωμένους συμβιβασμούς που δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, δεν τίποτα τελικά διότι ο φόβος να πάρουμε απόφαση, ο φόβος μας να δημιουργήσουμε πλήρη πολιτική ένωση, μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση και στα προβλήματα. Να ξεκαθαρίσω και κάτι, ότι ανήκω σε εκείνους που είναι υπέρ της δημοσιονομικής πειθαρχία και πολύ μάλιστα. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να με χρήματα να βγούμε από την κρίση. Δεν είναι καλό συστηματικά να δαπανά κανείς περισσότερα από αυτά που κερδίζει. Το ξεκαθαρίζω. Ε, αυτή είναι η θέση μου. Όμως αυτοί οι ηθικοί κίνδυνοι που αναφέρονται καθιστά όμοιρο τη συζήτηση. Τι είναι αυτό ο ηθικός κίνδυνος. Γιατί λέμε ότι υπάρχουν ηθικές και μη ηθικές χώρες. Για ποιο ήθος μιλάμε. Εδώ μιλάμε για πολιτικές επιλογές. Δεν υπάρχει κάτι σαν πιο ηθικός βόρειος και σπάταλος νότιος. Είναι θέμα πολιτικών επιλογών και εδώ στον κύριο Φόξ. Ο συνάδελφός μας που εκπροσωπούσε είναι πολύ κοντά σε Ολλανδικά κόμματα που προσπαθούν να μπλοκάρουν τη λιτότητα. Λοιπόν, έχουμε τους βόρειους ηθικούς παραγωγικούς βόρειους που είναι κατά των ανήθικων νότιων. Τι είναι αυτό. Οι νότιες χώρες που συζητούμε κάνουν πολλά περισσότερα για να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις από τη χώρα μου που υποτίθεται είναι πάρα πολύ προκομμένη και εργατική. Δεν είναι θέμα μαύρου με άσπρο, αν υπάρχουν μέτρα διαφύλαξης και εγγύησης σε ένα σύστημα που θα δημιουργήσουμε που δημιουργούν εμπιστοσύνη, αυτό είναι το πιο σημαντικό, διότι περί αυτού πρόκειται. Εμπιστοσύνη. Δεν θα υπάρχουν εγγύησει 100%. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο, δεν θα χρειαζόταν εμπιστοσύνη. Πρέπει να εμπιστευτούμε ένα τον άλλον. Σε κάποιο στάδιο είναι και θέμα εμπιστοσύνη. Αν συμφωνούμε επί κανόνων, ότι όλοι θα συμμορφωθούν με του κανόνε. Και αυτό δεν είναι το πρόβλημα μέχρι τώρα. Το πρόβλημα μέχρι τώρα δεν ήταν η κοινή αντιμετώπιση του χρέους. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Αντιθέτως, το πρόβλημα ήταν ότι δεν εμπιστευόμασταν οι μεν τους δε. Και δεν είχαμε και κανόνες που να γίνονται σεβαστοί από όλους. Όταν η Ευρωπαϊκή Επίτροπη πρότεινε να έχουμε πιο δεσμευτικούς κανόνες, αυτό το σταμάτησαν αυτές οι προκομμένες χώρες υπό την ηγεσία Ολλανδίας-Γερμανίας ό,τι και αν διαλέξουμε, ας οδηγήσει σε μια πλήρη πολιτική ένωση, όχι μη μέτρα, όχι συμβιβασμούς, που δεν αποτελούν ούτε εθνική ούτε ευρωπαϊκή λύση. Ας πάμε για πλήρη πολιτική ένωση, ας διαλέξουμε αυτό. Καλώς. Ξερόβα, που είμαι Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Τέρχο, και ευχαριστώ την συγκήτρια, είναι σαφές το κείμενο. Στο παράρτημα αναφέρονται τα ευρωομόλογα και διάφορα άλλα χρηματοπιστωτικά ε, μέτρα της ε, αντιμετώπισης του χρέους. Αναφέρεται και διάφορα ηθικά ειδική κίνδυνη για την αντιμετώπιση του χρέους και η δημοκρατική νομιμότητα που είναι απαραίτητη για την κοινή αντιμετώπιση του χρέους. Από την πλευρά μου πρέπει να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε πώς τα ευρωμόλογα ή η αδίποτε, κοινή ευθύνη, η κοινή αντιμετώπιση σαν αφετηρία δίνει κάποια λύση και εγώ αναφέρομαι σε όλες τις χώρες Ευρώπης και τις νότιες και τις βόρειες όταν αναπτύσσω τα επιχειρήματά μου. Δεν κρίνω ηθικά τις χώρες γεωγραφικά. Και η δική μου χώρα, η Φιλανδία, ξοδεύει περισσότερα από αυτά που εισπράττει. Λοιπόν, η κοινή αντιμετώπιση, η κοινή ευθύνη στον φωτοχρέος είναι ένα βήμα προς ομοσπονδιακή λύση. Και εδώ η δημοκρατική νομιμότητα είναι κρίσιμη σημασία. Αν δεν υπάρχει αυτή η νομιμότητα και αν δεν τη δώσουν οι πολίτες τις αποφάσεις που παίρνουμε, αυτή την δημοκρατική νομιμότητα, τότε οι λαοί δεν θα εγκρίνουν τις αποφάσεις. Και θα αναπτυχθεί μια νοοτροπία αντιευρωπαϊκή, θα δημιουργηθούν κοινωνικέ αναταραχές και ο κόσμο δεν θέλει να πληρώνει φόρου πια. Δημιουργείται αυτός ο κίνδυνο Γι' αυτό πριν την κοινή αντιμετώπιση του χρέου, πριν οποιαδήποτε λύση χρειάζεται μια σοβαρή κουβέντα. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν τα μέτρα. Όχι μόνο οι πολιτικοί, αλλά και οι πολίτε. Είναι ζωτική σημασία η υποστήριξη των πολιτών. Όσον αφορά τη χώρα μου, τη Φιλανδία. Πρέπει να πω ότι στη χώρα μου οι πολιτικοί μας δεν υποστηρίζουν τα ευρωομόλογα και η κυβέρνησή μα και η αντιπολίτευση ήταν κατά των ευρωομολόγων. Έχουν δημιουργήσει ένα σχηματίσει ένα κοινό μέτωπο. Και πιστεύω ότι στη Φιλανδία ίσω μόνο οι πράσινοι που έχουν το 5% των εδρών ίσω να είναι υπέρ των ευρωομολόγων. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ο Βέρνερ θέλει να επιτεθεί εκ νέου στο Λουξεμβούργο. Ε, Όχι, εγώ προ Θεού. Απλώ να εξηγήσω κάτι γιατί ε, συνεχώς αναφέρεται η πρόταση της ε, Γερμανικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Αν είναι ε, πάνω από 60% το χρέος. Σε αυτό το ταμείο το πολύ πολύ να συμμετέχουν 8 από τις 17 χώρες της Ευρωζώνης. Γιατί είπαν ότι οι χώρες που είναι σε άλλο πρόγραμμα προστασίας δεν συμμετέχουν. Πορτογαλία, Ελλάδα, ε, Ιρλανδία και πρόσφατα Ισπανία. Δεύτερον, χώρες που έχουν κάτω από 60% χρέους επίσης αποκλείονται. Εστονία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Σλοβακία. Αποτέλεσμα. Ταμείο Πόσβεσης που αποφασίσαμε την περασμένη εβδομάδα με αυτή τη στιγμή όγκο 2,3 δις ευρώ ε, σε μεγάλο βαθμό ε, αφορά την Ιταλία. 975 δισεκατομμύρια και 530 ε, ως Γερμανία, που είναι ο δεύτερος υπερχρεωμένος. Δηλαδή το δίλημα που παρουσιάσει ο κύριος Μόντι δεν ε, είναι ε, σωστά. Για να καταλάβουμε τι εννοεί αυτή η Επιτροπή. Είναι 2,33, όχι δις προφανώς. θα πρέπει να τα διαβάζουμε σωστά αυτά. Πρώτα να κάνουμε ε, βήματα για την πολιτική ένωση, μετά αύξηση σημαντική του κοινοτικού προπολογισμού. Πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν υπογράψει αυτό το γράμμα για το πολύ 1% μέγα σφάλμα για μένα. Και το τρίτο, δημοσιονομική ένωση ε, με Ευρωπαίο Υπουργό και ε, θέση σε ισχύ τους μηχανισμούς σταθεροποίησης. Όλα αυτά με αν θα το τροποποιήσουμε και θα αναθεωρήσουμε τις συνθήκες για τα ευρωμόλογα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έβαλα και εγώ τον αυτό μου στον κατάλογο των ε, αγορητών. Προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Βεβαίω ήδη ψηφίσαμε υπέρ του Ταμείου πληρωμή του χρέου, το ΤΟΥΠΑΚ. Φοβούμαι όμω ε, ψηφίσαμε για σωτηρία, αλλά κανείς δεν έχει ε, δηλώσει θελοντής για τη σταύρωση, για τη σωτηρία. Και αυτό πρέπει να το επιλύσουμε. Όπως ανέφεραν και κάποιοι άλλοι, Ζαν Πολ, Ήδη έχουμε τη σωτηρία. Άρα δεν χρειάζεται η σταύρωση. Το σχόλιο. Α, μάλιστα. Χαίρομαι που θεωρείς ότι ήδη λυτρωθήκαμε. νομίζω ότι είναι ή όλα τίποτα τώρα, γι' αυτό παίζουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι που μπορούμε να το λύσουμε γρήγορα, παρά το γεγονό ότι μου στην πρώτη γραμμή διαμαρτυρώμενοι τα κράτη-μέλη έκαναν πολύ λίγα πράγματα πολύ αργά όταν προσπαθούσαν να δημιουργήσουμε μηχανισμό διάσωση όσον αφορά τεράστια θέματα. Για τη δημιουργία μια οικονομική ένωση είναι σαφέ ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει γρήγορα. Και αν δούμε την αμοιβαία αντιμετώπιση, την κοινή αντιμετώπιση, νομίζω ότι έχουμε μεγάλα προβλήματα αν προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι που γίνεται πολύ γρήγορα, όταν ουσιαστικά ζητούμε τη Γερμανία και τη Γαλλία να επομισθούν τρεις με τέσσερις φορές το ΑΕΠ τους σε έκθεση έναν ευθυνών. Λοιπόν, εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι πιο βραχυπρόθεσμα, ξεκινήσουμε από αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε περιορισμένη ευθύνη, κοινή προσέγγιση μέσω περιορισμένη ευθύνη, κάτι που έγινε με τι εγγυήσει στο EFSF. Αυτό από μόνο του όμως ε, ε, δεν καλύπτει το μακροπρόθεσμο, τη μακροπρόθεσμη λύση. Μακροπρόθεσμα είναι μια απόφαση. Ή όλα ή τίποτα. Αλλά χρειαζόμαστε χρόνο για αυτή την απόφαση. Γι' αυτό επί μακρόν υποστήριζα κάτι που είναι πιο πράχη πρόθεσμος μηχανισμός σωτηρίας. Όπως ε, τα T-bills, μικρότερα χρήματα διατίθεται με αυτόν τον τρόπο, μικρότερα ποσά, περιορίζεται, δεσμεύεσαι για μικρότερο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω, δύο χρόνια, τέσσερα χρόνια. Μας δίνουν χρόνο όμως, ούτω ώστε τα μελλοντικά βήματα, τα πιο μακροπρόθεσμα προς τη μελλοντική οικονομική ένωση, που πιστεύω πως εκεί πρέπει να πάμε, να εφαρμοστεί σωστά. Δεν μπορούμε να επιδείξουμε όμως μέσω λοιπόν λύσεων βιαστικών, όπως κάναμε αρχικά με το ευρώ. Πρέπει να είμαστε και ειλικρινεί. Ήταν πιο ειλικρινέ από τα άλλα θεσμικά όργανα το Κοινοβούλιο. Εμείς δεν φοβόμαστε. Παρουσιάζουμε ε, τα κρατικά ομόλογα, τα προβλήματα, τη μη ύπαρξη μηδενικού κινδύνου, κάτι που δεν μπορεί να επιληθεί άμεσα. Αλλά η διαφορά στο τριμερή διάλογο είναι αυτή. Κάθε εβδομάδα αντιμετωπίζουμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο που δεν ανέχονται την εξέταση των κρατικών ομολόγων μηδενικού κινδύνου. Και στο, στο θα Και αυτό δείχνει ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πριν φτάσουμε στην απόφαση αυτή ή όλα ή τίποτα. Ευχαριστώ λοιπόν που έλαβες υπόψη σου αυτή την πρόταση για αυτά τα ομόλογα σταθερότητα. Ε, ίσως και θα πρέπει να είναι και ε, να μπούμε και στην προσέγγιση πιο περιορισμένης ευθύνη αντί κοινή προς, ε, αντιμετώπιση του χρέους. Αν το δεις πώς το βλέπουν οι αναλυτές των αγορών, το θέμα λέτε σε κάποιους κατοίκους μιας χώρας αναλαμβάνετε όλο το χρέος στα κοιτάπια σας. Δεν ισχύει αυτό. Ελπίζετε να μην χρεοκοπήσουν όλοι όμως τελικά. Πρέπει να είμαστε πιο φευρετικοί. Πρέπει να δούμε όλες τις επιλογές. Να βρούμε ποιος ήταν ο δρόμος για το μέλλον. Και είναι καλό που είναι μαζεμένες όλες οι εναλλακτικές και δίνω το λόγο στη Σιλβίου ώστε να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ λοιπόν, ευχαριστώντας όλους όσους μίλησαν και όσους άκουσαν με τα προσοχής. Να πω λοιπόν το θέμα της πειθαρχίας και το θέμα ηθικό. Δεν θα πρέπει αυτή την έκθεση να την εξετάσουμε ανεξάρτητα με αυτά που ήδη κάναμε και προσωπικά στο Six Pack έδωσα μάχη και κατά της γαλλικής κυβερνήσεως της του παρελθόντος για την αυτόματο χαρακτήρα των κυρώσεων. Μια εποχή που η κυρία Μαρκέλ και ο κ. Σαρκοζή έκαναν συμφωνίε για να περιοριστεί ο αυτόματο χαρακτήρα τη θεσισχή τη πειθαρχία. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να σταματήσει ο διαγωνισμό του πιο πειθαρχημένου και του πιο ηθικού κλπ. Έχουμε κείμενα, τα θετήσαμε αυτά και θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη δική μα την νομοθεσία όπου μπορούμε να ε, προσθέσουμε και το Fiscal Compact. Δεν θα απαντήσει τον κύριο Φόξ, που όπως συνήθω έκανε ένα νούμερο όπου μας έδωσε μαθήματα για μια ευρωζώνη στην οποία δεν ανήκει. Δεύτερον, όσον αφορά το νομικό ζήτημα, απαντώντας στον Βέρναρ Λάγκεν, εγώ για μία ακόμη φορά είμαι πολύ ευαίσθητο όσον αφορά τα νομικά επιχειρήματα που προβλήθηκαν στη Γερμανία και εδώ δεν θέλουμε σε μια κοινότητα δικαίων να παραβιάσουμε τι συνθήκε. Νομίζω απλώ ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε επί του τρόπου με τον οποίο ερμηνεύουμε τι συνθήκε, διότι υπάρχουν δύο οπτικέ γωνίε. Είτε έχουμε εμπόδια νομικά, τα οποία σεβόμαι και προσπαθούμε να βρούμε λύσει, είτε κρυβόμαστε πίσω από τα νομικά εμπόδια για να ρυθούμε τα πάντα. Και εκεί, Βέρνερ, καμιά φορά δεν αισθάνομαι πολύ άνετα. Ανησυχώ. Διότι βλέπω κάποια αρνητικά μηνύματα που αποστέλλονται από τη Γερμανία ή τουλάχιστον από ένα κομμάτι τη κοινή γνώμη στη Γερμανία. Πολύ συχνά είμαι στη Γερμανία επί τόπου για να μιλήσω άμεσα με το κοινό. Ξέρω ποια είναι η κοινή γνώμη. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε μια ένωση εντός της οποίας υπάρχει καταρχήν άρνηση και κάποιοι που κρύβονται πίσω από την ομολογία ενό δικαστηρίου που σέβομαι πάρα πολύ. Και επισημαίνω στου Γερμανού φίλου ότι ακόμα μπήκα στο κόπο να συναντήσω και ένα δικαστή του δικαστηρίου. Μπορούμε να συζητήσουμε. Σίγουρα υπάρχει μια δέσμευση μέχρι τώρα των χωρών τη Ευρωζώνη. Μιλώ και για τη Γαλλία και τη Γερμανία. Εντό του ευρωπαϊκού συστήματο και με το Target 2 και με το σύστημα αυτό, ήδη έχουμε εγγύσει που προχωρούν πολύ μακριά. Λοιπόν, θα πρέπει όλοι να έχουμε μια προσέγγιση που μας επιτρέπει να δούμε ποιο είναι το εφικτό, τι μπορεί να εφαρμοστεί με φύη προσέγγιση εντός του δικαίου. Όταν λένε οι Αμερικανοί yes we can, εμείς ε, πρέπει να πούμε το ανάλογο. Και πρέπει να βρούμε τη σωστή απάντηση που θα πείσει τις αγορές. Είμαι ανοιχτή όσον αφορά τις τροπολογίες που θα έρθουν από το ΕΛ και από τους συναδέλφους κάθε εθνικότητας, αλλά λέω απλώς α προσπαθήσουμε να έχουμε προσέγγιση η οποία θα είναι επικοδομητική και η οποία θα ενοποιεί την Ευρωζώνη και τη στερεώνει. Διότι αν διατηρηθεί η, η, τελικά η τελειομανία των νομικών, ίσως κολλήσουμε. Λοιπόν, αυτά που στον Μπεζέ. Εγώ έλεγα ότι θα έπρεπε να γίνει μια ανάλυση και μια ανάλυση που δεν έχει γίνει από τους Υπουργούς Οικονομικών εν πρώτης όσον αφορά τη λύση των ομολογών. Μπορεί κάποιο άλλο να το αναλάβει. Αλλά εκείνοι που είναι ικανοί και εκπροσωπούν τη χώρα του, αλλά οι οποίοι δεν είναι στην κυβέρνηση άμεσα, ε, νομίζω ότι αν το συζητήσουν αυτοί θα βοηθούσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεύτερον, λοιπόν, απαντώ στην Περβάουνς. Είπε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν ήταν μια αναφορά κλπ. Σημείο αναφορά. Εγώ παρατηρώ ότι παρόλα αυτά πάντα γίνεται αναφορά στη ΣΥΠΑ. Τι έχουν υπόψη του οι διάφοροι. Ε, την αγορά του T-bill του Αμερικανικού. Είτε μα αρέσουν είτε όχι, είναι το σημείο αναφορά. Κάνουμε σύγκριση μεταξύ ενό ομοσπονδιακού κράτου που έχει ηλικία 200 ετών και τη Ευρώπη οικοδομείται πολλοί που κρίνουν το ευρώ έχουν αυτό υπόψη τους. Πρέπει να να δούμε ότι η κοινή αντιμετώπιση των εθνικών χρεών είναι μια πρωτότυπη προσέγγιση που θα μπορούσε να ακολουθήσει η Ευρώπη, αλλά υπάρχουν και άλλες λύσεις. Απαντώντας στην Astrid Luling, ναι, βεβαίως υπάρχουν και τα συν και τα πλήν, ε, διαφορετικά ωφέλη και μειονεκτήματα εναντί της λύσης Blue Bond και του Redemption Fund, εγώ δεν κρύβω από την έκθεσή μου, παρόλο που είναι πολύ σύντομη, ότι υπάρχουν και αρνητικά στοιχεία. Με το Ταμείο Διάσωσης, το Redemption Fund Σωτηρίας, μπορούμε να συγκρατήσουμε το χρέος και στην εκδοχή τη γερμανική έχουμε αιρεσιμότητα ότι δεν καλύπτουμε το χρέος πάνω 60%, θέλουμε να μειώνεται το χρέος και αφήνουμε τα κράτη-μέλη να χρεωθούν για τα υπόλοιπα. Αυτό προϋποθέτει βεβαίως για μια ακόμη φορά ελέγχους οι οποίοι είναι πάρα πολύ προθυμένοι. Εγώ πρέπει να πω ότι σε επαφές που ήρθα στις διάφορες πρωτεύουσες σχεδόν στις χώρες του Νότου έχουν περισσότερες αντιστάσεις όσον αφορά το Ταμείο Σωτηρίας. Διότι υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τις εκδόσεις εθνικών ομολόγων. Όσον αφορά το Blue Red των Γερμανών ειδικών, αυτό που λένε οι συντάκτες του κειμένου και οι οικονομολόγοι λένε ότι το επιπλέον χρέος, χρηματοδότηση στο χρέος πέρα από το 60% θα μπορούσε να γίνει μεγάλο πρόβλημα για τις χώρες που έχουν πολύ μεγάλο χρέος πέρα από το 60%. Άρα υπάρχει ένα κίνητρο πράγματι να περιοριστεί το εθνικό χρέος. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι χώρες μόνες τους πρέπει να πάνε τότε στην αγορά Αντίθετα θα πρέπει το επιπλέον κόστος που δημιουργείται λόγω του κόκκινου χρέους πάνω το 60% δεν εξουδετερώνει τα ωφέλη από την κοινή έκδοση ομολόγων που καλύπτουν το κάτω από το 60%. Όπως λέει και η Σοφή θα πρέπει να επιλέξουμε. Εγώ ειλικρινά θέλω να το ξαναπώ εδώ προσωπικά. Δεν έχω καμία ε, προκατάληψη. Εγώ μπορώ να απολύσω και το blue και το red και το redemption κλπ βλέπω ότι έχουμε δι, ε, διχασμό βορρά-νότου στη Γαλλία. Σαν Γαλλίδα που είμαι κοντά στους Ιταλούς, στους Γερμανούς κλπ. Το βλέπω. Και αυτό με στενοχωρεί φάνταστα. Αν δι, αυτό το χάσμα συνεχιστεί βορρά-νότου εντός της Ευρωζώνης θα έχουμε τεράστια προβλήματα για να βγούμε όλοι μαζί από το πρόβλημα από κοινού. Ας προσπαθήσουμε να αποφασίσουμε μαζί, είμαι ανοιχτή σε τροπολογίες, αν υπάρχουν και δεν θα τις ακούσω, αλλά προσπαθήσουμε να έχουμε υπόψη ότι χρειάζεται μια λύση και για τους μεν και για τους δε. Για όλους και μιλά μια μητέρα πολυτέχνης ε, οικογένειας. Λοιπόν, ανέφερα στο πράγμα της τράπεζες. Είναι η έκθεση για το μέλλον του ευρώ, δεν είναι για τις τράπεζες. Σε μια μικρή παραγραφούλα έλεγα ότι αν δεν βρούμε λύση όσον αφορά το τραπεζικό τομέα, Μπορούμε να φανταστούμε ό,τι ευρωμόλογα θέλετε, ό,τι είδου ευρωμόλογα, δεν θα τα καταφέρουμε όμω. Πρέπει να γίνει μια τράπεζα τραπεζικό τομέα. Μπορούμε να επανεξετάσουμε την παράγραφα αν θέλετε, αλλά ήθελα να σα δείξω απλώ τη συζήτηση αυτό. Ότι είχα δει το πρόβλημα. Θυμίζω όμω ότι ξεκινήσαμε σε αυτό το κοινοβούλιο, στο πακέτο για την εποπτεία, να υπογραμμίζουμε και στην έκθεση τη Ελίζα Φεραίρα όσον αφορά τη λύση του προβλήματο, το ψήφισμα τη τράπεζε, ότι χρειάζονται πράγματα να γίνουν. Το είπαμε εδώ και δύο χρόνια. Νομίζω ότι συνόψισα τα πάντα, αν κάποια πράγματα. Ε, ζητώ συγγνώμη και ευχαριστώ για αυτή την πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Ε, ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία. Κατάθεση τροπολογιών. 9η Ιουλίου. Συζήτηση 3η Σεπτεμβρίου. Στι 12 το μεσημέρι. Ε, και ψηφίζουμε στις 19 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια ελπίζουμε τον Οκτώβριο. Θα δείξει όμως ακόμα, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ και προχωρούμε στο σημείο 5, τροποποίηση του άρθρου 70. Μήπως να σας αφήσω δύο-τρία λεπτά να αποχωρήσουν ως θέλουν για να μην χρειάζεται να φωνάζω. Okay, λοιπόν, Αν θέλετε να αποχωρήσετε παρακαλώ συντόμως γιατί έχουμε και θέμα. Σβέρν um, και Βέρνα, σας παρακαλώ τα πηγαδάκια έξω, γιατί θα θέλαμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Okay. Right. Um, this is the... Λοιπόν, που είχαμε μείνει στην τροποποίηση του άρθρου 70 του κανονισμού σχετικά με τις διοργανικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών. Μήπως να σας θυμίσω γιατί είμαι εγώ η συγγήτρια, διότι την χάνω πρόεδρος της Επιτροπής και δεν υπήρχε ομάδα που να ήθελε να αναλάβει αυτό το θέμα. Και μου είπε ο κλήρος να είναι εγώ η συγγήτρια. Συμβαίνει συχνά κάτι τέτοιο, συνήθως με στατιστικές και τέτοια θέματα, αλλά τώρα πρόκειται για ένα διοργανικό ζήτημα. Λοιπόν, η συζήτηση των τροπολογιών, εξέταση, 19 των αριθμών κατατέθηκαν, αρκετές δικές μου. Ε, προσπάθησα να ε, ε, αντανακλάται έτσι η συζήτηση που είχαμε για την αρχική έκθεση. Και στην αρχική έκθεση προσπάθησα να συμπεριλάβω και αυτά που ζητάει η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ΑΦΚΟ, γιατί δεν μας άρεσε πάρα πολύ η αρχική διατύπωσή τους και έκανα και κάποιες τροπολογίες για να το προσαρμόσω λίγο στη δική μας γλώσσα. Τέσσερα είναι τα κύρια θέματα ε, στις τροπολογίες. Πρώτον, για απόφαση της Επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Και πώς θα γίνει αυτό. Στις δικές μου τροπολογίες εγώ τι ζητώ. Να προσπαθήσουμε να καταγράψουμε και να περιγράψουμε τι κάνουμε ήδη εδώ. Ότι έχουμε τακτική έκθεση για την πορεία των διαπραγματεύσεων στους τριμερείς διαλόγους, αλλά πριν γίνει αυτό, όπως έκανα και σήμερα, το φέρνουμε στην Επιτροπή. Και αν κάποιος έχει αντίρρηση να προχωρήσει το θέμα, τότε ε, αν χρειαστεί προχωρούμε και σε ψηφοφορία. Νομίζω ότι είναι σωστό αυτό να μην γίνεται ψηφοφορία όταν δεν το περιμένουν οι βουλευτές αλλά να είναι ενήμερη, Όταν έχουμε και άλλες ε, ψηφοφορίες δοντάσουμε ε, και αυτό. Και όχι ξαφνικά και απροειδοποίητα όταν έχουμε τέσσερις βουλευτές παρόντες ξαφνικά ε, ψηφοφορία. Έτσι, προτείνω λοιπόν μαζί με πολλούς άλλους ότι όταν ε, υπάρχει η ψηφοφορία να είναι με απλή πλειοψηφία. Ο Βέρνερ Λάγκεν ήθελε πλειοψηφία δύο τρίτων σε δική του τροπολογία. Αν εφαρμόσουμε αυτό το κανόνα, καήκαμε με το six pack. Δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσει. Γιατί πού να βρει πλειοψηφία δύο τρίτων για να αρχίσουν διαπραγματεύσει για τι συζητήσει για το πακέτο, το δέσμευτη των έξι νομοθετημάτων. Οπότε, θα έπρεπε να πάμε και σε δεύτερη ανάγνωση. Και ξέρετε ότι στη δεύτερη ανάγνωση δεν έχουμε νέε τροπολογίε. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να έρθουμε μέτωποι ε, το Συμβούλιο, γιατί ήταν πολύ σφιχτέ οι ψηφοφορίε, έξι ψήφοι αν δεν απατώμε, όταν πήγαμε στην Ολομέλεια. Επί τη βάσεως αυτή, λοιπόν πιστεύω ότι δύο τρίτα πλειοψηφία για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, ε, ε, πλειοψηφία τη Επιτροπής δεν είναι καλή ιδέα. Οι ειδικέ πλειοψηφίε ενισχυμένε έχουν τη θέση του, αλλά στη διαδικασία δεύτερη ανάγνωση στην Ολομέλεια και όχι σε επίπεδο ε, κοινοβουλευτική Αλλά περιμένω να ακούσω με ενδιαφέρον τι έχετε να πείτε. Υπάρχει και πρόταση του κυρίου Γκουαλτιέρη η απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων να μεταφράζεται και να μοιράζεται σε όλα τα μέλη. Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι απαραίτητο αυτό. Στις ανακοινώσεις της Προέδρου θα ζητούμε καμιά φορά να υπάρξει ψηφοφορία ή απόφαση για την έναξη διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της Επιτροπής. Και αν είναι επίσημη και τυπική ψηφοφορία, να είναι στη διάθεση όλων, αλλά ουσιαστικά είναι προφορική ε, διαδικασία, αφόσον έχουμε και διαρμηνία, δεν χρειάζεται να μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες και να διανέμεται. Επίσης, η εντολή μπορεί να ενημερώνεται στην πορεία των διαπραγματεύσεων, να ανανεώνεται το κάναμε αυτό για το six pack χωρίς να αλλάξουμε την ψηφοφορία. Σε τακτά χρονικά διαστήματα αναφέραμε την κατάσταση των πραγμάτων και συζητούσαμε τις προτεραιότητες. Νομίζω είχε γίνει τότε από τους εισηγητές αυτό και ε, υπάρχει συνένεση ε, κατά τη διάρκεια της πορείας. Αυτό μπορεί να θεσμοθετηθεί και να επισημοποιηθεί. Το τρίτο αφορά την αναπομπή στην ολομέλεια της απόφασης έναρξης διαπραγματεύσεων. Προφανώς αν διαφωνεί η Επιτροπή ή αν διαφωνούν με τα όσα έκανε η Επιτροπή μας, γιατί δεν είναι μόνο η δική μας, είναι και άλλες επιτροπές, παραπέμπεται το θέμα στην Ολομέλεια. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικέ εδώ, ενδεχομένως κατόπιν αιτήματο μιας πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον 40 μελών, που είναι η συνήθις διαδικασία υποθέτω, για να πηγαίνουν τα θέματα στην Ολομέλεια. Εγώ πρότεινα ενδεχομένω δύο πολιτικές ομάδες ή 40 μέλη. Για να μην μας γίνει αυτό ρουτίνα και συνήθεια να τα πηγαίνουμε όλα στην Ολομέλεια, μία πολιτική ομάδα, πάγια, ε, θα ήταν περίεργο κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό ε, είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσουμε. Άλλη εναλλακτική ήταν ένα δέκατο των μελών του Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν τουλάχιστον δύο πολιτικές ομάδες ή αν έτσι αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων. Να μπορεί δηλαδή να επεμβαίνει η διάσκεψη των Προέδρων σε περίπτωση ε, που υπάρχουν πολύ έντονες ε, διπαραθέσεις και θέλουν να το πάνε στην Ολομέλεια. Αυτές είναι οι εναλλακτικέ λύσεις που προτείνονται και πρέπει να αποφασίσουμε η σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας. Είναι κάτι που με απασχόλησε και πάλι. Ε, ε, η πρόεδρος συν εισηγητής, συν σκιώδης εισηγητές. Και διευκρινίζω ποιος κάνει τι. Ο πρόεδρος προεδρεύει επίσημα στις διαδικασίες και ενδεχομένως ε, ηγείται και στα διοργανικά ζητήματα. Αυτό κάνω εγώ αυτόν τον καιρό για θέματα όπως είναι η κατεξουσιοδότηση πράξης. Δηλαδή, αυτά τα διοργανικά ελπίζω να τα λύσουμε και να ξεπεράσουμε τα εμπόδια για πολλές διαπραγματεύσεις που ε, διεξάγονται για τις πολιτικές. Δηλαδή, έχω ξεχωρίσει τις διοργανικές μάχες που δίνουμε από τα ζητήματα της πολιτικής ουσίας και αυτό έχει γίνει και με τρόπο χρήσιμο και εποφελή στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, ο εισηγητή επίση έτσι κι αλλιώ που ε, συνηθίζει να ηγείται σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαπραγμάτευση και την εντολή. Και όλες οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να εκπροσωπούνται και αν χρειάζεται χωρίς να ενθαρρύνουμε αυτή την ε, ε, οδό να μπορούν να εκπροσωπούνται από αναπληρωτές σκιώδεις και τέτοιους χωρίς να γίνει αυτό κάτι πάγιο και σε ορισμένες περιπτώσεις διαπραγματευτική ομάδα μπορεί να διευρύνεται. Το έχουμε ξανακάνει και πάλι στο Six Pack είχαμε και τους συντονιστές όλους γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητη η παρουσία τους. Μην νομίζετε ότι θέλω πάντα να έρχονται όλοι οι συντονιστές δικαιωματικά. Γιατί έχουμε πάρει απόφαση που λέει ότι δεν χρειάζονται συντονιστέ. Όταν το απαιτούν οι συνθήκε, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα όμω. Και ένα τελευταίο που έχει να κάνει με θέματα κυκλοφορίας των ε, εγγράφων του τριμερούς διάλογου, διαλόγου. Έχουμε το κλασικό έγγραφο με τις τέσσερις στήλες στο ε, τριμερή διάλογο και προτείνω και μια προφορική τροπολογία. Το βασικό ερώτημα είναι θα έχουμε non-papers και ενημερωμένα έγγραφα τα οποία θα συζητούμε επίσημα στον τριμερή διάλογο. Και πόσο καιρό πριν. Εγώ προτείνω 24 ώρες. Ο κύριος Γκουαλτιέρη προτείνει 48 ώρες. Εντάξει. Το συντομότερο όταν έχουμε πολλούς τριμερεί διαλόγους την ίδια εβδομάδα, δεν ξέρω εάν το 48ωρο μας επιτρέπει να παρακολουθούμε ε, τη δουλειά με αυτό το ρυθμό. Εδώ χρειάζεται λίγο να το διευκρινίσουμε. Έχω στείλει ένα σχέδιο συμβιβαστικό που δεν καλύπτει τα πάντα προφανώς, όλα όσα προτείνονται και μπορούμε και να ψηφίσουμε, ψηφίσουμε επιπλέον όπου ε, οι βουλευτές έχουν κάνει μακροσκελείς τροπολογίες, καλό θα ήταν να τις ψηφίσουμε ξεχωριστά. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας ε, όση ευελιξία χρειάζεται για να ε, η συλλογική βούληση της Επιτροπής. Αυτά ήθελα να πω εγώ εισαγωγικά. Δύο πράγματα που δεν καλύφθηκαν καθόλου στα σημεία που έχω μοιράσει ως πρώτο σχέδιο των συμβιβασμών. Το είναι, είναι το σημείο που σας ανέφερα για την έναρξη ε, διαπραγματεύσεων και αυτό να χρειάζεται ε, πλειοψηφία δύο τρίτων. Για τους λόγους που σας εξήγησα δεν υποστηρίζω αυτή την πρόταση. Ε, προφανώς θα χρειαστεί χωριστή ψηφοφορία γι' αυτό εάν το επιθυμεί, η, επιθυμεί, η πλειοψηφία της Επιτροπής. Και ένα άλλο που δεν ε, συμπεριέλαβα είναι αυτό που περιορίζει το ρόλο του Προέδρου ε, ο σκιώδη εισηγητή. Ο Πρόεδρος πολύ συχνά είναι κατά ανάγκη εισηγητής. Αυτή τη στιγμή για το είσαι ε, 2010. Εκεί στον τριμερή πολιτικό διάλογο όμως έρχεται ο κάθε ναι. πικραμένος από κάθε πολιτική ομάδα. Οπότε τι είμαι εγώ, είμαι πρόεδρος, είμαι εισηγητής, ας είμαστε ε, ρεαλιστές. Εάν καμία πολιτική ομάδα δεν θέλει να αναλάβει ένα ε, θέμα και πέφτει ο κλήρος στον πρόεδρο, θα πρέπει ο πρόεδρος να δρά ανάλογα και υπεύθυνα και σε μια διαπραγματευτική ομάδα συμμετέχουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Οπότε αυτή είναι μια πολύ καλή εγγύηση. Τώρα, για το αν είσαι σκιώδης, εισηγητής και πρόεδρος. Ε, αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. για το τι γίνεται σε σχέση με τις μικρές πολιτικές ομάδες απέναντι στις μεγάλες. Σε ένα ιδανικό κόσμο ο πρόεδρος δεν χρειάζεται να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο βάρος και να είναι σκιώδης. Εγώ είμαι από σχετικά μικρή ομάδα, αλλά ακόμα πιο μικρές ε, μπορεί να διαπιστώσουν ότι θα τους πέσει καμιά φορά και ο κλήρος. Σε ό,τι αφορά τις διοργανικές μάχες που δίνουμε, ο πρόεδρος και προκειμένου εγώ, θα ε, είναι ενδεχομένως καλύτερος και εγώ θα είμαι καλύτερη γιατί το κάνω συχνά αυτό το πράγμα σε σχέση με κάποιους άλλους ε, που δεν ε, ε, ασχολούνται τόσο συχνά. Και όποιος έχει αμφιβολίες για τη διάκριση των ρόλων να το πει και να πει με ποιο τρόπο προχωρήσαμε. Αν είδατε τι έγινε στην οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις στο CRD. Ε, αν έχετε να προτείνετε τίποτα άλλο, με χαρά να ε, το σεβαστώ και να το εφαρμόσω. Αλλά δεν θα κάνουμε τίποτα διαφορετικό από άλλες επιτροπές και είναι σχετικά κοινό στις άλλες επιτροπές, ακόμα και σε μείζωνα πολιτικά ζητήματα, να τα αναλαμβάνει ο εκάστοτε πρόεδρος. Είναι αρκετά συχνό αυτό. Υπάρχουν και άλλες διαδικασίες, άλλες επιτροπές, ας πούμε στην Επιτροπή Βιομηχανίας, όλες οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται από τον πρόεδρο. Δηλαδή και μόνο ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα λόγου. Εμείς είμαστε λίγο πιο χαλαροί στο δικαίωμα λόγου και σε ποιος μπορεί να μιλήσει στο τριμερή διάλογο και καμιά φορά διονύζεται η συνεδρίαση. Αλλιώς δεν θα ήταν και πολύ δημοκρατική. Αυτά. Νομίζω ότι κάλυψα όλα τα θέματα. Έδωσα και την προσωπική μου άποψη. Είναι θέμα επιτροπής και οι σκιώδεις έχουν το λόγο. Ζαν Πολ Γκοζές από το ΕΛΚΑ. Και πάει λέγοντα. Αν θέλει να μιλήσει, βέβαια. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω δει όμως τους συμβιβασμούς ως θέω εγώ, ε, τέλος πάντων. Ορισμένα σχόλια. Πρώτον, μεταξύ των τροπολογιών που έχουμε στο φάκελό μας, στο 5, γενικά είμαι κατά των τροπολογιών του κυρίου Γκουαλτιέρη. Και εγώ ήμουν νομομαθής 25 χρόνια, αλλά δεν πρέπει το δίκαιο να αντικαθιστά την δράση. Γνωρίζετε τη θέση μου, σας την έχω γράψει. Η τροπολογία κλούτ νομίζω είναι πολύ ικανοποιητική. Εδώ που την έχω Τώρα για τον πρόεδρο της Κομισιόν που... Α, η τροπολογία 14 του κυρίου Κλούτου, τη βρίσκω πολύ καλή. Πρέπει να ξέρουμε ότι εδώ στο Κοινοβούλιο λειτουργούμε κάπως περίεργα. Δεν τα λέω για σας. Έχουμε προέδρους επιτροπών που δεν έχουν εκλεγεί κανονικά. Δηλαδή για, το για τους απ' έξω, οι πρόεδροι των επιτροπών φαίνονται σαν κάτι το πολύ σημαντικό που έχουν εκλεγεί από την πλειοψηφία των μελών, από η χρυσορόπηση των πολιτικών ομάδων και στις ομάδες υπάρχει το σύστημα αντών το όπως κάνουμε και εμείς αλλά ο πρόεδρος της Επιτροπής έχει κάποια ιδιαίτερη θέση θεσμικά φαίνεται πιο πολύ αλλά ταυτόχρονα δεν αντιπροσωπεύει αναγκαστικά όταν μιλάει και την πλειοψηφία της Επιτροπής του. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Και υποφελούνται από αυτό οι πρόεδροι, αλλά τέλος πάντων. Δεν θα κάνουμε και επανάσταση εδώ. Τέλος πάντων, χρειάζεται να είναι ουδέτερος στον τριμερή διάλογο πρόεδρος της Επιτροπής. Το είπατε και εσείς, υπάρχει διαφορά μεγάλων και μικρών ομάδων, γιατί χρειάζεται να κατανεμηθούν οι εκθέσεις και μεταξύ μεγάλων και μικρών ομάδων. Είπατε για την Επιτροπή Βιομηχανίας, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Υπάρχουν θέματα ιδιαίτερα σημαντικά. Δεν λέω τα δικά σας που τα αναλάβατε γιατί δεν ήθελε κανείς να τα αναλάβει. αυτά που σας έγραψα ισχύουν. Πρέπει να είναι σαφή τα πράγματα, δεν αμφισβητώ την προσωπική εντιμότητα προέδρων, απλώς είναι θέμα διαφάνειας. Όλοι σήμερα μιλάνε γι' αυτό, οι Αγγλοσάξονες μιλούν για διαμάχη συμφερόντων, αντιμαχόμενα συμφέροντα. Εγώ δεν, δεν μου αρέσουν τόσο πολύ αυτές οι έννοιες, αλλά αφού το βάζουμε παντού πρέπει να το κάνουμε τίμια. Στη Γαλλία είχε τεθεί το πρόβλημα αν ήταν πρόεδρος του Κοινοβουλίου ή πρώην σύντροφος του Προέδρου. Τέλος πάντων δεν τίθεται αυτό γιατί δεν εξελέγει, αλλά το βρίσκω όλα αυτά σοκαριστικά. Αυτή είναι όμως η προσωπική μου θέση, την ξέρετε, την είπα ότι την έχω γράψει και σταματώ εδώ. Δεν έχω άλλον από την σοσιαλιστάς, ο Σβέν. Α, ναι. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ για τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Μετά την τελευταία συζήτησή μας για το θέμα, είπαμε να μην πάμε στο ποια πλειοψηφία χρειάζεται για να επανυποβληθούν ορισμένες ή για να προχωρήσουμε σε άμεσο τριμερή διάλογο. Η διαφορά μεταξύ πλειοψηφίας δύο τρίτων και απλής είναι μάλλον φιλοσοφική από άποψη νομιμότητα ίσω τα δύο τρίτα να είναι καλύτερα από μια απλή πλειοψηφία αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το κύριο θέμα. Οι συμβιβαστικέ σα είναι ισορροπημένε και προ την κατανομή, διανομή των υλικών που, του υλικού που αναφέρεται και στην τροπολογία 14 του Γιούργεν που ανέφερε και ο Ζαν Πολ πρέπει να πω ότι αν δίνουμε όλα τα υλικά του τριμερούς διαλόγου σε όλες τις ομάδες τότε θα έμοιαζε με το να τα βάλουμε στο ίντερνετ η διανομή του υλικού μεταξύ των ομάδων, των διαπραγματευτικών ομάδων, των μελών των διαπραγματευτικών ομάδων. Ε, ναι, ναι. Ε, εδώ λέει μεταφράζω από τα γερμανικά του Γιούργεν, άντε ας τα πω γερμανικά, ας τα πω γερμανικά κατευθείαν. Η ε, τροπολογία 14 που μόλις επένεσες. Γράφει όλα τα γραπτά και επίσημα έγγραφα που ελέγχονται διανέμονται σε ολόκληρη διαπραγματευτική ομάδα και ενδεχομένως αυτό μπορεί να γίνει μέσω των πολιτικών ομάδων. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι καταρχήν θα πρέπει να τα παίρνουν όλοι τα έγγραφα. Σε ποια παράγραφο, στην 4. 4. Α, εγώ στα γαλλικά κατάλαβα ότι αναφέρεσαι στη 14 του Γιούργεν και την επένεσες. Όχι τη 14, την 4. Μα εγώ εδώ λέει τροπολογία 14, Γιούργεν Κλούτε. Παράγραφο 4 της τροπολογίας αυτή. Εν περιπτώσει, αφού έχω το λόγο, θέλω να πω, για να τελειώσω, ότι αυτό το πρόβλημα, ποιος παίρνει ποια έγγραφα από τους τριμερείς ε, διαλόγους και τις συζητήσεις των σκιωδών είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε ξανά. Γιατί αυτά τα χαρτιά κυκλοφορούν και τα σπέρνουν διάφοροι δεξιά και αριστερά. Παράδειγμα, από ένα κράτος μέλος πήρα σχέδιο για συμβιβασμούς για ένα άλλο κράτος πριν τα λάβω επίσημα ως και ηγητής. Ε, αυτά είναι μυστήρια πράγματα. Λοιπόν, και ποιος μοιράζει τι χαρτιά σε ποιον είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε καμία φορά οι συντονιστές. Εν πάση περιπτώσει, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ευχαριστώ για τις τροπολογίες, όλα καλά και όλα τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε εν ευθέτω χρόνο για την έκθεση που θα κάνετε και τις εκθέσεις που παίρνετε αναγκαστικά γιατί δεν τις θέλει κανένας. Ξέρετε ποια είναι η γραμμή του Κοινοβουλίου. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και στην επόμενη φορά θα είμαστε παρόντες στη συνεδρίαση των σκιωδών και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, just to clarify... Ευχαριστώ. Αλλά για να καταλάβουμε, έχει 7 παραγράφους η τροπολογία 14 του Γιούργεν, ενώ ο Ζαν Πολ μιλούσε για την παράγραφο 2 της τροπολογίας αυτής, ενώ εσύ για την παράγραφο 4. Όχι, υπήρχαν δύο θέματα. Εγώ προηγουμένως, αναφερόμενος στην 14, μιλούσα για την παράγραφο 2 της. Αλλά ο φίλος μας ο Σβέν, που μίλησε για τη διανομή των εγγράφων, για όλους τους βουλευτές, εγώ βλέπω ότι στην παράγραφο 4 γίνεται λόγος μόνο για τη διαπραγματευτική ομάδα, για τα μέλη της, όχι για όλους τους βουλευτές. Όχι για όλους. Α, ναι. Και μετά λέει να δίνεται και στις ομάδες όπως χρειάζεται. Ναι, πρέπει να συζητήσουμε πώς μοιράζονται και πόσο τα έγγραφα. Ο Γιούργεν να μας τα πει. Να σας τα πω. Ευχαριστώ. Αρχικά μια σύντομη παρατήρηση σε σχέση με αυτά που είπε ο Σφέν. Ότι πήρε από μια χώρα μέλος συμβαστικές προτάσεις. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όταν είχα κάνει εγώ έκθεση για την κοινωνική ένταξη και την οικονομική ένταξη, μας παίρναν τηλέφωνο διάφορα λόμπι και τους βοηθούς μας ε, για να μας πούν τι να κάνουμε και τι να προτείνουμε. Και ότι οι συμβιβασμοί ως σχέδια να στέλνονται ε, προηγουμένως στα λόμπι. Προφανώς εμείς δεν αντιδράσαμε, το συζήτησα με τους ε, συναδέλφους και τους υπαλλήλου και τους έδωσα σαφείς εντολές. Δεν πρόκειται να βγει τίποτα έξω που να μην έχει τεθεί υπόψη της διαπραγματευτικής ομάδας ή των μελών της Επιτροπής. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι, να το συζητήσουμε και αυτό καμιά φορά. Ε, γιατί θεωρώ ότι οι βουλευτές είναι εδώ επειδή είναι εκλεγμένοι και έχουν ε, το δικαίωμα να βλέπουν πρώτοι τους συμβασμούς και τα αντικείμενα της διαπραγμάτευσης. Αλλά για να έρθω σε αυτή την παράγραφο 4 ή 5, ε, ε, αυτό έχει να κάνει με την Επιτροπή μας. Ότι εμεί θέλουμε στην Επιτροπή να διαπραγματευόμαστε και να επιβεβαιώνουμε ότι αυτά που έκανε η διαπραγματευτική ομάδα ε, ισχύουν ε, και τι κάνει, θα πρέπει να ξέρει η Επιτροπή τι διαπραγματεύεται η ομάδα και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Βεβαίως να προσέξουμε να μην κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, αλλά κάπως πρέπει να ενημερώνεται και το σύνολο της Επιτροπής, όχι μόνο η διαπραγματευτική ομάδα, εφόσον καλείται να, να αποφασίσει η ε, Επιτροπή. Πώς θα το εξασφαλίσουμε αυτό, πώς θα το κλειδώσουμε να μην διαραίουν τα έγγραφα προς τα έξω, θα τα δούμε. Μπορεί ο καθένα να λαμβάνει ή διευθύνει ο βουλευτή ότι ορισμένα πράγματα δεν θα τα πει παρά έξω. Υπάρχει και το εμπιστευτικό και το απόρριτο και τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας ε, βέβαια δεν επιτρέπουν πάντα την απόλυτη εχεμήθεια. Λοιπόν, ε, ε, δύο-τρεις μεμονωμένες παρατηρήσεις γιατί τελείωσε αυτό για τους συμβιβασμούς που πρότεινε η Σάρων. Ε, πρέπει να πω ότι συμφωνώ σε γενικές γραμμές πάντως. Αυτή η παράγραφος στην οποία αναφέρθηκε ο Ζαμπόρ, ε, να τα πω πιο ξεκάθαρα στην ε, τροπολογία μου, μα είναι μια ουδέτερη θέση. Ο πρόεδρος προεδρεύει. Η Σάρων το κάνει πολύ ωραία, είναι και το βρετανικό στυλ, αλλά δεν ήθιστε παντού και καλό είναι να γράφουμε κανόνες. Οι κανόνες ισχύουν για τις περιπτώσεις συγκρουσιακές, όχι τις ε, κανονικές συνθήκες ε, και θα πρέπει να ξέρουμε τι είναι αποδεκτό, τι είναι παραδεκτό και τι απαράδεκτο και θα παρακαλούσα να ε, το εξηγήσουμε με τρόπο πιο οξύ, ότι η θέση του Προέδρου είναι δέτερη, απλώς προεδρεύει. Και ειδικά σε περίπτωση συγκρούσεων. Αυτό το 24ωρο ή 48ωρο, καλύτερα 24 ώρες. Γιατί θα προτιμούσα. Γιατί είναι τόσο σφιχτές οι διαπραγματεύσεις και τόσο κοντά η μία με την άλλη που δεν προλαβαίνουμε με 48 ώρες. 24 εντάξει. Το παραπάνω δεν μου φαίνεται φυκτό και εφαρμόσιμο. Και αυτό το θέμα, το 2 τρίτα το μελών, συμφωνώ με τη Σάρων απλή πλειοψηφία για να μπορούμε και να λειτουργούμε. Τι να τα κάνουμε τα δύο τρίτα στην Επιτροπή. Αρκεί η απλή πλειοψηφία. Αυτά. Α, ένα τελευταίο που ξέχασα. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε οπωσδήποτε, αλλά είπε κάτι η Σάρον για το πώς εκπροσωπείται ο Πρόεδρος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για το πώς θα γίνει αυτό. Είναι δύσκολο και με τους αντιπροέδρους πάντα. Να τα αφήσουμε τελείως αρρύθμιση αυτό, ανοιχτό στη διακριτική ευχαίρεια. Κάποιος από τη διαπραγματευτική ομάδα να εκπροσωπεί τον πρόεδρο. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο να πούμε ξαφνικά ότι μπορεί οποιοδήποτε χωρίς καμία ρύθμιση και κανένα κανόνα. Αυτά. Ευχαριστώ. Um, thank you very much. I've got uh, Thomas Mann and Udo Bullman, as we haven't had anybody as... Δεν ήταν εδώ ο Γκαλτιέρη. Ούντο πήγαινε, πάρε το λόγο πρώτο. Δεν είχαμε πρόσωπο το XND. Ήδη ξεπεράσαμε το χρονικό μα περιθώριο. Ελπίζω να μείνουν και άλλοι διερμηνεί, λέει ο πρόεδρο. Μπα. Ευχαριστώ Σάρων. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος για αυτό το θέμα στην ομάδα μας. Αλλά μια που είμαι παρόν να μιλήσω εξ ονόματος του η εισηγητού, γενικά είναι εύκολο να γίνει αυτό, συμφωνεί ο Σκιώδης με τους συμβιβασμού που προτείνονται, τον αντιπροσωπεύουν και είμαι βέβαιος ότι θα χαρεί ιδιαίτερα που τον επένεσε ο Γκοζές και θα το διαβιβάσω αρμοδίω. Κατά τα άλλα όλα καλά. Ευχαριστώ, Σάρον. Επειδή δεν έχουμε και τόσο πολύ χρόνο, ε, τρία σύντομα. Πρώτον, για την τροπολογία 14. Έχω πρόβλημα με την πέμπτη παράγραφο για τα έγγραφα και τα άλλα τα ανεπίσημα έγγραφα να τα παίρνουν τόσοι πολλοί. Και εγώ είμαι υπέρ της διαφάνειας όπως όλοι. Αλλά όταν έχουμε δώσει σε κάποιους ηγετικέ ε, αρμοδιότητες να ηγούνται κιόλας. Και η ηγεσία συμβαδίζει με την εμπιστοσύνη. Λοιπόν, έχετε αυτό το έργο επομιστεί και ελπίζουμε να ανταποκριθείτε και να είστε στο ύψος των περιστάσεων και ε, θα κριθείτε εκ του αποτελέσματος. Άλλο, για το 24ωρο συμφωνώ, 48 μου φαίνεται πολύ. Ε, Και μετά ε, κάτι άλλο επίση σημαντικό για μένα. Στο θέμα το ποιο εκπροσωπεί ποιο. Μα του αντιπροέδρους γιατί τους έχουμε. Δεν μας αρκούν. Και όχι να έχουμε περιτροπή προεδρία. Όχι. Είναι πολύ ε, σημαντικές αυτές οι ιστορίες και θέλουμε και αποτελέσματα. Και για το 13 του κυρίου Λάγκερ να το συζητήσουμε μαζί του. Τώρα τα δύο τρίτα είναι ευρύτερη πλειοψηφία. Να πούμε πριν ληφθούν αποφάσεις χρειάζεται ευρία πλειοψηφία. Άρα τα δύο τρίτα παρά είναι. Ε, ίσως να το σκεφτούμε και αυτό. Αυτά γενικά δεν διαφωνούμε με τον Λάγκεν. Και δεν είμαστε και μακριά. Λοιπόν, χάνουμε τη διερμηνία, λέει η πρόεδρος, διότι σχολάνε οι διερμηνείς. Σβέν, πολύ σύντομα. Ε, θα προτιμούσα έτσι και αλλιώς αγγλικά, ακόμα και σε κακά αγγλικά, χωρίς διερμηνία.